Καλημέρα σας. Λέω ο πρόεδρο, να σας χαιρετώ αυτή τη φορά επισήμω. Σύμφωνα με την ημερησία διάταξη αρχίζουμε και έχω μία ανακοίνωση να κάνω. Κατόπιν της ε, παρετήσεως του κυρίου Γιάκοπ Φων Βάστσεκερ το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει το ότι χειρεύει η έδρα του από τις 7 πρώτου του 2019 σύμφωνα με τον κανονισμό και έχουμε ενημερώσει τι αρμόδιε εθνικέ αρχέ. Και τώρα, προχωρούμε στο πρώτο θέμα τη Μέση και πρόκειται για τη δήλωση τη Επιτροπή για την κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα Βοσνία Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δίνουμε το λόγο στον Επίτροπο Αντριουκάτης για να μας παρουσιάσει τις ε, απόψεις της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Ναι, επιτρέψατε μου και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τις οικογένειες των ε, θυμάτων ε, της ε, τρομοκρατικής επίθεσης εδώ στο Στρασβούργο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα, να σας δώσω μία γενική εικόνα. Η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη δεν είχαν επηρεαστεί από την μεταναστευτική κρίση του 2015 όμως μεταξύ Ιανουαρίου και 30 Νοεμβρίου 2018 γύρω στους 33.000 μετανάστες μπήκαν στη χώρα. Μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2017 αλλά διαχειρίσιμη. 92% εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ζητήσουν άσυλο αλλά μόνο 5 το έκαναν οι περισσότεροι ήθελαν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως ε, θεωρούν την Βοσνία Ζεγοβίνη ως μια χώρα διέλευσης. Από 4 Δεκεμβρίου, μα, στις 4 Δεκεμβρίου υπήρχαν 1.139 πρόσφυγες και μετανάστες που έλαβαν βοήθεια. 3.000 ε, δε στο καντόνι της ε, Ουνασάνα στα βόρειο-δυτικά της χώρας ε, στα σύνορα με την Κροατία. Άλλοι χίλιοι δεν έχουν ζητήσει ακόμα βοήθεια και υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην περιοχή. Η Κομισιόν αντέδρασε αμέσως στις ανάγκες της χώρας από τον Ιούνιο του 2018 η Κομισιόν διέθεσε ένα σημαντικό ποσό κονδυλίων για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες ε, των ανθρώπων αυτών. Δεύτερον, ε, για να υπάρξει επαρκή στέγαση και βασικές υπηρεσίες. Τρίτον, να αυξηθούν οι δυνατότητες ταυτοποίησης και τέταρτον να στηριχθεί η συνοριακή αστυνομία της ε, χώρας. Αυτό περιλαμβάνει και 2 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια και 7,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω ενός ειδικού μέσου του, της προενταξιακής βοήθειας. Αυτά τα εφαρμόζει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την υπατιαρμοστία του ΟΗΕ και τη UNICEF. Αυτά τα κονδύλια προστίθενται σε αυτά στα οποία έχουν ήδη δοθεί στη Βοσνία Ζεγοβίνη μέσω του κυρίου προενταξιακού μέσου για την διαχείριση των συνόρων, τη μετανάστευση και το ασύλο. Χάρη στην βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άτομα που βρίσκονται στο καντόνι της να πηγαίνουν σε οργανωμένα κέντρα υποδοχής. Ο στόχος είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής. 4.000 άτομα αυτή τη στιγμή να έχουν στέγη και κανείς δεν είναι στο κρύο. 61 παιδιά θα ξεκινήσουν ε, το σχολείο προσεχώς και η περαιτέρω βοήθεια θα είναι διαθέσιμη για να καλυφθούν οι ανάγκες από τον Απρίλιο 2019 και μετά. Αυτό θα βασιστεί στην αξιολόγηση των αρχών. Όπως γνωρίζετε, η διαπραγματεύσει με την Βοσνία Ζεγοβίνη για μια συμφωνία κάθε στότος για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένουμε την υπογραφή της συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν. Η συμφωνία καθεστώτος θα μας βοηθήσει να βοηθήσουμε την ε, συνοριακή αστυνομία. Η κύρια ευθύνη βεβαίως παραμένει στη χέρια των δύο χωρών. Η Βοσνία ανέπτυξε τις προηγούμενες εβδομάδες άλλους 180 αστυνομικούς. Οι σχέσεις ε, μεταξύ της συνοριακής αστυνομία και των μεταναστών φαίνεται ότι συνολικά είναι θετικές όπως ε, μαθαίνουν ε, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όπως είπα, η χώρα θεωρείται μια χώρα διέλευσης. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη και για τον τοπικό πληθυσμό που αναφέρει εντάσεις και φόβο για περιστατικά ασφαλείας. Τους τελευταίους μήνες είχαμε αναφορές σοβαρών κατηγοριών για κακομεταχείριση των ε, ανθρώπων αυτών από την αστυνομία. Η Κομισιόν παρακολουθεί τις εξελίξεις ε, και τις καταγγελίες αυτές. Να τονίσω πως η συμφωνία επανεισδοχής ε, θα πρέπει να ισχύσει για όσους διασχίζουν παράνομα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αυτό να επηρεάζει το δικαίωμα υποβολής ασύλου και γενικότερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο. Και βεβαίω ε, η αρχή της μη επαναπρόθεσης. Ε, η Λόρα Βίντεβιτς, η συνήγορος του Κροάτι πολίτη παρουσίασε μία έκθεση στην Βουλή της Κροατίας και εξέφρασε τις ανησυχίες της για το ότι η αστυνομία παραβίαζε τα δικαιώματα των μεταναστών για την διεθνή προστασία και δεν τις επέτρεπαν να βρει πληροφορίες. Παρακολουθούμε την κατάσταση στενά. Συμφωνούμε όλοι ότι τα σύνορα μεταξύ Βοσνίας και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξωτερικά σύνορα και η Κροατία είναι υπεύθυνη για την διαχείρισή τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αναλογικά και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, να τονίσω πως είμαστε πεπισμένοι πως οι αρχές της χώρας θα λάβουν υπόψη σοβαρά τι καταγγελίε και θα διεξάγουν γρήγορε ε, και ενδελεχείς έρευνες. Δεύτερον, οι συνοριοφύλακες ε, αναμένουμε να διεξάγουν τα καθήκοντά τους σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση τώρα. Η συνάδελφος Σούτσα. Ξέρετε ότι τα κροατικά σύνορα είναι χίλια περίπου χιλιόμετρα, κυρίως με την Βοσνία Ευζεγοβίνη, είναι τα πιο μακρά σύνορα εξωτερικά σε υπηρετική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα λοιπόν η Κροατία προσπαθεί να σεβαστεί όλους τους διεθνείς κανονισμούς και τις διεθνείς συμβάσεις. Είπατε ότι ο αριθμός των μεταναστών στη Βοσνία δεν είναι ο ίδιος με το 2015. Τα επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι έχει υπάρξει αύξηση 57%. 6.500 περισσότεροι σε σχέση με το 2015. Λόγω των συμφωνιών που έχουν υπάρξει και με τις τρίτες χώρες, οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την Τουρκία. Αλλά επειδή το σύστημα θεωρήσεων δεν είναι εναρμονισμένο, υπάρχουν και από άλλες χώρες. Οι χώρες της Δυτικής Βαλκανικής λοιπόν αντιμετωπίζουν μια τεράστια πίεση από μεταναστευτικές ροές. Οι Κροάτες ε, έχουν περισσότερους ε, φύλακες, σύνοριοφύλακες από όλες τις άλλες βαλκανικές χώρες και πρέπει να αντιμετωπιστεί όποιο πρόβλημα έχει υπάρξει και θα πρέπει επίσης και οι διαδικασίες επαναπατρισμού όπου εφαρμόζονται να εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο. Υπάρχει βοήθεια και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δύο εκατομμύρια ε, ευρώ δόθηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια και έξι εκατομμύρια για ενίσχυση του συστήματος επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φαγιόν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 23 ε, εγγεγραμμένες αφήξεις στη Βοσνία Ευζεγοβίνης από την αρχή του χρόνου. 5.500 ε, είναι στη Βέλικα Κλάντουσα και στο Μπίχατς και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί να δοθούν απαντήσεις είναι στην πορεία την οποία ακολουθούν οι μετανάστες αυτοί για την Δυτική Ευρώπη. Ξέρουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Ε, κάποια πολιτικά κόμματα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα το μεταναστευτικό για να προκαλέσουν το μίσος της κοινωνίας εις βάρος τους. Κυκλοφορούν φήμες ότι οι μετανάστες συστηματικά κάνουν απαγωγές νέων παιδιών, ότι βιάζουν νέα κορίτσια κτλ. Η επιπλέον οικονομική βοήθεια λοιπόν είναι απαραίτητη για τη Βοσνία. Αναφερθήκατε στον ρόλο των συνοριοφυλάκων. Και η Κροατία και η Βοσνία Ευζεγοβίνη θα πρέπει να λύσουν το πρόβλημα με τρόπο ο οποίος να σέβεται τις αρχές της ανθρωπιστικές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φαγιώνη, κυρία Τόμασίτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών στην Βοσνία Ευζεγοβίνη ε, προκαλεί πλέον προβλήματα και ανησυχίες γιατί η χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνη της. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ανθρωπιστικές διαστάσεις και ε, προβλήματα σε επίπεδο δημόσιας υγιεινής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μένουν είναι απαράδεκτες και γι' αυτό προσπαθούν να περάσουν στην Κροατία η οποία έχει μακρά σύνορα και διαπερατά σύνορα με την Βοσνία Ευζεγοβίνη. Η Κροατία προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά έχει ανάγκη και αυτή από οικονομική βοήθεια. Η Κροατία θα πρέπει να ενταχθεί πλέον στον χώρο Σέγγεν αυτό θα ήταν ένα σωστό μήνυμα. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για δύο λόγους ζήτησα να ενταχθεί στη μέση διάταξη προς συζήτηση η κατάσταση στα σύνορα Βοσνίας και Κροατίας. Πρώτα πρώτα, ο πρώτος λόγος είναι ανθρωπιστικός, δηλαδή η κατάσταση των προσφύγων. Έχουν παγώσει στο κρύο. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Μεγάλες δυσκολίες. Αλλά υπάρχουν και δυσκολίες όσον αφορά τις σχέσεις τους με τον ντόπιο πληθυσμό. Οι ντόπιοι φοβούνται και οπότε θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορεί αυτό το πρόβλημα να το αφήνουμε κατά μέρος. Επίσης, η Κροατία από τη μια μεριά κατηγορείται γιατί λένε ότι δεν ε, τους φέρονται δίκαια από την άλλη μεριά. Όμως έχει την υποχρέωση η χώρα να φροεί τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα προστατεύει. Οπότε σας ευχαριστώ που συζητούμε το πρόβλημα. Αυτό θα βοηθήσει στην κατάσταση εκεί. Αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά τις εξελίξεις. Οι θεσμοί στη χώρα δεν λειτουργούν εύρεθμα και τα προβλήματα έχουν επιπτώσεις στο σύνολο της Ένωσης. Οπότε παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει την χρηματοδότηση. Και γι' αυτός ε, απευθύνω έκκληση όλοι οι μετανάστες εκεί να έχουν μεταχείριση ανθρώπινη, αλλά να παρακολουθούμε από κοντά τι γίνεται και εκεί. Επίσης, τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι οι εξελίξεις οδήγησαν στο να μειωθεί κάπως μετανάστευση, αλλά πάντως δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας. Επομένως, από το 2016 αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι με κάθε θυσία να κλείσουν τα Βαλκάνια και τους διαδρόμους μετανάστευσης. οπότε έχουμε χιλιάδες που μπλοκαρίστηκαν στην Βοσνία και η κατάσταση εκεί είναι απάνθρωπη να πρέπει να δούμε τι κάνουν οι κροατικές αρχές εκεί στη Μεθόριο μόνο από Ιανουάριο ή από Αύγουστο έχουμε πάνω από 2.500 επαναπατρισμούς και επίσης έχουν καταγγελθεί βίες ενέργειες από πλευράς των δικτικών αργών προς τους και εις βάρος των ε, μεταναστών. Πολλοί ε, αναφέρονται ότι έχουν πεθάνει από όλα αυτά και τελευταία πέθανε από τέτοιες ε, ενέργειες ένα παιδάκι 6 ετών, ένα κοριτσάκι και είδαμε ότι ε, κατηγορούνται, διώκονται, καταστέλλονται από τις αστυνομικές αρχές και τελικά τι κάνει η Κροατία. Η Κροατία ε, είναι σε εμπλοκή ε, και ακολουθεί ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεταναστή. Δεν γίνεται τίποτα διαφορετικό από ό,τι στα υπόλοιπα σύνορα της Ένωσης. Στη Θέουτα και στην Μιλίγια και εκεί έχουμε αυτούς τους ε, φράχτες, έχουμε βία, έχουμε βίες επίσης βίους επανεπατρισμούς και στην Ουγγαρία του Όρμπαν καταπαντώνται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης έχουμε αυτό το τεράστιο σύνορο, την ε, Μεσόγειο. Και τι γίνεται εκεί πέρα, πνίγεται ο κόσμος. Όλα αυτά αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό το πολιτικό όραμα, το πολιτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταπατά το ίδιο το κοινοτικό δίκαιο. Κροατία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιταλία, δεν, δεν πάσχει η κατάσταση μόνο εκεί. Το κλείσιμο των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ότι η πολιτική είναι κανένας να μην πατήσει στην ε, Ευρώπη, όλοι να, ε, να διωχτούν. Ε, αυτό, αυτό είναι η βάση του και η πηγή του κακού. Άρα όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι, όλοι είμαστε συνεργοί σε αυτό το έγκλημα και κυρίως και εμείς. Βαλέρο, συγγνώμη. Έκανε λάθο ο πρόεδρος, η Βαλέρο μόλις μίλησε. Έχετε μια επερώτηση, μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε κύριε Βαλέρο. Μάλιστα. Δύο, δύο μπλε κάρτες για σα κύριε Βαλέρο. Κύριε Βαλέρο, να σας ε, απαντήσω. Άδικα κα, καταδικάζεται και άδεια κατηγορείται την ε, Κροατία. Πήγαμε στο Μαρακές, προσπαθήσαμε να ρυθμιστούν τα της μετανάστευσης. Δεν θέλουμε να είναι διχασμένη η Ευρώπη. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους φουκαράδες να προστατευθούν, να βρίσκονται σε ασφάλεια. Όχι, μην κατηγορείτε την Κροατία, γιατί αυτό είναι νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Ε, αυτό ήταν ε, σχόλιο, δεν ήταν ερώτηση. Θέλετε να ακούσετε τη δεύτερη ερώτηση και να, ακούσετε, και να απαντήσετε και στις δύο, κύριε Βαλέρο, ή θέλετε να απαντήσετε μία-μία. Ναι, εντάξει, τώρα θέλετε. Σας ακούμε. Δεν κατηγορώ την Κροατία. Κατηγορώ όλες τις κυβερνήσεις της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταναστευτική πολιτική που είναι απάνθρωποι, καμία σχέση με την ελεγγύη. Δεν φέρει ευθύνη μόνο η Κροατία, η Ιταλία, η Κροατία. Όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Η Κομισιόν, το Συμβούλιο. Και σας το είπα και η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών που δίνουν πράσινο φως με την ψήφο τους σε τέτοιες πολιτικές. Κυρία Σουίκα, Σουίτσα τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακολουθούσα τις ομιλίες κύριε Γκουσμάν ε, τους τελευταίους μήνες ε, χρησιμοποιείτε το θέμα αυτό για την προώθησή σας και τη, τη μοίρα, την άθλια των μεταναστών αυτών για να κάνετε διαφήμιση. Όταν μιλάτε για την Κροατία, ε, εμείς εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα που πρότεινε η Αυστριακή Προεδρία και οι Κροάτες αστυνομικοί σέβονται όλους του διεθνείς ε, κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, όχι, μην μου λέτε εμένα ότι πάνε κερδίσω ψήφους και ότι είμαι λαϊκίστρια όταν ε, στην ε, συζήτηση για το μεταναστευτικό κάποιος το συνδέει με την τρομοκρατία. Αυτό είναι χειρότερα από λαϊκισμό. Αυτό είναι ακροδεξιά να τα ανακατεύετε όλα στην ίδια συζήτηση, την τρομοκρατία και το μεταναστευτικό. Ε, αυτό είναι ξενόφοβο και ρατσιστικό. Βαλέρο, Βαλέρο, δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ με την ε, προηγούμενη ομιλήτρια. Το θέμα είναι γενικώ η ευρωπαϊκή πολιτική και τι βλέπω εγώ εδώ. Μιλάμε για αριθμούς αντί για ανθρώπους. Δηλαδή σαν να μην είναι άνθρωποι. Μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται εδώ. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, και εμείς ε, μιλάμε σαν να ήταν αριθμοί. Στατιστικά στοιχεία. Και αυτό είναι το πρόβλημα νομίζω για όλους μας. Είμαστε στη σημερινή κατάσταση επειδή οι χώρες ε, δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους στο μέτωπο της αλληλεγγύης και της υποδοχής όσων έρχονται. Κάποιοι αρνούνται ξεκάθαρα να δεχτούν. Η χώρα μου η έχει πάρει πάρα πολλούς. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά μαζί. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική και να μην βλέπουμε τους ανθρώπους σαν αριθμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, για να έρθουμε και στο σημερινό μας το θέμα, τα σύνορα με την Βοσνία. Είναι καλό αυτό το οποίο είπε ο Επίτροπος, ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί προφανώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σέβονται τους κανόνες μας. Δηλαδή αν κάποιος καταφέρει να φτάσει στην Κροατία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο. Δεν μπορεί να το στέλνουμε πίσω σε μια άλλη χώρα, έτσι απλά. Ανεξαρτητός του αν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες επιστροφής με τη χώρα έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να τον ταπεινώνουμε, να του αφαιρούμε τα προσωπικά του είδη κλπ. Πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και τον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Σέθεριτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή πως ε, θα πρέπει βεβαίως ε, όλοι να ευχόμαστε ότι καλύτερο για όλους τους ανθρώπους, ε, ειδικά όσους δυσκολεύονται χριστουγεννιάτικα να κοιμηθούν σε ένα ζεστό κρεβάτι. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο ένα θέμα εμπορίου, αλλά βλέπουμε μια πραγματική κατάσταση που υπάρχει με τη μετανάστευση και τα ζητήματα συνόρων. Και μιλάμε για την ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, τα λεφτά που ξοδεύονται. Δηλαδή, θεωρώ βαθιά μέσα μου ότι εάν δούμε την μετανάστευση σε χώρες, σε κυρίαρχα κράτη, θα ήταν καλύτερο να έχουν τον έλεγχο των συνόρων τους. Και αν χρειάζονται βοήθεια, υπάρχει προϋπολογισμός ξένης βοήθειας. Έχουμε ε, τεράστιο τέτοιο προϋπολογισμό στο Ενωμένο Βασίλειο. Και διπλάσιο, δηλαδή ε, από όσο δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογικά. Οπωσδήποτε λοιπόν είναι καλύτερο το κάθε κράτος να ελέγχει τα σύνορά του και αν χρειάζεται βοήθεια να το δούμε μέσω της βοήθειας πάλι μέσω άλλων κρατών. Μποργέτσιο για ένα λεπτό. Ο Αντώνιο Μεγκαλίτσι, 28 ετών, παλεύει να μείνει στη ζωή μετά από την απόπειρα την προχθεσινή θύμα της Ισλαμικής τρομοκρατίας του Στρασβούργο. Αυτό έχει άμεση σχέση με το θέμα το οποίο συζητάμε, γιατί οι εξελίξεις με τους μετανάστες κρύβουν μερικές φορές μαχητές του Ισλαμικού κράτους οι οποίοι έχασαν τη μάχη στη Συρία και προσπαθούν να βρουν ε, διεξόδους και μέσω της Βοσνίας Ευζεγοβίνας. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, τα πρόσωπα αυτά να εισέλθουν στην Ευρώπη ε, και να προσπαθήσουν να επηρεάσουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τους Ευρωπαίους νέους μουσουλμάνες. απαιτείται να υπάρξει μια πραγματική προσπάθεια από ριζοσπαστικοποίησης, να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι τους βοηθούν να ριζοσπαστικοποιηθούν και να σταματήσουν οι απόπειρες ε, της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε να κάνουμε με την Ισλαμική τρομοκρατία. Ο κύριος Διάστε Μέρα, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των αφήξεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη κατά τη διάρκεια του ενεστώτος έτους έχει αυξηθεί ιδιαίτερα και σε σχέση με τις ε, πολύ λιγότερες αφήξεις το 2017 προσπαθούν μέσα από τη Βοσνία να έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνώντας και από την Κροανία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι ήδη από το Νοέμβριο του 18 που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Στερούνται ε, βασικής βοήθειας, τροφίμων, ιατρικής βοήθειας οι δυνατότητες της χώρας έχουν πλέον ξεπεραστεί και ε, τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για βοήθεια μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη διευκολύνει αλλά λίγο τα πράγματα και διευκολύνει λίγο γενικά τη βελτίωση των συνθήκων ε, στα δίκτυα διακίνησης των μεταναστών. Ε, πρόκειται για ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και τη Συρία οι αριθμοί αυξάνονται ε, και δυστυχώς και τα εγκληματικά δίκτυα ε, προσπαθούν να εντατικοποιήσουν τις δραστηριότητες τους στα πλαίσια της ε, εμπορίας ουσιαστικά ανθρώπινων ψυχών. Απαιτείται λοιπόν αύξηση της συνεργασίας με τη Βοσνία Ευζεγοβίνη, η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Σύμβαση 67, ε, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Προσφύγων ε, μας υποχρεώνει να βελτιώσουμε τις ανθρωπιστικές συνθήκες υποδοχής των ανθρώπων αυτών. Και επίσης ε, χειροκροτώ και την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών με την απόφαση που ελήφθη πριν λίγες μέρες στο Μαρακές. Βάιντεν Χόλτσερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ πέρα θέλουμε να ρίξουμε λίγο φως ε, στην κατάσταση στη Βοσνία που είναι ανησυχητική. Έχουμε από το συμβολικό κλείσιμο της διόδου των Βαλκανίων χιλιάδες ανθρώπους ε, στην περιοχή έχουν ξεχαστεί από την κοινή γνώμη και ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Και έχουμε πάντα απεγνωσμένες προσπάθειες για να ξεφύγουν από αυτήν την κατάσταση, κάτι το οποίο βεβαίως ευνοεί τις εγκληματικές συμμορίες. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα περιστατικά των θάνατων ω κοριτσιού τη κυρία ε, Δεσμηνίδο Ροζίνη. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί το τι συνέβη εκεί πέρα, ποιο είναι ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται, πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα θα λυθούν εάν δεν τα κοιτάμε. Ε, αυτά ήδη το 2015 οδήγησαν σε τρομακτικές συνέπειες. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να μάθει από τα τότε λάθη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κέλμελ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή δείχνει πως κάποιοι ομιλητές προσπαθούν με την ανθρωπιστική πτυχή να υπονομεύσουν την κυριαρχία των κρατών μελών. Κυριαρχία σημαίνει διασφάλιση των συνόρων. Δεν είναι τίποτα το καινούριο το ότι μεγάλο κομμάτι των μεταναστών αυτών είναι οι λεγόμενοι οικονομικοί μετανάστες. Δηλαδή δεν υφίστανται δίωξη, αναζητούν καλύτερη ζωή. Εντάξει, θεμητό. Αλλά οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να δεχτούν απεριόριστο και ανεξέλεγκτο αριθμό ανθρώπων. Βλέπουμε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό. Και πρέπει να σας πω κυρία Γκουσμάν της Γκουε. Εδώ πέρα με τρόπο εσχρό προσπαθήσατε να παραστήσετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ε, άγιοι. Δηλαδή αφού λένε ότι δεν κάναν τίποτα, δεν κάναν τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, σαφώς δεν είναι όλοι εγκληματίες και αυτό είναι χαζό αλλά μπορούν και αυτοί να εγκληματίσουν. Και αυτό πρέπει να ελέγξουμε τα σύνορά μας. Σελίμοβιτς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι χώρα μετανάστευσης που μεταναστεύουν δηλαδή οι νέοι από τη Βοσνία. Και τώρα φτάσαμε να έχουμε 23.000 φέτος που έρχονται στη χώρα και λέμε σαν χώρα διέλευσης και θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα. Οπότε οι υποδομέ είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Η χώρα έχει μόνο δύο κέντρα για του έντοντες άσυλο Και στο γόνατο προσπαθούν να αυτοσχεδιάσουν. Ε, χρησιμοποιούν εγκαταλειμμένα εργοστάσια κλπ. Μα δυστυχώ, με θερμοκρασίε κατά το μηδέν κοιμάται ο κόσμο έξω. Πολύ δύσκολε συνθήκε. Και όσο πάει και ο χειμώνα γίνεται βαρύτερος. Δεν έχει χώρα ούτε οικονομικά ούτε δικαιωτικά τις δυνατότητες να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε. Μέχρι τώρα βοηθάει ο απλός κόσμος. Κάνει προσπάθεια φιλότιμη προσπάθεια με, με δεδομένο των δυσκολιών αλλά τα πράγματα στα σύνορα είναι πάρα πολύ δύσκολα έχουμε και φαινόμενα βίας, τα έχουν πει άνθρωποι που είναι επιτόπου και το Human Rights Watch και μας είπαν ότι οι διοκτικές αρχές χρησιμοποιούν βία, βία κατά και οι, οι Κροάτες αστυνομικοί πρόχνουν τον κόσμο πίσω στην ε, Βοσνία. Πρέπει αυτό να σταματήσει, να ερευνηθούν τα φαινόμενα και μπράβο στην Επιτροπή που ανέλαβε την πρωτοβουλία. Θα πρέπει, θα πρέπει να βοηθήσουμε στην χώρα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κόμπερν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χριστός ήταν μετανάστης. Όχι, δεν θα πρέπει κανείς να είναι έτσι σκληρός, βάρβαρος με αυτούς τους φουκαράδες που υποφέρουν. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα. Πιο πολλά λεφτά, πιο πολλή βοήθεια. Έτσι όμως ενθαρρύνουμε περισσότερους μετανάστες. Ή κάποιους που είναι οικονομικοί μετανάστες. Δεν τους κατηγορώ. Και εγώ στις τα θα κάνω. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τους χωρέσουμε. Ούτε για μας δεν έχει τις δουλειές. Δεν συμφωνείτε ότι το να δίνουμε κι άλλα κι άλλα λεφτά θα ενθαρρύνουμε να έρχονται περισσότεροι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σελίμωβιτς, ευχαριστώ κύριε Κόμπερν για την ερώτηση. Διαφώνω. 100% μαζί σας γιατί το να μπορούμε να βοηθήσουμε μια χώρα αυτό δεν το ξέρουν οι μετανάστες. Ούτε κακό ούτε καλό είναι για αυτούς. Δεν θα έρθουν εξαιτία αυτού δεν θα σταματήσουν να έρχονται εξαιτία αυτού. Απλώ βολεύουμε τι χώρε που εντοπίζουν την κατάσταση για να μπορέσουν με έναν ανθρώπινο τρόπο να ενεργήσουν. Είναι υποχρέωσή μα. Ευχαριστώ. Μπίλτε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο σκληρός βαλκανικός χειμώνας δεν μπορεί να αποκρύψει μια πραγματικότητα που ακόμα και ο συντονιστής του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση στο Σεράγεβο το λέει και αυτός ξεκάθαρα. Το 80% των προσφύγων είναι οικονομικοί μετανάστες. Μπροστά σε αυτή την πλημμυρίδα των μεταναστών δεν πρέπει να κρύβουμε την πραγματικότητα. Η προσπάθεια να περάσουν από τα Βαλκάνια ε, έχει πλέον επιτυχία. Τα τρία τέταρτα περνούν από τη Βοσνία Ευζεγοβίνη, έρχονται ελεύθεροι στην Ευρώπη ε, και δεν θα απελαθούν ποτέ. Ποιος φταίει, μα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ευχαριστημένη, αλλά στο δίνει, ξοδεύει τεράστια ποσά ε, μόνο και μόνο για να βοηθά τους ε, ε μετανάστες. Υπάρχουν βέβαια δυνάμεις στην Κροατία οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μία μάστιγα μπροστά στην οποία οι υπόλοιποι υποκύπτουν. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πλαίσιο ασφάλειας για όλους. Ε, και οι καταστάσεις που εξελίσσονται στη Βοσνία, Ευζεγοβίνη και την Κροατία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα ε, τα σύνορα κάθε χώρας είναι κοινά εξωτερικά σύνορα, ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες του Σέγγεν για την διαχείριση αυτών των εξωτερικών σύνορων και σε σχέση με τις θεωρήσεις και σε σχέση με τους επαναπατρισμούς θα πρέπει ε, φυσικά να βρούμε τελικές λύσεις έτσι ώστε να αξιολογήσουμε σωστά τη λειτουργία του Σέγγεν και να εντοπίσουμε ε, τις καταστάσεις οι οποίες απαιτούν τη λήψη άμεσα μέτρων. Αυτό δεν σημαίνει πολιτική ανοιχτής θύρας, σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αμφισβητηθούν οι αρχές του ανθρωπισμού. Αυτό το οποίο είναι χειρότερο είναι η αδράνεια από πλευράς κρατών μελών και η ανικανότητά τους, τις οποίες στο Κοινοβούλιο εμείς ζητάμε να δημιουργηθούν χρόνια. Θέλουμε ένα σύστημα επαναπατρισμού αποτελεσματικό, θέλουμε μια εξωτερική υπηρεσία συνόρων αποτελεσματική, και δυστυχώς ε, οι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν την αδράνεια των πολλών. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η... Σε όλη τη διάρκεια του 2018 η Κροατία έχει δει δραματική αύξηση των διελεύσεων συνόρων από την Βοσνία. Κατά 57% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Να σας πενθυμίσω πως η Κροατία έχει τα πιο εκτεταμένα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύοντας αυτά τα σύνορα βεβαίως δεν κάνει ό,τι οι γειτονικέ χώρες που προστατεύουν τα σύνορά τους με σειρματοπλέγματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6.500 άτομα στην Βοσνία, περισσότεροι σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς κοντά στα σύνορα. Εμείς ως κράτος μέλος ε, αναμένουμε προσεχώς να μπούμε στην ε, ζώνη Σέγγεν και γνωρίζουμε πως η μετανάστευση είναι μια παγκόσμια στήριξη. Γι' αυτό υποστήριξαμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο στο Μαρακές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα να αναμένει από τα κράτα μέλη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διώξει ως παραπέζουν αυτά τα δικαιώματα. Ταυτόχρονα πρέπει να βοηθήσει τις χώρες που έχουν περιορισμένα οικονομικά μέσα και πολύ εκτεταμένα σύνορα που αντιμετωπίζουν το τεράστιο αυτό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριο και ένα λεπτό και 30. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Κροατία. Ε, πολύτως ε, δικαιολογημένα δρά. Έχει κάθε δικαίωμα να προστατεύσει τα σύνορά τη, που είναι και εξωτερικά σύνορα τη Ένωση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι προστατεύει όλου μα. Η Κροατία ε, δεν μπορεί να κατηγορείται επειδή κάνει το σωστό. Οπότε ας μην ενθαρρύνουμε το έγκλημα. Γιατί η παράνομη διέλευση των συνόρων είναι έγκλημα. Δεν είναι μια απλή παρατυπία. Και δεν μπορούμε να το ενθαρρύνουμε. Τα συνότα περνάμε στα κατάλληλα φυλάκια. Οπότε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση που ενθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση παραβιάζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Η παράτυπη μετανάστευση δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Η προστασία της ευημερίας των πολιτών μας είναι αντιθετός υποχρέωση των κρατών μελών. Υπάρχει μπλε κάρτα? Ναι. Την δέχεστε? Ας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση στον συνάδελφο. Συνέχεια λένε ότι δίνουν κίνητρο σε λάθρο μετανάστευση. Εμείς που λέμε ότι παντρεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα πρέπει επαρκώς να πιάνουν τόπο τα λεφτά της Ένωσης που ανήκουν σε όλους τους Ευρωπαίους. Μας λένε λοιπόν Ούτε κακώ λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έφτακτη κατάσταση στα σύνορα, να σεβόμαστε τις συμφωνίες μας και τα σχετικά με την αποδοχή των ε, μεταναστευτών. Επομένως, από πού και ω πού, κύριε συνάδελφε, εμεί θέλουμε λάθρο μετανάστευση. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Πολλοί συνάδελφοι εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα ενθαρρύνουν την παράνομη μετανάστευση. Την δικαιολογούν. Είναι συνήγοροι εδώ πέρα της ε, λαθρομετανάστευσης. Αυτό βλάπτει τους πολίτες μας. Βλάπτει τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών. Η παρανοϊκή ιδέα ότι είναι κάποιο δικαίωμα αυτό δεν ισχύει. Σας ευχαριστώ, Ράντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Κροατία βρίσκεται σε μια κατάσταση που οι γειτονικές χώρες άνοιξαν τα σύνορά τους γιατί δεν μπορούν να τα ελέγξουν και να ελέγξουν τις ροές και οι χώρες που δέχονται μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι υπόλοιπες χώρες ε, προσβοράν, έχουν βάλει σειρματοπλέγματα. Οπότε είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Έχουμε υπογράψει διάφορες ε, διεθνείς ε, συνθήκες και το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Ταυτόχρονα όμως δεν έχουμε αναπτύξει τρόπους να τις τηρήσουμε. Γι' αυτό έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα μιλάμε για την έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που λέει ότι το σύστημα αυτό μεταφοράς ε, προσφύγων ε, και τον τον άσυλο δεν λειτουργεί, δεν εφαρμόζεται. Ταυτόχρονα λέει ότι κάποια κομμάτια εδώ αφορούν την διέλευση παραβιάζουν τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ε, δηλαδή πρέπει να δούμε ποια είναι η αλληλεγγύη με χώρες και μη ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την αστυνομία της Κροατίας που κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά με μεγάλο επαγγελματισμό. Προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα από τις παράνομες διελεύσεις και έτσι προστατεύουν τους Ευρωπαίους και Κροάτες πολίτες. Πάνω από 2.000 ε, άτομα ε, μπήκαν ε, Πάνω από 20.000 άτομα μπήκαν στην Βοσνία Ζεκοβίνη. 4.000 ζήτησαν ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 4 εκατομμύρια για την στέγασή τους και από την αρχή της κρίσης έχει δώσει 31 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βοηθήσουμε τις αρχές της ε, Βοσνίας και τους διεθνείς οργανισμούς για να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη. Πρέπει να αυξηθεί η βοήθεια προς την Βοσνία για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στα αιτήματα και να επαναπατρίσει όσους δεν ε, λαμβάνουν άσυλο. Η Βοσνία και η Ζεγοβίνη πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτά τα κονδύλια για να καταπολεμήσει την ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό που ε, αυξάνεται στη χώρα. Ε, οι άνθρωποι στη Βοσνία πάντα ζούσαν ε, εν ειρήνη και ανεκτικότητα. Σήμερα όμως βλέπουμε άλλες αξίες να εξαπλώνονται που απειλούν την ασφάλεια της περιοχής. Πρέπει να σταματήσουν τα λεφτά που ενισχύουν την ριζοσπαστικοποίηση, όπω και η ριζοσπαστικοποίηση η ίδια, αν θέλουμε να αποφύγουμε τι τραγωδίες που βλέπουμε στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Κιέγγε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά το κλείσιμο των συνόρων στην Ουγγαρία εύκολα να φανταστεί κανείς ότι ο βαργανικός διάβλος μετακινήθηκε και το καλοκαίρι η κατάσταση στα βοσνιοκροατικά σύνορα κατέστη χειρότερη και ήδη έχουν καταγραφεί καταπατήσεις των δικαιωμάτων και υπάρχουν κερνά στο νόμο σε σχέση με το άσυλο. Τον χειμώνα κατάσταση πρόκειται να γίνει χειρότερη και έχουμε τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες οι οποίοι συνεχώς αποθούνται και ε, γίνονται παιχνίδι στα χέρια των διακινητών και βοηθάει και η αστυνομία. Έχουμε τουλάχιστον 5.000 οι οποίοι κινδυνεύουν από το κρύο, από την έλλειψη τροφίμων ε, και η υγειονομική κατάσταση είναι κακή. Είναι ιερή ανθρώπινη ζωή, πρέπει να γίνεται σεβαστή και το είπαμε την ευκαιρία του διαλόγου για το Παγκόσμιο Σύμφωνο στο Μαρακές πριν από λίγες μέρες. Είναι παγκόσμιο σύμφωνο, παγκόσμιο φαινόμενο η μετανάστευση και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και από εμά. Δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε Κροατία και Βοσνία σε αυτή την κατεπίκουσα κατάσταση και σας υπενθυμίζω ότι είχαμε την αρχή της χρονιάς 23.000 που μπήκαν στην Βοσνία και είχαν όνειρο την Ευρώπη. Το λέω συνέχεια. Δεν σταματάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σύνορα για όλους, για τους μικρούς και τους μεγάλους. Άρα θα πρέπει άξονά μας και, και κίνητρό μας να είναι η ανθρωπιά μας. Και θα πρέπει να δεσμευτούμε όσον αφορά το καλό όλων των ανθρώπων. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μόνιμο συζητητή για την Βοσνία, οπότε και φυσικά παρακολουθώ από κοντά όσα γίνονται στην χώρα. Αυτά τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την μετανάστευση πήγα επί τόπου στα σύνορα για να δω πώς διαχειρίζονται την κατάσταση. Όμως, με το που ήρθε ο χειμώνα, η κατάσταση έγινε δύσκολη. Οπότε έχουμε εκτός από αυτούς που μπαίνουν στη Βοσνία και αυτούς που αποθούνται από την Κροατία. Έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα ε, και βλέπω τι γίνεται εδώ πέρα στο ημικύκλιο από την ακροδεξιά λένε ότι ο Πούτιν έχει βάλει το δάχτυλό του ε, στις ε, προεδρικές εκλογές. Ναι, ναι. Το είπε και ο Επίτροπος. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Κροατία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει περισσότερη νυφαλιότητα στον πολιτικό βίο της χώρας. Και τώρα ξεκινάμε το Catch the Eye, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε πέντε συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Ξεκινούμε με την κυρία Ζόφκο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πιστεύω Ότι είπε ο κ. Μπρέντα, ο συγητής μα για Βοσνία Ζεγοβίνη, ότι έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα των προσφύγων στη χώρα. Υπάρχει δυσλειτουργία από πλευρά κυβέρνηση. Δεν είναι πρόβλημα τα χρήματα μαζεύονται οι πρόσφυγες, θα συνομιλούν με την Κροατία και η Κροατία πρέπει να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προστατεύσει τα σύνορα της Ένωσης. Όλα αυτά τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο. Θα πρέπει το Σαραϊβό να ξέβρει κάποια λύση, να ενεργήσουν με σοβαρότητα, να συνοηθούν με τη διεθνή κοινότητα, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε στην πηγή του να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν αρκετά χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουν τους μετανάστες στα σύνορα της Ένωσης. Είναι και θέμα ασφάλειας. Η κυρία Γκραπίνη. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτά τα οποία είπατε. Η κατάσταση για τους τοπικούς πληθυσμούς είναι πολύ δύσκολη. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε, να καταδικάσουμε και να κατηγορήσουμε τη Βοσνία και την Κροατία. Θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε ότι προφανώς δεν έχουν βρει λύσεις τα πάντα. Οι διαδικασίες για το άσυλο είναι αυτές οι οποίες είναι, αλλά δυστυχώς η καθημερινότητα είναι διαφορετική. Υπάρχουν προβλήματα με την τρομοκρατία. Ξέρετε τι συνέβη στο Στρασβούργο πριν μερικές μέρες και ακόμα και ένα σωστά προετοιμασμένο κράτος ε, θα δυσκολευτεί να προετοιμάσει τις σωστές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Απαιτείται λοιπόν μια σωστή ανάλυση για το τι συμβαίνει σε σχέση ε, με την μετανάστευση. Προφανώς και θα πρέπει να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προφανώς ε, και αναφέρομαι εδώ σε αυτούς οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες. Ο κύριος Μαριάς ακούστηκε από τους συναδέλφους ότι υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στα σύνορα της βοσνίας με την κροατία. είπατε ότι 5.500 πρόσφυγες συνοστίζονται. φανταστείτε λοιπόν τι πρόβλημα υπάρχει στο νησί της σάμου όπου μόνο σε ένα νησί υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες. αλλά δεν άκουσα προτάσεις δεν άκουσα να δίνονται λύσεις μόνο ευχολόγια. ερώτημα πρώτο πώς έχουν φτάσει στη βοσνία αυτές οι χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες με ποιο τρόπο πέρασαν από άλλες χώρες είπατε ότι προέρχονται από την τουρκία πώς έφτασαν όμως μέχρι τη βοσνία μήπως υπάρχει κάποια αεροπορική σύνδεση με την turkish airlines ποιος έχει ευθύνες που φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί αυτό πρέπει να αναζητήσουμε. και δεύτερον οπωσδήποτε υπάρχουν υποχρεώσεις της βοσνίας διότι έχει και συμφωνία σύνδεσης με την ευρωπαϊκή ένωση όσο δε για την κροατία που κάποιος συνάδελφος είπε να μπει η κροατία στη σέγγεν σας λέω ότι αν μπει η κροατία στη σέγγεν θα είστε μαγνήτης για περισσότερους πρόσφυγες και παράνομους ε. μετανάστες όπως γίνεται με την περίπτωση της ελλάδας. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Ward. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ντροπή, συνάδελφοι της άκρας δεξιάς, που εκμεταλλεύεστε ε, την τραγωδία της Τρίτης το βράδυ για να προωθήσετε τις ισλαμοφοβικές σας απόψεις. Η μετανάστευση είναι ένα ανθρώπινο φαινόμενο. Όταν η ζωή είναι ανυπόφορη λόγω οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή κλιματικών αλλαγών, οι άνθρωποι μετακινούνται και τα προβλήματα που δημιουργούνται πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο φίλος μου Γιουρίσιτς είναι πρόσφυγας από το Βαλκανικό πόλεμο, από τη Βοσνία. Ξέρει τι σημαίνει απώλεια και τι κάνει. Βοηθάει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην δική της χώρα και τους βοηθάει επίσης και εδώ στη Γαλλία στην οποία έχει βρει μια δεύτερη πατρίδα. Είναι αυτή η οποία στο Παρίσι συνεργάζεται με το κέφο Καλέ ε, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι μετανάστες. Η κυρία Σλάιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ικανοποιημένη που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδέησε για να συζητήσει την ε, κατάσταση στην Βοσνία και την Κροατία. Πριν τέσσερις μήνες είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρεις μήνες συγγνώμη, να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρώπων αυτών, των εγκαταλελειμμένων αυτών ψυχών στην Βέλικα Κλάντουσα. Ε, το Human Rights Watch ε, έχει επιβεβαιώσει ότι ο τρόπος με τον οποίο διαβιούν οι άνθρωποι αυτοί είναι απαράδεκτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τη συστηματική βία την οποία ασκεί η, ε, κροατική, οι κροατικές δυνάμεις ασφαλείας. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει μια απάντηση που να σέβεται την ανθρώπινη προσωπικότητα. Και δεν αναφέρομαι σε ε, επαναπροωθήσεις βίαιες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο σε χώρες όπως η Κροατία. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας έλεγχος, μια έρευνα γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς υποφέρουν. Ο κύριος Ανδρουκάητης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και έντονη. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι διαφωνώ με όσους κατηγορούν την Κομισιόν. Απολύτως. Βεβαίως όλοι είμαστε υπεύθυνοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά μην κατηγορούμε ένα τον άλλον και την Κομισιόν γιατί έχουμε εμπλακεί ε, ουσιαστικά κάθε μέρα εκεί πέρα. τα προβλήματα. Αντέδρασε αμέσως η Ευρωπαϊκή Ένωση με ανθρωπιστική χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις άμεσες ανάγκες ε, μεταναστών και προσφύγων ε, που διοχετεύεται μέσω εταίρων όπως οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και αφορά την παροχή τροφίμων, ε, ρούχων, υπηρεσιών υγείας και στέγης. Γνωρίζουμε βεβαίως πως το είναι χειμώνας Επιπλέον, ε, η Κομισιόν έδωσε 7,2 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθούν οι ικανότητες ταυτοποίησης και προστασίας για να στηριχθεί η συνοριοφυλακή της Βοσνίας και για να δοθεί και επαρκή στέγαση για το χειμώνα. Η Κομισιόν συνεχίζει να παρέχει σημαντική στήριξη στη Βοσνία Ζεγοβίνη και στους Δήμους που πλήττονται. Και βεβαίως η στήριξη αυτή προστίθεται στα 24,6 εκατομμύρια ευρώ που έχει ήδη δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 ε, για το θέμα αυτό ακριβώς. Να σας διαβεβαιώσω πως είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση της Κορατίας για την εφαρμογή των κανόνων ασύλου και επανεισδοχής. Και τώρα υπάρχουν κατηγορίες ε, κακομεταχείρισης ή το ότι δεν τους δίνει τη δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο. Τα ερευνούμε αυτά και θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θεωρούμε ότι η Κροατία θα δώσει συνέχεια στις καταγγελίες και θα συνεχίσει τη συνεργασία με τη Βοσνία. Ταυτόχρονα η Κομισιόν υπενθυμίζει την ανάγκη η Βοσνία να εντείνει τις ε, προσπάθειές της ε, συντονισμό και βεβαίως ε, να εφαρμόσει τις σχετικές διαδικασίες. Τι θα πρέπει και η κυβέρνηση της χώρας να ενισχύσει τις δυνατότητες επίλυσης του ζητήματος. Τέλος, να σας διαβεβαίωσω πως η Κομισιόν καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να αποφύγει την επιδείνωση της ε, κατάστασης. Ε, βεβαίως, ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Και εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Και σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. τα κατεπήγοντα και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συζητήσουμε λοιπόν το Ιράν και συγκεκριμένα την περίπτωση της ε, Νασαρίν Σούτουντε. Τον λόγο έχει κυρία Χάουταλα. Ναι. Καλημέρα Πρόεδρε, Επίτροπε. Συζητούμε τώρα την υπόθεση Νασρίν Σούτουντεχ συγκεκριμένα τα της διώξεώς της. Είναι δικαιός με ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πάρα πολύ γενναία και καταδικάστηκε για το έργο της, για τη δουλειά της στο Ιράν. Προσπαθούσε να μην φορούν ε, το, τη, τη μαντήλα οι, οι γυναίκες. Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς την χειράβηση των γυναίκων και γι' αυτό και τόσοι ακτιβιστές ε, τώρα προσπαθούν στο Ιράν για αυτό το λόγο, γιατί είναι σημαντική δύναμη της χώρας οι γυναίκε. Οπότε, αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε είναι η άμεση αποφυλάκηση της Νασρίν Σοτουντέ. Είχε κερδίσει το βραβείο Ζαχάρ το 2012. Οπότε έχουμε ιδιαίτερα έντονη υποχρέωση να τη βοηθήσουμε για τη δουλειά της. Ε, αυτό κάνουμε για κάθε βράδυ με τον Ζαχαρόφ. Φυσικά και οι διπλωματικοί διάβλοι χρησιμοποιούνται, αλλά τώρα θα πρέπει και εμείς να προτάξουμε ε, αυτή μας την μέρημνα εδώ στο Κοινοβούλιο και για αυτό ζητούμε η αντιπροσωπεία στο Ιράν που εκπροσωπεί την Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, να συνεχίσει να παρακολουθεί τις ε, εξελίξεις να την επισκεφθεί στην φυλακή και να απαιτήσει την αποφυλάκησή της. Επίσης, αυτό το ψήφισμα αφορά και το ότι πρόσφατα ανησυχούμε για τις βιωτικές συνθήκες του κόσμου στο Ιράν. Ε, η ξηρασία τους έχει πλήξει, οπότε ακριβώς ε, περνούν δύσκολες ώρες. Και ακριβώ είναι και θέμα των συνεπειών του εμπάργου των ΗΠΑ κατά του Ιράκ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που σήμερα ασχολούμαστε με το θέμα της ε, Ναστρίν, ε, μιας ε, πιθανούς δικηγόρου. Η παρενόχληση των δικηγόρων και ανθρωπιστών πραγματικά είναι ενισχυτική και υπάρχει έλλειψη βασικών πολιτικών δικαιωμάτων στο Ιράν με το θεοκρατικό καθώς βεβαίως ε, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απελευθερωθεί αμέσω, αλλά δεν είναι μεμονωμένη αυτή η περίπτωση. Εγώ υποστηρίζω την ε, οργάνωση αυτή αλλά και την σχετική συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε στην δραματική κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης ε, γύρεται το ζήτημα ανθρώπων με δύο υπηκότητες ε, που κρατούνται στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Η χώρα αυτή, η περίπτωση αυτή με συγχωρείτε, επηρεάζει τις σχέσεις του Ιράν με την Βρετανία και ελπίζω να προλάβει να γυρίσει στην οικογένειά της ε, στη Βρετανία για τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ, Ernst, για ένα λεπτό και 30. Ναι, θα ήθελα να αναφέρω τρία πράγματα. Πρώτον, είμαστε αλληλέγγυοι χωρίς ε, ναι με όλους τους ανθρώπους ε, του Ιράν που παλεύουν κατά της ε, διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Γιατί η ζωή τους έχει γίνει αφόρητη. Με τους συνταλικέριδες που δεν πληρώνονται. Με τους ανθρώπους που παλεύουν για το κλίμα. Ε, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να συλλαμβάνεται μόνο και μόνο επειδή διαδηλώνει. Δεν είναι δυνατόν να του ρίχνουν στη φυλακή επειδή διαμαρτύρονται. Είναι απαράδεκτο. Δεύτερον, ζητάμε την άμεση απελευθέρωση της Νασρίν Σούτουντε και του συζύγου της. Ε, είναι μια θαραλέα γυναίκα που παρέμεινε στο Ιράν και εκπροσωπεί τις γυναίκες που παλεύουν για την ελευθερία τους. Για μένα είναι αδιανόητο μια γυναίκα που έχει λάβει το βραβείο Ζαχάροφ να φυλακίζεται. Στηρίζουμε τις ιρενές, αλλά και τις γυναίκες εκείνες που κρατούνται γιατί δεν φοράνε τη μαντήλα. Οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και έτσι πρέπει να μείνουν και να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Είναι το ελάχιστο. Και το τρίτο, ναι, στηρίζουμε την συμφωνία για τα πυρηνικά γιατί δεν θέλουμε πυρηνικούς ανταγωνισμούς και έχει επιτέλους ε, φτάσει η στιγμή να σταματήσουμε τον πρόεδρο των ΙΠΑ που συμπεριφέρεται σαν έρωνας. Η Ευρώπη χρειάζεται μια δική της πολιτική στην Μέση Ανατολή και να αντισταθεί στις κυρώσεις ε, των ΙΠΑ. Κύριε Γκόμες, για ένα λεπτό φυλακίστηκε η Σουτουντέ και ήταν φυλακιασμένη όταν είχαμε δώσει το βραβείο. Ποτέ δεν μπόρεσε να έλθει να μας συναντήσει. Εξακολουθεί ε, να είναι φυλακισμένη επειδή φροντίζει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ο άνδρας της επίσης ε, φυλακίστηκε ε, διότι διαμαρτυρήθηκε για την κράτησή της. Ε, γελίες κατηγορίες δείχνουν την τραγωδία στην οποία ζει το Ιράκ. Πρόκειται για ένα λαό με πολύ μεγάλη ιστορία και δυστυχώς διοικείται από ένα αρχαϊκό καθεστώς το οποίο ε, επιβάλλει τυφλή καταστολή. Ε, έγιναν κάποιοι νόμοι οι οποίοι επιτρέπουν σε πάρα πολλούς ε, ε, Ιρανούς να γλιτώσουν την θανατική εκτέλεση. Δυστυχώς όμως οι υπόλοιπες κατασταλτικές διατάξεις εξακολουθούν να καταπιέζουν τους πολίτες του Ιράν. Το Φεβράριο είχα πάει στο Ιράν και ένιωθα ότι ο κόσμος μιλούσε πιο ελεύθερα Γι' αυτό ζητάμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών προσφύγων Ευχαριστώ η κυρία Σάκε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Σουτουντέ είναι μία από τις πιο θαραλές υπερασπίτριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Η οικογένειά της και αυτή η ίδια πληρώνουν υψηλότατο τίμημα μόνο και μόνο γιατί κάνει σωστά τη δουλειά της. Εμείς έχουμε ευθύνες επειδή δώσαμε το φαφείο Σαχάροφ να απαιτήσουμε την απελευθέρωσή της. έχει υπερασπιστεί τις θαραλές γυναίκες οι οποίες θέλουν να αποφασίζουν αυτές το αν θα φορούν ή δεν θα φορούν χιτζάπ. Και είναι σημαντικό η κυρία Μογκερίνη και δημόσια και ιδιωτικά να μπορούν να υπερασπίζονται, να μπορεί να υπερασπίζεται τη γυναίκα αυτή και τα δικαιώματα των Ιρανών και κυρίως των γυναικών οι οποίες ε, απλά έχουν δίκιο όταν ε, θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωμένες να φορούν συγκεκριμένα θρησκευτικά σύμβολα. Ο κύριος Κέλαμ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι συμβολικό της κατάστασης στο Ιράν ότι ακόμα και μια επιφανής ε, υπερασπιστήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βραβείο Σαχάροφ ε, να κρατείται εδώ και μήνες γιατί παραβίασε τον νόμο περί καλύπτρας ε, της κεφαλής. Πρόκειται λοιπόν για μέρος των διαμαρτυριών που συνεχίζονται σε όλο το 2018. Συμφωνώ με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας πριν από λίγες μέρες που λέει το Ιράν αντιμετωπίζει μια πολύπλευρη κρίση οικονομική, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και περιβαλλοντική. Αντιδρώντας, οι αρχές εντείνουν την καταστολή. Το θέμα πλέον δεν αφορά μικρές ομάδες, αλλά πολύ διαδεδομένε απεργίες οδηγών φορτηγών, δασκάλων, εργατών, φοιτητών, εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που εξεγείρονται για τις ε, δραματικές ε, συνθήκες ε, για την διαφορά και την καταστολή. Οπότε απαιτούμε πρώτα απ' όλα την άμεση απελευθέρωση της κυρίας Σουτουντέ. Όμως το να απευθύνουμε απλά εκκλήσεις δεν αρκεί για να έχουμε ένα πραγματικό αντίκτυπο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες να ακολουθήσουν μια διαφορετική συνταγή. Εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με ψηφίσματα. Οποιαδήποτε βοήθεια θα πρέπει να είναι υπό τον όρο ουσιαστικής βελτίωσης των ελευθεριών των πολιτών και της ελευθερίας έκφρασης. Τίποτα λιγότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει την διαφορά αρκεί να συνδέσουμε την Realpolitik με τις αξίες μας. Σας ευχαριστώ κυρία Σόιντροβα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Ιράν ε, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια κρατούνται άνθρωποι ε, μεταξύ των οποίων ε, και η κυρία Σουτουντέ και πολλές ε, γυναίκες που έβγαλαν την μαντήλα. Και τώρα η κυρία Σουτουντέ κάνει απεργία πείνας. Έχει λάβει το βραβείο Ζαχάροφ. Παλεύει για την ισότητα ανθρώπων και γυναικών, για τα δικαιώματα θρησκευτικών μειονοτήτων που δεν γίνονται σεβαστά έτσι, πραγματικά κινδυνεύει η ζωή της. Ε, υπάρχουν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι στο Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα ζητάει την απελευθέρωση της Νασρίν και άλλων πολιτικών κρατουμένων. Το θέμα λοιπόν εδώ πέρα δεν αφορά ένα πολιτικό κόμμα. Όλες οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου το ζητάνε αυτό και αυτή είναι η δύναμή μας. Σας ευχαριστώ λέει ο κύριος Χόλτσερ ε, Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όταν είχε τιμηθεί η κυρία Σότουντε με το βραβείο Ζαχάροφ, επίσης ήταν στη φυλακή. Και λέγαμε τότε ότι όταν αφέθηκε ελεύθερη ε, είχαμε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Και η αντιπροσωπεία τότε του Κοινοβουλίου μπόρεσε να την συναντήσει και εντυπωσιάστηκε πραγματικά. Λοιπόν, η κράτησή της τώρα είναι πάλι σοκαριστική και είναι ένα καμπανάκι. Ζητάμε από το Ιράν να ε, λάβει στα σοβαρά το δικαίωμα του διαλόγου, ειδικά επίσης ε, στην περίπτωση ατόμων με διπλή υπηκότητα όπως και η κάμαραν Καντέρη. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή η κυρία Σούτουντέ και η κυρία Πάναγη που επίσης κρατείται εδώ και έξι χρόνια να έρθουν επιτέλους στο Στρασβούργο για να παραλάβουν το βραβείο τους. Σας ευχαριστώ Μπέλτερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ε, παραμένει μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Παραδείγματος χάρη ε, υπάρχει ακριβώς η ανησυχία για το καθεστώς ε, και το εάν και κατά πόσον μπορεί να σταθεί. Το ψήφισμά μας λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Η δίωξη της κυρίας ε, Σότουντε είναι ενδεικτική για την κατάσταση στην χώρα. Έχουμε επίσης την ε, σύλληψη χριστιανών 102 τον προηγούμενο μήνα και τον Δεκέμβριο μέχρι στιγμής πάνω από 100. Έχουμε βάρβαρη δίωξη των χριστιανών που θα πρέπει να καταδικαστεί. Αναμένω λοιπόν να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα που θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανεξιθρησκεία στο Ιράν. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπετσέρα Βαστερετσέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Δύση περνά στιγμές φεμινιστικές. Δηλαδή πρόκειται για τις ανισότητες βάσει των γυναικών, αλλά θα πρέπει να τα μάτια γιατί γίνεται σε άλλες μακρινές χώρες. Είδαμε τι έγινε στο Ιράν όταν διαμαρτύρεται για κάτι πολιτικό κάποια γυναίκα. Αυτό είναι κάτι ηρωικό γιατί ξέρει ότι μπορεί να κατάξει στη φυλακή, αλλά δεν αφορά μόνο μόνο αυτέ τι τις γυναίκε. Γιατί και η γυναίκα αυτή, η δικηγόρο των ανθρώπινων δικαιώματων που πήρε το Ζαχάροφ και πάλι φυλακίστηκε αυτή τη φορά γιατί περασπίστηκε τι γυναίκε που κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο διαμαρτυρηθούν. Αν πιστεύουμε στην ισότητα, θα πρέπει να τίνουμε μια χείρα βοηθεία προ την ε, γυναίκα αυτή. Αν πιστεύουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ούτω ώστε κάτι να γίνει για αυτέ τι εξαφανίσει, τι δεκάδε χιλιάδε και εκτελέσει που έχουν γίνει η δεκαετία του 80 στο Ιράν. Πρόκειται για αξίε ανθρώπινε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε αυτόν τον τομέα πρωτοπόρα. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ένα λεπτό, κυρία Πάρκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τίποτα ε, δεν είναι πιο σημαντικό μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου από τα θρησκευτικά πιστεύω. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα αλλά πολύ λίγοι απολαύουν αυτό το δικαίωμα. και για κάποιε γυναίκε η μαντήλα είναι εκδήλωση πίστη, για άλλου είναι εκδήλωση καταπίεση. Αλλά θα πρέπει να είναι δικαίωμα τη γυναίκα να διαλέξει αν θα το φορέσει και πώ θα τοποθετηθεί, πώ θα εκφραστεί. Οι Ιρανέ δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Υπάρχει κοινωνική πίεση, υπάρχει καταστολή από το δίκαιο, από το κράτο. Προβολή τη αξιοπρέπεια είναι αυτό. Θα πρέπει το Ιράν να αφουγκραστεί τι θέλουν οι πολίτε. Θα πρέπει να καταργηθούν αυτοί οι κατα... σταλτικοί νόμοι. Θα πρέπει να δώσω το δικαίωμα επιλογή στους Ιρανού. Φόικτ δεν παρίσταται. Τζανονάτο. Κύριε Τζανονάτο. Θα συμφωνήσω με αυτούς που ζητούν η Σουτουντέ να επελευθερωθεί άμεσα και όλοι όσοι προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι στη φυλακή μόνο και μόνο γιατί θέλησαν να εκφραστούν ελεύθερα. Ανησυχώ για την χειροτέρευση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι ο διάλογος με τη χώρα αυτή ε, πρέπει ε, να ενισχυθεί. Νομίζω ότι η συμφωνία επίσης για την πυρηνική ενέργεια στο Ιράν πρέπει να παραμείνει ε, θα έλεγα ζωντανή γιατί είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά επίσης και την κοινωνική κατάσταση. Οι αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε επηρεάζουν όχι μόνο τις οικονομικές εξελίξεις, αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις. Πρέπει να ενισχύσουμε τον διάλογο ε, με την χώρα αυτή, σεβόμενοι ε, τα δικαιώματα των πολιτών της χώρας. Ευχαριστώ. Διαδικασία Catch the Eye πλέον. Τρεις συνάδελφοι. Κυρία Πετήρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έχουν υπάρξει πάρα πολλές συλλήψεις αντιπολιτευομένων στο καθεστώς στο Ιράν. Δυστυχώς συνεχίζουν οι ε, εκτελέσεις και πάρα πολλοί είναι αυτοί που χάνουν τη ζωή τους. Συλλαμβάνονται επίσης γυναίκες και ε, συλλαμβάνονται επίσης και αυτοί που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πολιτικοί κρατούμενοι κάνουν ε, απεργίες πείνας, δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό. Υπάρχουν επίσης ε, θρησκευτικέ μειονότητες οι οποίες ε, διώκονται. Ανησυχούμε για την κατάσταση αυτή. Ανησυχούμε επίσης και για τις έρευνες στον τομέα των πυρηνικών όπλων. Θα ήθελα να μάθω τι συμβαίνει λοιπόν με τον διάλογο με την Ιρανική κυβέρνηση η κυρία Ward. Εμείς δώσαμε το βραβείο Σαχάροφ στον Ολέγκα Σεντσόφ, αλλά τέσσερις που έχουν πάρει το βραβείο. Αυτό είναι φυλακή πάντα, όπως και η Σούτιντε. Είναι ο άνθρωπος που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπέστη την επίθεση της κυβέρνησης λόγω ακριβώς του ότι κάνει τη δουλειά της θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. πρέπει να βοηθήσουμε τους μηχανισμούς προστασίας των ανθρώπων αυτών και σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καθήκον μας να παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση αυτών που έχουν βραβευθεί απαιτούμε από τις Ιρανικές αρχές άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις να απελευθερώσουν την Σουτουντέ. Να μεταφέρω και την άποψη του κυρίου Τάνοκ ζητώντας από τις Ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν την Σαγκαράη Ράτκλιφ, μητέρα τριών παιδιών, φυλακισμένη από το 16. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάμε τώρα στον κύριο Σαφχάουζερ και μετά στον κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Σαν να λάβω το λόγο με αυτή την ευκαιρία γιατί ε, αυτό το θέμα με ενδιαφέρει πολύ και θέλω να σας πω ότι εννοείται πως ε, καταλαβαίνω ότι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με αυτή την καταδίκη αλλά σας υπενθυμίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και έχω στο μυαλό μου τους ε, χριστιανούς που σε Κίνα, Τουρκία, Αλγερία διώκονται και θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Επίσης προσθέτω ότι το Ιράν έχει έναν μεγάλο πολιτισμό, σπουδαίο πολιτισμό. Πολλές φορές το έχουν επιτεθεί, είναι οι μουλάδες. Και να, είδατε τι πολιτική έχει η Γαλλία που θέλει να είναι και πυρηνική δύναμη γιατί τώρα θέλουμε ε, ανεξαρτησία, η εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνω τι θέλει το Ισραήλ, τι θέλουν οι ΙΠΑ και ε, υποστηρίζω αυτά τα οποία θέλουν. Οπότε θα πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών ε, μεγάλων δυνάμεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριος Λόπε Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χτες το Κοινοβούλιο απένιμε το βραβείο Ζαχάροφ για φέτος. Το 2012 έγινε αυτό και τιμήθηκε η Νασρίν Σοτουντέχ, αυτή η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη. Στο Ιράν, ο Αλή είναι ο ανώτατος ηγέτης και το 18 Διεθνής Φορές Δικηγόρων του έστειλε μια επιστολή και ε, ζήτησε την άμεση αποφυλάκηση της δικηγορού αυτής. Έχει επανειλημμένα φυλακιστεί για δίκαιους αγώνες, για την ελευθερία της έφρασης και για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και ως ε, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάντοτε ε, ήμουν υπέρ του να υπάρχει δικαίωμα υπεράσπισης και αυτή η γυναίκα επίσης να έχει δίκαιη μεταχείριση. Οπότε θα πρέπει να απαιτήσουμε την αμήση αποφυλάκηση. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Κύριε Μίμητσα, έχετε τον λόγο. Κύριε Επίτροπε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. βουλευτές. βουλευτέ. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε παγκοσμίω τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μέσω ε, οικονομική ε, πίεση και με άμεσε επαφέ με τι αρμόδιε αρχέ. Αυτό ανέκαθεν ήταν η δική μα προσέγγιση όποτε είχαμε παραβίαση δικαιωμάτων στο Ιράν και υπάρχει εκπρόσωπο και όλοι μα το έχουμε θέσει αυτό σε όλες τις συναντήσει με τι ιρανικέ αρχέ σε κάθε επίπεδο. Κανεί δεν στρατεύεται τόσο πολύ όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση θανατική ποινή. Για κάθε περιστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε του αγωνιστέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα και εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούμε τι γίνεται με την ασύρνηση του ε, και του συζύγου της, του κ. Χαμντάν. Η κυρία Σοτουντεχ ε, κέρδισε το βραβείο Ζαχαρόφ το 12 και αυτό έγινε για το έργο της, ούτω ώστε να είναι συνήγορος αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και επίσης κάποιων κατηγορουμένων ε, για τους οποίους ε, είχε απαγγελθεί θανατική ποινή οπότε για αυτές τις προσπάθειες διώχθη, εμποδίστηκε από το έργο της και τελικά καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση αφού καταδικάστηκε για εγκλήματα κατά της δημόσιας ασφάλειας. Το 2013 αποφυλακίστηκε και συνέχισε το έργο της. Οπότε και πάλι συνελήφθη τον Ιούνιο φέτος ο σύζυγός της, ο οποίος είχε κάνει εξτρατή για να αποφυλακίσει και αυτός συνελήφθη αργότερα. Επανειλημμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει το ζήτημα ενώπιον των ελληνικών αρχών από τότε που έγιναν αυτές οι συλλήψεις σε κάθε επίπεδο και στα πλαίσια του διαλόγου υψηλού επίπεδου Ένωσης Ιράν. Και κάθε φορά διαπιστώνουμε την ανησυχία μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα και για τη μεταχείριση των αγωνιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τα κρατημέλη επίσης έχουν θέσει το ζήτημα στις διμερείς επαφές με τις αρχές της χώρας. Αυτές μας οι προσπάθειες οδήγησαν σε κάποιες θετικές ε, εξελίξεις. Πριν από ένα χρόνο η χώρα τροποποίησε ε, την νομοθεσία για τα ναρκωτικά, οπότε και έτσι είχαμε μείωση των ε, εκτελέσεων κατόπιν σχετικών καταδικών. Επίσης ε, έχουμε και άλλες βελτιώσεις και είχαμε και κάποιο είδους ε, αναστολή ε, κάποιων καταδικών, θανατικών, οπότε συνεχίζουμε και πιέζουμε για την αποφυλάξη της κύριας Οντέχ και του συζύγου. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να έχουν όποιον δικηγόρο, όποιον συνήγορο θέλουν, θα πρέπει να τους επιτραπεί η επικοινωνία με τα δύο παιδιά τους. Και δεν θα πρέπει να υφίστανται οποιαδήποτε κάκο μεταχείριση. Εγκατακλείδη σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για να αποφυλακιστεί και και ο σύζυγός της. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσμου για αυτή τη συζήτηση η οποία τώρα ολοκληρώνεται και η ψηφορία θα γίνει σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα, την Αίγυπτο και συγκεκριμένα την κατάσταση των υπέρμαχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε πολλούς συντάκτες. Θα ακούσουμε πρώτη την κυρία Σολε... Α, συγγνώμη, ο κύριος τον κύριο Σολέ. Σας ευχαριστώ. Το συμβαστικό αυτό ψήφισμα, το οποίο στηρίζουν πολλές ομάδες, είναι ξεκάθαρο σε δύο μέτωπα. Πρώτα απ' όλα, είναι η πιο ισχυρή καταδίκη μέχρι στιγμής ε, της φρικτής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και δεύτερον, ε, λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει τις ευθύνες της και να δώσει προτεραιότητα στην κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον διάλογο με την Αίγυπτο. Το Κοινοβούλιο λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση με την Αίγυπτο με ένα καθιστός που έχει αφανίσει όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν στοχευμένες κυρώσεις ε, κατά ατόμων για την ευθύνη τους ε, στην τρέχουσα κατάσταση. Θα παρακολουθήσουμε στενά το Συμβουλίο Σύνδεσης σε λίγες μέρες και αναμένουμε συγκεκριμένη δράση για τους ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται στο ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τάνοκ τώρα από τους συντάκτες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ Είμαι φίλος της Αιγύπτου και στηρίζω τις προσπάθειες της κυβέρνησης ε, του κυρίου Σίση για σταθεροποίηση της χώρας και γνωρίζω και την δύσκολη κατάσταση ασφαλείας που υπάρχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Αίγυπτος αντιμετωπίζει έναν σαφή κίνδυνο από την τρομοκρατία. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για όλο και περισσότερους περιορισμούς στα βασικά πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της. Ανησυχώ ιδιαιτέρως για την ελευθερία των ΜΜΕ, τις εξαφανίσεις δημοσιογράφων. 1.500 άτομα φαίνονται να έχουν εκτελεστεί τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό δεδομένου του ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δικαστεί σε ομαδικές δίκες. Όπως μαθαίνουμε στην Ευρώπη, υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε μέτρα αντιτρομοκρατίας και να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η ισορροπία έχει διαταραχθεί στην Αίγυπτο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ιγνάτσιο Κοράου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα Επίτροπε και συνάδελφε. Για άλλη μια φορά συζητούμε για την Αίγυπτο. Είναι πρωταθλήτρια στην παραβίαση των δικαιωμάτων χρησιμοποιούν το ηλεκτροσόκ ακόμα και στα γενικά όργανα των παιδιών. Ένα μικρό παράδειγμα. Έχουν περάσει ψηφίσματα, διεθνή διαβήματα, εκθέσεις, μικιό, αλλά τίποτα. Απλώς μια υπεροψία και γενική ατιμορρησία. Και ένας δικός μας, ένας Ιταλός, Ευρωπαίος, ο Τζούλερ Τζένι, ο οποίος βασανίστηκε και δολοφονήθηκε εδώ και λίγα χρόνια. Θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας με αυτό το ψήφισμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά αν θέλει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα τι είδου εκβιασμό είναι αυτό από την Αίγυπτο. Πώ είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να ανεχόμαστε τέτοιε ε, παραβιάσει δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Το 2013 ο Αιγυπτιακός στρατός εκατοντάδες σκότωσε, διαμαρτυρώντουσαν στην πλατεία Ραμπά και κανείς από αυτούς δεν δικάστηκε αλλά 75 ε, διαδηλωτές καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ακόμα ένα παράδειγμα της γενικής, γενικευμένης καταστολής και ατιμορρησίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια 65.000 πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν και επίσης εξαφανίστηκαν πάνω από 1500 και εκεί οι γνωστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώκονται οι γυναίκες όπως η Αμάλ Φατίχ έχουν φυλακιστεί δεν υπάρχει καμία προστασία για τέτοιες γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας αυτούς που ζητούν ε, ε, άσυλο από Σουδάνιε, Εμένη, Συρία, τούτους ε, επαναπροωθούν. Να τι κάνουμε. Και ήμουν συνεργάτε μα στη μεταναστευτική πολιτική και στο εμπόριο. Άρα θα πρέπει να διακοπεί, να καταργηθεί η Συμφωνία Σύνδεση, όλα τα προγράμματα ενίσχυση. Μέχρι ότου οι Αιγυπτιακές αρχές σεβαστούν τα βασικά θρόνα δικαιώματα. Απαιτούμε οι Ισπανοί και όλα τα κρατημέλη να σταματήσουν να πουλάνε όπλα γιατί τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται για καταστολή της κοινωνίας των πολιτών. Για άλλη μια φορά το παραλαμβάνουμε στο ημικύκλιο. Τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα είναι δυνατόν να κατησχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. πώς Ευχαριστώ η Αμαλφάτη που πρασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο καταδικάστηκε για δύο χρόνια. στη σελίδα της στο facebook ε, περιγράφει τις εμπειρίες που είχε ε, σε επίπεδο σεξουαλικής καταπίεσης ε, και γι' αυτό και συνελήφθη από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Η Αμάλ δεν είναι η μόνη που βρίσκεται στη φυλακή. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους δημοσιογράφους, νομικούς, bloggers, και να σταματήσει τις διώξεις εις βάρος των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ε, τις διώξεις εναντίον μεμονωμένων προσώπων μεταξύ των οποίων και ανηλίκων. Είναι ντροπή αυτό το οποίο κάνει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Σάκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι πολλοί θεωρούν την Αίγυπτο σημαντικό εταίρο στην τρομοκρατία, στη μετανάστευση και για να διασφαλίσουμε σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Και ναι, η Αίγυπτος είναι σημαντική χώρα, γι' αυτό έχει σημασία να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Η καταστολή δεν ε, οδήγησε σε σταθερότητα και νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη των ίδιων πραγμάτων. Έχουμε εξαφανίσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις, καταστολή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και άλλων υπηρεσιτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αυτή η κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι εξαφανίσεις ε, θυμίζουν ε, βεβαίως και έγιναν αντιληπτές στην Ευρώπη με την περίπτωση Τζούλιο Ριτζένι. Θέλαμε λοιπόν να δούμε την κατάσταση διεισόμαση, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάμε στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα όπως θέλαμε. Είναι προβληματικό αυτό και πρέπει να το δούμε γιατί πρέπει να είμαστε σε επαφή για να εκφράσουμε προσωπικά τις ανησυχίες μας για την έλλειψη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ έχω ενδιαφερθεί προσωπικά για τη συγκεκριμένη πρόταση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Αίγυπτος είναι ένας πολιτικός και οικονομικός εταίρος στρατηγικής φύσης. Και δεύτερον, ε, υπάρχει πάντα ανοιχτή υπόθεση στην Αίγυπτο και την Ιταλία του Ρετζένι που δολοφονήθηκε αφού βασανίστηκε το 16 έχει ξεκινήσει μια διαδικασία θεσμικών αλλαγών στην Αίγυπτο και εμείς θέλουμε να σταθούμε φίλοι στην Αίγυπτο και στο λαό της έτσι ώστε να συνοδεύσουμε αυτές τις θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία έκφρασης όπως επίσης και η ελευθερία του συνέρχεστε και η ελεύθερη πολιτική έκφραση. Αυτά χαρακτηρίζουν τις ε, ε, προοδευμένες πλουραλιστικές χώρες και αυτά θα αποτρέψουν τους πολέμους και τις συγκρούσεις. Η δημοκρατία δεν είναι σίγουρα τέλεια, αλλά δίνει εγγυήσει ε, για ειρήνη και ασφάλεια. Και εμείς ζητάμε λοιπόν την αλήθεια από τους Αιγυπτίους για τον Ρετζένι, ο οποίος αγαπούσε τη χώρα, ερευνούσε τη χώρα αυτή και δεν το κάνουμε αυτό για πολιτικούς λόγους, θέλουμε το τι συνέβη ε, στη ζωή αυτού του νέου ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων τώρα. Σβόμποντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Αίγυπτο δυστυχώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σοβαρές. Εκατοντάδες ε, φυλακίζονται μόνο και μόνο γιατί θέλουν να είναι ελεύθεροι, θέλουν να εκφράζονται ελεύθεροι. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καν δικαστεί ή δικάζονται κάτω από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι σωστές. Θέλουμε όλοι αυτοί λοιπόν να απελευθερωθούν. Οι Αιγύπτιοι δεν προστατεύουν και τους χριστιανούς, ενώ είναι το 10% του πληθυσμού και υφίστανται συστηματικά επιθέσεις των φανατικών μουσουλμάνων. Δυστυχώς η Αίγυπτος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών όπου η ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης είναι περιορισμένη. και το 17 δολοφονήθηκαν 17 χριστιανοί στο λοφορείο. Εμείς, σε πάση περιπτώσει, θέλουμε καλές σχέσεις. Κύριε Σβόμποντα, θα δεχθείτε μια, μια μπλε κάρτα. Μια μπλε κάρτα. Σε ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ποιον κατηγορείτε εσείς ε, για τον πόλεμο κατά των Ισλαμιστών. Την κυβέρνηση που πολεμά τους Ισλαμιστές, ε, ε, ποιος διώκει τους χριστιανούς τελικά. Μην τα μπερδεύουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ναι, το, γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό που λέτε. Γι' αυτό ακριβώς είπα πως η κυβέρνηση της χώρας πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία των ε, χριστιανών ε, αφού υπάρχουν αυτοί οι φανατικοί. Σας ευχαριστώ κύριος Πιεραντόνια Παντσέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Αίγυπτο δημιουργήθηκε η Ανώτατη Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό ακούγεται καλό. Αποτελείται από εκπροσώπους της κυβέρνησης, η οποία ελέγχει τις υπηρεσίες ασφαλείας που κατηγορούνται για παραβιάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρητικά η χώρα αυτή, η οργάνωση αυτή μάλλον, η επιτροπή αυτή προστατεύει περισσότερο σε επίπεδο διπλωματικό την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό παρά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ευρωπαϊκή Realpolitik ε, δυστυχώς επηρεάζεται από τα εμπορικά συμφέροντα. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζονται τα θρησκευτικά δικαιώματα. Δυστυχώς στην Αίγυπτο υπάρχουν πάρα πολλοί ακτιβιστές νομικοί που έχουν καταδικαστεί για τις ιδέες τους. Υπάρχουν μαζικές δίκες που οδηγούν σε εκτελέσεις, χωρίς αποδείξεις. Και υπάρχουν και δύο γονείς, οι γονείς του Σεύτζιο Ρετζένη, που εξακολουθούν να θέλουν να μάθουν γιατί βασανίστηκε, γιατί δολοφονήθηκε και γιατί αποκρύβουν την αλήθεια οι Αιγυπτιακές αρχές. Είναι κατεπίγουσα η δράση για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με δύναμη και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ για το ECR. Ο Βίστησεν. Σας ευχαριστώ. Και πάλι συζητάμε την κατάσταση στην Αίγυπτο και παρά το ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις ανησυχητικές πρέπει να θυμόμαστε όταν μιλάμε για κοινοβούλιο και κομισιόν δεν ξέρω τι έχουμε κάνει εμείς ε, ήμασταν υπέρ της Αραβικής Άνοιξης αλλά οι συνέπειε ε, ήταν δραματικές και οπωσδήποτε μια αποσταθεροποιημένη Αιγύπτος δεν μας συμφέρει. Τότε είναι πολύ μονομερές αυτό το ψήσιμο. Μπορούμε και άλλες χώρες να κατηγορήσουμε για τα ίδια πράγματα. Πρέπει να αφήσουμε τους Αιγύπτιους να επιδείξουν κάποια πρόοδο, αντί να προσπαθούμε συνεχώς να τους ε, κατηγορούμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ για την ε, γκουε, κυρία Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αίγυπτος οπωσδήποτε είναι μια χώρα στη γειτονιά μας. Έχουμε πολλούς αιώνες κοινή ιστορίας και από το 2009 η κατάσταση επιδεινώθηκε. Πρέπει να είμαστε σαφείς για το ότι συμβαίνει, υπάρχουν συμφωνίες ε, με την ε, Αίγυπτο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια στη σημαντική παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, στο όνομα κάποιων κοινών συμφερόντων. Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί των ελευθεριών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ατιμορρησία για αυτά τα ζητήματα. Ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε άλλο. Καλές ή καλές σχέσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τις καταγγελίες ε, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Και για το συμφέρον ε, του Αιγυπτιακού λαού. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσει με την Αίγυπτο. Η χώρα συνεχίζει να δολοφονεί αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα είπαμε και στην υπατή εκπρόσωπο στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου. Το ψήφισμά μας είναι έκκληση, κάτι επίγουσα. Να σταματήσει η πώληση υλικού ασφαλείας, τεχνολογίας κλπ. Κάθε στρατιωτική βοήθεια να πάυσει. Τα έχουμε πει. Συνεχίζεται όμως. Συνεχίζουμε να δίνουμε όπλα, τάγκς, μέσα βασανισμού του λαού και κυρίως των αγωνιστών δικαιωμάτων. Και η Ισπανία έκλεισε συμφωνία όπλων πάνω από 100 εκατομμύρια γύρω στο 17. Και τι θα γίνει. Και έχουμε τους αγωνιστές, έχουμε τον κόσμο που δολοφονείται με βόμβες ισπανικές θα πρέπει να σταματήσει αυτό το εμπόριο αίματος που στρέφεται κατά του Αιγυπτιακού λαού και έτσι καταπατάται κάθε ανθρωπινό δικαίωμα και το διεθνές δίκαιο. EFTD. Φάμπιο Καστάλ. Συνάδελφε, πέρασαν τρία χρόνια από τη βάναυση τηλεφωνία του Ρετζένια Μα πώς να σκέφτεται τώρα κάθε μέρα η οικογένεια, τι, αισθάνονται. Συνεχίζει να μην υπάρχει ε, απονομή δικαιοσύνης. Και πέραν των ε, διασφαλίσεων για τις δήλωση καλών προθέσεων συνεχίζουν να μην συνεργάζονται οι Αιγύπτιοι. Ε, ε της ατιμορρησίας. Συνεχίζω με τις επαφές ούτως ώστε να στείλουμε αυτό το μήνυμα στο ότι δεν ξεχνούμε. Ούτε ξεχνούμε ότι θα ξεχάσουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε γεωπολιτικός παίκτη, να επηρεάζουμε τα τεκτενόμενα στον κόσμο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται κάποιες απαντήσεις όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα εις βάρος κάποιου Ευρωπαίου που έχει τόσο βάναυσα βασανιστεί και δολοφονηθεί. Θα πρέπει να αναζητηθεί η αλήθεια. Αν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαμε τις απαντήσεις. Δεν είναι δυνατόν να κατησχεί η νοοτροπία της Realpolitik. Να υπάρξει ρήξη των σχέσεων μας με τη χώρα μέχρι ότου πριτανεύσει η δικαιοσύνη και η ελευθερία για τον Τζούλιο Ρετζένη. E Ο κύριος Λεμπρετόν για το ΕΝΕΦ. E Εφτά ομιλητές ε, έχουν ε, ξεσηκωθεί εναντίον της Αιγύπτου και όμως ο, ο Σίση καταπολεμά τον Ισλαμισμό. Ανέτρεψε το 16 τον Μόρση, τον Ισλαμιστή που οδηγούσε την Αίγυπτο στο χάος και πέρυσι εξελέγει στην, Προεδρία της Δημοκρατίας και καταπολεμά τον Ισλαμισμό και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε ιδεολογικό επίπεδο λέγει ότι θα πρέπει να ανανεωθεί το Ισλάμ και να καταδικαστούν οι σκοταδιστικές μορφές του. Λοιπόν, αντί να τον κατηγορούμε, πρέπει να τον στηρίξουμε. Γιατί αν πέσει το καθεστώς, τότε τα 90 εκατομμύρια των Αιγυπτίων θα γίνουν φανατικοί Ισλαμιστές και θα ενισχύσουν την τρομοκρατία. Η τραγωδία του Στρασβούργου πρέπει να μας οδηγήσει να σταθούμε πιο ρεαλιστές. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους και όχι να δίνουμε μαθήματα ηθικής στους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έτμαν. έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι. Ε, Τακτικέ ειδήσει για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Αιγυπτό με ανησυχούν. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα και τα θεμέλια της δημοκρατίας κινδυνεύουν. Οι πολιτικοί αντίπαλοι συλλαμβάνονται και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να τονίσω πως η Αίγυπτος είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στις ε, ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και είναι και παράγον σταθερότητας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να απομακρύνεται συνεχώς η Αίγυπτος από τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για δεύτερη φορά φέτος Χτυπάμε το καμπανάκι. Για την Αίγυπτο. Οι αρχές ε, πρέπει να σταματήσουν την καταστολή των των δικαιωμάτων που μυστηριωδώς εξαφανίζονται. Πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος ο Αμάλ Ισμαήλ Χασάν. Ζητά από όλα τα κράτη-μέλη να μιλήσουν με μια φωνή στο Συμβούλιο Σύνδεσης για να ασκηθεί πίεση στον πρόεδρο Αλσίση πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Αίγυπτο, αλλά όχι εάν συνεχίζουν να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εγγύηση για το κράτος δικαίου και τον πολιτικό πλουραλισμό. Εάν η Αίγυπτος θέλει πέρα από γείτονα να γίνει και εταίρος τη Ένωση, ένας τρόπος υπάρχει για να σημειωθεί συγκεκριμένη πρόοδο ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιούρεκ τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Προχτές στους δρόμους του Στρασβούργου είχαμε πάλι τραγικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο του πολέμου των Ισλαμιστών κατά των εθνών της Ευρώπης. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Αίγυπτο. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου πολεμά το Ισλαμικό κράτος ε, στη χερσόνησο του Σινά και προσπαθεί να σταματήσει τις ε, επιθέσεις τους κόπτες. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή μάχεται για την διεθνή ειρήνη. Κάθε κυβέρνηση κάνει λάθη. Αντιλαμβάνομαι και τους συναδέλφους από την Ιταλία που θέλουν εξηγήσει από την κυβέρνηση της Αιγύπτου για την περίπτωση Τζούλιο Ρετζένη. Αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε και την κυβέρνηση της χώρας αυτής για τον αγώνα που δίνει. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Τον κύριο Φρουντζουλίκα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Πράγματι. Πρέπει να δούμε την κατάσταση κάπως πιο ισορροπημένα. Αφενό δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αρχές Αιγύπτου κτλ. Από την άλλη συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της και κτλ. Αλλά εδώ, μια που έχουμε και μια επιτροπή ανάπτυξης, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει ένα μοχλό που έχει, γιατί του δίνουμε πολλά λεφτά για έργα κτλ. Ε, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Γιατί δίνουμε και λεφτά, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί στην Τανζανία ε, και παραβιάζουν μετά τις ε, ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Φρουντσουλίκα, δεν υπήρξε κάποια ερώτηση. Ε. Αυτό ήταν μια δήλωση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο στις διμερείς μας σχέσεις διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει πράγματι να μιλήσει για την κατάσταση εκεί όπου απαιτείται στο ζητήματα δημοσίας τάξης αλλά ε, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό είναι ότι δεν μιλάμε για τους ξεκάθαρους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα για το Χαλιφάτο, το Ισλαμικό κράτος Η προηγούμενη κυβέρνηση Μόση προς τα εκεί πήγαινε. Σας ευχαριστώ, ο κ. Σαφχάουζερ. Η τρομοκρατική απόπειρα στο Στρασβούργο την Τρίτη μας δείχνει ότι στην πολιτική πρέπει να διαλέγουμε τους φίλους και τους εχθρούς. Ε, ο εντοπισμός του εχθρού ε, νομίζω είναι βασική αποστολή ενός πολιτικού ηγέτη όπως ε, το έκανε και ο Winston Churchill. Ο στρατάρχης Σίσης στην Αίγυπτο κατανοεί τον κίνδυνο του Ισλαμισμού. Η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Αλατζάρ στο Κάιρο το 2015 ήταν ε, πραγματικά εξαιρετική. Ο πρόεδρος Σίση μουσουλμάνος θέλει να εγγράψει τους αδελφούς μουσουλμάνους στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων οι εχθρικές προτάσεις ε, των φιλελευθέρων, των σοσιαλιστών και των κομμουνιστών εναντίον της Αιγύπτου δεν στηρίζουν αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει. Πιστεύετε ότι το ριζοσπαστικό Ισλάμ σέβεται καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς υποστηρίζετε τους εχθρούς και φυσικά θα προκαλέσετε εμφύλιο πόλεμο γιατί ο Ισλαμισμός είναι ήδη εδώ Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε τις παρεμβάσεις. Περνάμε στη διαδικασία Catch Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Η Αίγυπτος είναι μια πανέμορφη χώρα είναι πάρα πολύ κοντά στο νότο της Ευρώπης και έχει σημειώσει και σημαντικό πρόοδο σε διάφορου τομείς. Δυστυχώς όμως, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες σκοτεινές πλευρές στην Αίγυπτο, ιδιαίτερα σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις άδικες μορφές ε, ε, φυλάκισης πρέπει τα θέματα αυτά να μην τα αγνοήσουμε και νομίζω ότι θα, αν πιέσουμε θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πριν μερικά χρόνια και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από την Ιρλανδία είχαμε κάνει μια έκθεση για τον Ιμπραήμ Χαλάουι, ένα Ιρλανδό πολίτη ο οποίος ήταν φυλακισμένος στην Αίγυπτο και χάρη στις προσπάθειες τις οποίες κάναμε απελευθερώθηκε. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν τις Αιγυπτιακές αρχές έτσι ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γουόρντα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο χειροτερεύει συνεχώς. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση εξαρτάται από θανατικές καταδίκες και άσκηση βίας. Ο κόσμος υφίσταται τα βασανιστήρια και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται. Υπάρχουν καταχρήσεις και εις βάρος ανηλίκων ε, όπως λέει το Human Rights Watch, στις χίλιες περιπτώσεις που δικάστηκαν στα στρατιωτικά δικαστήρια από το 2015 και μετά, 114 περιπτώσεις αφορούσαν ανηλίκων. Ιδιαίτερα και παιδιά με αναπηρίες δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν. Είναι μια χώρα που δεν φροντίζει τους νέους της. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος οι προτεραιότητες για τις σχέσεις 17-21 υιοθετήθηκαν πέρυσι. Έχουμε την δυνατότητα να πιέσουμε την Αιγυπτιακή κυβέρνηση να αναλάβει δράση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σλάιν έχει το λόγο. Εδώ και 35 μήνες ζητάμε και εξακολουθούμε να ζητάμε την αλήθεια για τον ε, Σέρτζο Ρετζένη. Ε, θα πρέπει με το ψήφισμα αυτό να απαιτήσουμε την πλήρη συνεργασία των Αιγυπτιακών αρχών με τις Ιταλικές αρχές, όπως επίσης και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των νομικών και των ερευνητών από Ιταλία και Αίγυπτο. Πρέπει να σταματήσουν τα βυσανιστήρια και οι απαγωγές στην Αίγυπτο πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα ο Αμαλφατή χωρίς καμία καθυστέρηση και το ίδιο ισχύει και για όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι σε καμία χώρα δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε την Αίγυπτο ως ασφαλή χώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε ε, να πουλάμε όπλα στο καθεστώς του Αλσίση γιατί πολλές κυβερνήσεις το κάνουν προωθώντας μόνο τα εμπορικά συμφέροντα. Και δεν πρέπει εμείς να παραβιάζουμε τις ίδιες μας τις ιδρυτικές αρχές. Ζητάμε λοιπόν την αλήθεια για ό,τι συνέβη στον Σέργιο Ρετζένι. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο. Ο κύριος Μίμητσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράγματι κάθε συμφέρον να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Αίγυπτο. Είμαστε πεπισμένοι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί εφόσον όμως γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ε, το εγγυάται. Το Σύνταγμα του 2014 και οι ανηλυμένες υποχρεώσεις μέσω των διεθνών συμβάσεων της Αιγύπτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει την Αίγυπτο να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. και στον ψηφιακό κόσμο και γενικότερα θα πρέπει να σεβαστούμε το ανθρώπινο δίκαιο ε, όπως το προβλέπει και το Αιγυπτιακό Σύνταγμα επαναλαμβάνω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Κοινωνία των Πολιτών λειτουργούν διαδραστικά και προσπαθούν να επηρεάσουν την κατάσταση στην Αίγυπτο για τους ε, προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αιτίε ε, κατηγορίας οι πιο συχνές εις βάρος αυτών των προασπιστών είναι η διάδοση ψευδών ειδήσεων και η χρήση ε, ε, χρηματοδοτούμενων από το εξωτερικό μέσων. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει ε, τελικά. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει και παλαιότερα. Η κυρία Μογκερίνη έχει κάνει τον Μάιο του 2018 δημόσιες δηλώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ανήσυχη επίσης και από αυτά τα οποία ακούμε στον τομέα της, ε, των βασανισμών και των ε, κακών συνθήκων κράτησης, των βασανιστήριων κτλ. Απαιτείται λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πιέσουμε την Αιγυπτιακή κυβέρνηση στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανακοίνωση η οποία έγινε ε, για την ε, συγκεκριμένη Επιτροπή για τον Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί, αλλά θα πρέπει να τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή. Οι δραστηριότητες των ΜΚΟ θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται να διεξάγονται χωρίς περιορισμούς ζητάμε από την Αίγυπτο να ξεκινήσει ένα πλήρη διάλογο με την κοινωνία των πολιτών της χώρας στα πλαίσια των δυνατοτήτων που δίδει ο νόμος. Η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας με την Αίγυπτο ήδη την επόμενη εβδομάδα θα μας δώσει τη δυνατότητα να το συζητήσουμε το θέμα αυτό για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση περατώθηκε. Έχουμε 7 σχέδια ψηφίσματος επ' αυτού. Πράσινη, ECR, EFDD, GUE, Σοσιαλιστές, ΑΝΤΕ και ΕΛΚ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αργότερα. Επόμενο σημείο της ημέρα διατάξης, η Τανζανία. Οργανώθηκε η συζήτηση παρομοίως. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους συντάκτες του ψηφίσματο, την κυρία Σαρτζεντίνη, που είναι η πρώτη που θα μιλήσει. Έχετε το λόγο, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το 2015 ήμουν εισηγήτρια για την αποστολή παρατηρητών στην Ταζανία και εκλογές που έφεραν τον πρόεδρο Μαγκαφούλη στην εξουσία. Λοιπόν, και τελικά είχαμε ένα νέο υποψήφιο από το κυβερνών κόμμα και αυτό είναι ευχάριστο, διότι βλέπουμε ότι κάπως αλλάζει η κατάσταση. Υπάρχει άλλος υποψήφιος. Οι εκλογές εξελίχθηκαν αρκετά ομαλά. Υπήρξαν κάποια προβλήματα σε κάποιες ε, περιοχές, αλλά ουσιαστικά τα πράγματα πήγαν καλά, έγινε εκστρατεία κατά της διαφθοράς και η Τανζανία αναγνωρίζεται σαν χώρα η ειρηνική περιοχή ειρήνης σε αυτή την περιοχή του κόσμου είναι μια περιοχή η οποία έχει περάσει πολλά. Υπήρξαν ε, πολλές δύσκολες περίοδοι, αλλά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα, διότι ε, υπάρχουν απειλές κατά της αντιπολίτευσης, σημειώθηκαν κάποιοι θάνατοι και γίνεται ένα κυνήγι μαγισσών όσον αφορά τους ΛΟΑΔΜ. Και είχαμε και λιντσαρίσματα ε, διότι δεν ήταν ετεροφιλόφιλα άτομα. Και ο πρόεδρος Μαγκαφούλη εμποδίζει εγγύου, έγκυα κορίτσια από το να πηγαίνουν στο σχολείο. Και τα προγράμματα κατά της διαφθοράς έχουν παγώσει πια. Και πήγαμε από μια χώρα που ήταν σταθερή, έχουμε μια χώρα που επικρατεί μεγάλη αστάθεια και αναταραχή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προσπαθεί να κάνει κάτι για την κατάσταση. Ε, επέστρεψε, ανε, ανεκλήθη ο πρόεδρο τη εκεί αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και διακόπησαν οι σχέσει. Κατανοώ αυτά που μα είπε η κυρία Μογκερίνη, καταλαβαίνω πολύ καλά. Α, θα πρέπει να δώσουμε υποστήριξη στη δημοκρατική αντιπολίτευση. Πρέπει να δει η αντιπολίτευση ότι έχει κάποια υποστήριξη και ότι δεν είναι μόνη της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Σαρτζεντίνη. Η κυρία Κριστίν Βεργιά έχει το λόγο. Ε, μετά από την άφηξη στην εξουσία του Τζον Μαγκουφούλη. Το 2015 επιδεινώθηκε η κατάσταση στην Τανζανία και από την αρχή του έτους ακόμα χειρότερα. Μπλόγκερ, αντιπολιτευόμενοι, προσπιστέ δικαιωμάτων μπορούν να συλληφθούν. Το 20 Φεβρουαρίου ο κ. Ζωφρέ Λουένα, βουλευτής του Βασικού Κόμματος Αντιπολιτεύσεως, σκοτώθηκε με μαχαίρι ε, και έξι κανάλια και δύο σταθμοί ραδιοφωνικοί έχουν διακόψει εκπομπέ. Το Μάρτιο έχουμε νέο νόμο επικοινωνιών και δημιουργεί προβλήματα στα ΜΜΕ και χρειάζεται να πληρώνει 900 ευρώ φόρο και ειδική άδεια. Και είναι υπερβολικό το ποσό που ζητείται για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ε, τελικά υπάρχει μια έλλειψη τάξη δημόσιας και έχουμε νόμο για την ε, κυβερνοασφάλεια, η ομοφιλοφιλία, ε, κατημορείται με 30 χρόνια μέχρι σόβια φυλακή. Και στον Τάραλ Σαλάμ η κυβέρνηση τοπική απείλησε να λιθοβολεί όσους είναι ομοφιλόφιλοι ή μάλλον να τους κάνει ε, θεραπεία για να αλλάξουν. Οι νέες ε, ε, περνάνε από καταναγκαστικό γάμο και υπάρχει διάκριση εναντίον τους άμα είναι έγκυος. Και δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός, κυρίως στην περιοχή του Σερενγκέτη. Έχει βλαφτεί ο τουρισμός από όλα αυτά. Θα μπορούσε να είναι ευλογία ο τουρισμός. Λοιπόν, και έχουμε και αρπαγή γεών και κερδοσκοπία όσον αφορά τη γη. Και στρέφεται αυτή κατά τον Μασάη έχουν ε, διάφορες μπουλντόζες που καταστρέφουν ε, περισσότερα πράγματα από αυτά που οικοδομούν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, η κυρία Σοράγια Πόστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς είναι θλιβερό και πρέπει να θυμίσουμε τις αρχές και την κυβέρνηση της Τανζανίας ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυβέρνηση Τανζανία υπέχει υποχρέωση να προστατεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών τη χώρα. Ζητώ, απαιτώ να ακυρώσει του νόμου που ποινικοποιούν την ομοφιλοφιλία και να σταματήσει η σύλληψη και η βία κατά των μελών των ΛΟΑΔΜ και θα πρέπει ε, να προστατευτούν και ακτιβιστές των δικαιωμάτων. Απαιτούμε η κυβέρνηση Τανζανίας αμελητή να ακυρώσει τον νόμο που απαγορεύει τις, τα έγκυα κορίτσια από το να πηγαίνουν στο σχολείο. Και κορίτσια που έχουν γεννήσει θα πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και θα πρέπει να γίνεται σεβαστό πανταχού σε όλη την Ιφίλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απευθύνω Απευθύνω κράτη-μέλη για μια ακόμη φορά να βοηθήσουν τρίτε χώρε όπω η Τανζανία να προστατεύσουν του υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινότητα ΛΟΑΔΜΑ, να αποποινικοποιηθεί η σεξουαλικότητα, που είναι ποινικοποιημένη σε πολλέ ε, χώρε ε, του κόσμου. Η επιδείνωση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τανζανία εμποδίζει την ανάπτυξη, την ευημερία, την ειρήνη και την ασφάλεια τη χώρα και πράγματι και τι καλέ ε, σχέσει τη με όλε τι άλλε χώρε μεταξύ αυτών και τη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα οι περιορισμοί στον τύπο να αρθούν, να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια για όλου του πολίτε. Ο αποκλεισμό των εγγύων κοριτσιών, μητέρων από τα σχολεία είναι κάτι άκρο ανησυχητικό και οπισθοδρομικό. Είναι νέα κορίτσια που έχουν δικαίωμα σε ποιοτική εκπαίδευση. Είναι σημαντικό η Τανζανία να πάψει άμεσα αυτήν την απαγόρευση. Στηρίζω την ε, Επίτροπο Μογκερίνη στην προσπάθεια που κάνει να ε, βάλει τάξη και λογική σε αυτή την κατάσταση και σε αυτόν τον παραλογισμό. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρο. Τώρα, εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει η κυρία Βαλενθιάνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Δεν είναι απλά μια συζήτηση, αλλά μια καταγγελία για τη σοβαρή επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρατηρείται στην Τανζανία. Επιδείνωση που είναι ορατή από όλους εμάς που έχουμε μια ευαισθησία για την προστασία των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και απέναντι σε αυτή την επιδεινούμενη ε, κατάσταση ε, και πραγματικά το κυνήγι, τη δίωξη στην κοινότητα ΛΟΑΔΜΑ. Αυτό που ζητούμε εμείς, τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι άμεσα να επανεξετάσει τις σχέσεις ε, της Ένωσης με την Τανζανία και να απαιτήσει αλλαγή της κατασταλτικής νομοθεσίας. Η νομοθεσία της χώρας είναι υποβαθμιστική. Ε, απέναντι ιδίω πιο ευάλωτε ομάδε, γκέι, λεσβείε, τρανσέξουαλ, αλλά και γυναίκε, παιδιά. Απαιτούμε λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ, απαιτούμε από το Συμβούλιο να ε, δει υπό αυτό το οπτικό πρίσμα τη σχέση με την Τανζάνη. Σεβασμό στα ανθρωπίνα δικαιώματα, σεβασμό στι μειονότητε, σεβασμό σε όλου ε, του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αλλιώ θα πρέπει οι σχέσει με τη χώρα αυτή να διακοπούν. Ευχαριστώ πολύ. Ιγνάσιο Κοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η καταστατική πολιτική του Τζον Μαγκουφούλη κάνει γιγάντια βήματα προς ναζισμό και τώρα τα, είναι επίθεση κατά τον γκέι που πραγματοποιείται. Ο Πολ Μακοντάγκο, κυβερνήτης του Ντάρελ Σαλάμ, θέλει ε, να απαλλάξει την κοινωνία κατά του κακού της ε, δύσεως που επηρεάζει αρνητικά τους κατοίκους της Ανζανίας, κυρίως ε, λόγω τη ομοφιλοφιλίας. Λοιπόν, σε εξοξοβική αυτή ε, η προπαγάνδα τη κυβερνήσεω και δημιουργήθηκε και task force για να εντοπίζει και να συλλαμβάνει τα μέλη τη κοινότητα των ΛΟΑΔΜ. Σαν δεν έφτανε αυτό, ο πρόεδρο Μαγκουφούλη απαγόρευσε την στο σχολείο των ε, κοριτσιών που είναι μητέρε. Ε, και είναι κάτι που εμποδίζει να έχουν παιδεία και εκπαίδευση και τι εμποδίζει αυτέ τι καημένε να μπουν και στην αγορά εργασία. Και γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ανησυχού, μας ανησυχούν οι δράσεις αυτού του Προέδρου και του κυβερνήτη που παίρνει τις εντολές από το Θείο. Λοιπόν, αυτά είναι βήματα που ταιριάζουν τον πολιτισμό. Είναι παρά, παράλογη προσέγγιση. Πρέπει να επανεξετάσουμε τον δεχόμενο αναστολή της σχέση με την Τανζανία μέχρι ότου να τεθεί θέμα σε αυτή την ε, απαράδεκτη ε, καταδίωξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντέιβιντ Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα η κατάσταση είναι απελπιστική. Για πολλές δεκαετίες η Τανζανία φαίνεται ε, να πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση και ε, την εκλογή του Προέδρου Μαγκαφού το 2015 την καλωσορίσαμε ε, γιατί είπε ότι θα μειώσει τη διαφθορά, θα βελτιώσει την οικονομία. Όμως αντί να καταστέλει τη διαφθορά, καταστέλει οποιονδήποτε ασκή κριτική στην εξουσία του. Παρανοχλούνται και διώκονται και κρατούνται δημοσιογράφοι, τίθενται επιτίθεται το κράτο και απειλεί ε, πολιτικούς και σε μια περίπτωση είχαμε και δολοφονία. Διεθνεί οργανισμοί επίσης δεν είναι στο απειρόβλητο. Ένας πρέσβη επίση ανακλήθη και ε, πραγματικά παρατηρούμε και η κοινότητα των λάδων να διώκεται και πραγματικά δεν γίνεται τίποτα στο κράτος για να τους προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους. Πολλά χρόνια έλεγα ότι πρέπει να έχουμε πιο στενές σχέσεις με την Τανζανία, αλλά πλέον να συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι πρέπει να επαναξετάσουμε τη σχέση μας με τη χώρα αυτή. Κυρία Νίνα Τζιλ, ευχαριστώ. Και εγώ θα προσθέσω τη δική μου φωνή στις ανησυχίες των συναδέλφων για την επιδείνωση κατάσταση των δικαιωμάτων στην Τανζανία όχι μόνο η κυβέρνηση, ο πρόεδρος ε, Μαγκοφούλη συγκεκριμένα καταστέλει τα μέσα μέσα και σε όπως ακούσαμε, αλλά κάτι πιο ανησυχητικό παραβιάζει και τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων, ε, και τις έγκυες ε, νέες γυναίκες δεν τους αφήνει να πάνε σχολείο. Επίσης, ο Επίτροπος Μακόντα επίλησε να διώξει στην Τάρη Σαλάμ τους γκέι άντρες. Αυτό είναι αποκρουστικό, ανήκουστο. Οι σχέσεις μας ε, με την Τανζανία πρέπει να πανεξεταστούν από την Κομισιόν, ε, γιατί εδώ μιλάμε για βασικές μας αρχές, ε, ιδίω την ανάκληση, μετά την ανάκληση και του πρέσβη το Line Denmark έκανε κάποια πράγματα και ακούσαμε και τι είπε ο πρέσβης. Ε, ε, ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Και ένα πιο ευρύ θέμα τώρα που με απασχολεί είναι η πολιτική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που φαίνεται ότι θα έπρεπε να μην είναι τόσο ε, αποτρεπτική στον προσανατολισμό της, αλλά προεξοφλητική, να βλέπει από πριν τι συμβαίνει. Τι βήματα παίρνουμε επίσης για την χάραξη και του διεθνούς δικαίου. Περνάμε τώρα στη δικασία προσέλκυσης της προσοχής του Πρόεδρου Πόσπης, είναι ο πρώτος ομιλητής. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Μαγκουφούλη είναι μεγάλη απογοήτευση για μας. Ε, να μέναμε να μεταρρυθμίσει τη χώρα, να καταπολεμήσει την ε, διαφθορά και αντί αυτού διαπιστάνουμε πόλεμο κατά των ε, διαφόρων σεξουαλικών μειονοτήτων. Μεταξύ αυτών και γυναικών και κοριτσιών. Πώς θα αντιδράσει λοιπόν η Κομισιόν. Νομίζω πως αυτή, την κατάσταση θα πρέπει, αυτή η κομισιον νομιζω πως αυτη κατασταση θα πρέπει να αλλάξει ε, και να αλλάξει τη σχέση μας ε, μεταξύ Ένωσης ε, και Τανζανίας. Δεν θα πρέπει με απλές δηλώσεις καταδίκης να περιμένουμε ότι κάτι θα γίνει. Ας αναλάβουμε οικονομική δράση κατά της χώρας αυτής και διπλωματική πίεση θα πρέπει να ασκηθεί ε, ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ η κυρία Τζούλι Ward. Ε, έχω φρίξει από αυτή την κατάσταση στην Τανζανία. Οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών και οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχονται καθημερινέ επιθέσει. Τον περασμένο μήνα οι αρχές ζήτησαν από το κόσμο να καταγγέλει οποιονδήποτε είναι ύποπτο ότι είναι γκέι και μάλιστα ε, το ζήτησαν να μην τους ε, ακουμπούν καν. Ε, πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές λόγω της, του σεξουαλικού προσανατολισμού, πραγματικού ή ε, εικονικού. Η κυβέρνηση προφανώς και παροτρύνει τη βία και την ξενοφοβία, ενώ ο σεβασμός όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καθήκον της Τανζανίας δεν θα πρέπει να, ε, να παροτρύνει τη βία κατά οποιασδήποτε μειονότητα. Εγώ ε, ε, στηρίζω την ανάκληση του πρέσβη μας τον Ταρεσαλάμ ώστε να αναθεωρήσουμε την κατάσταση αλλά και τη σχέση μας με την χώρα αυτή. Στην περασμένη εβδομάδα στο Μπενίν, στην κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση ΕΟΚ, Ένωσης μάλλον και ρώτησα τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση χωρίς να πάρω καμία καμιά απάντηση. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Τανζανία είναι εκτός ελέγχου. Παρατηρούμε ότι ο πρόεδρος Μαγκαφούλη πλέον διώκει την αντιπολίτευση, ε, τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, τα κόμματα με τα οποία δεν συμφωνεί έχει θέσει εκτός λειτουργίας ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες. από εκεί και πέρα αυτό που κάνει είναι να ασκεί και μια πολιτική η οποία επί της ουσίας ενθαρρύνει τη σεξουαλική βία. έχουμε αποκλεισμό των εγγύων γυναικών και κοριτσιών από τα σχολεία γεγονός απαράδεκτο. και παρατηρούμε επίσης ότι ε, στην περιοχή της γης των μασάι πλέον γίνεται μια αρπαγή των γεών γέες οι οποίες είναι αρρώσιμες αρπάζονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς. είναι προφανές ότι η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα κατά της κυβέρνησης της τανζανίας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μασιμό Καστάλτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στον Τάρελ Σαλάμ η ομοφιλοφιλία δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα και με αυτά τα ντροπιαστικά λόγια το περασμένο Οκτώβριο ο Πάολ Μακοντά, ο κυβερνήτης της περιοχής, ε, ε, ξεκίνησε ένα πραγματικό κυνηγητό των ομοφιλόφιλων. Στιγματίζει αυτούς τους ανθρώπους ε, για το ότι αμαρτάνουν κατά της φύσης. Πολύ καιρό έχουμε ανεχτεί αυτή την κατάσταση στη μια χώρα όπου οι άνθρωποι, ε, οι ομοφιλόφιλοι τιμωρούνται με 30 χρόνια κάθριξης. Όμως δεν είναι μόνο οι ομοφιλόφιλοι στο στόχαστρο. Από την εκλογή του Μαγκουφούλη έχει υπάρξει τεράστια επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τρελή απαγόρευση των κοριτσιών ε, μητέρων να επανέλθουν στα θρανία. Αυτοί, αυτές οι νέες που συχνά είναι θύματα βίας πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο, στην, ε, στην ε, εκπαίδευσή τους και το παιδί τους. Ε, παρακαλώ να ζητήσουμε να αρθεί αυτός ο παράλογος νόμος, όπως και οι άλλοι νόμοι κατά των κοινότητα των LGBTI. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα τι πολιτικέ μα απέναντι στη Τανζανία. Α ε, ισχύσει η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντό του Κοτονού, εντό άλλων συμφωνιών που έχουμε ε, υπογράψει. Διαφορετικά μένουν μόνο παλιόχαρτα αυτέ τι συμφωνίε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο e- Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι ανέκαθεν κατά τέτοιου είδου ψηφισμάτων που προετοιμάζει το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και θα πρέπει να κάνει, να περνάει νομοθεσίε και να λύσει τα προβλήματα των λαών τη Ευρώπη και όχι να προσπαθεί να διορθώσει τα πάντα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε φτιάξει, φτιάχνουμε τρία ψηφίσματα ανασύνοδο, δηλαδή πάνω από 300 ψηφίσματα κάθε χρόνο, ασχολούμαστε με οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, αλλά τελικά δεν εξυπηρετεί αυτό κανένα σκοπό. Απολύτως. Κανένας δεν διαβάζει εκτός από τους ίδιους τους ευρωβουλευτές. Οπότε είναι σπατάλη χρόνου και προκαλεί μόνο ε, έκπληξη. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει καν ε, τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ούτε που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρουν. Βασικά λοιπόν ε, είναι παράλογο το ότι ασχολούμαστε με αυτή την κατάσταση. Ε, ασχολούμαστε δίθεν με την κατάσταση των γυναικών, των LGBTI. Ο κόσμος ε, εκπλήσεται με αυτές μας τις ενέργειες. Ο κύριος Κέλλη. Μάλιστα κύριε Κέλλη, έχετε μια ερώτηση με γαλάζια κάρτα, μπορείτε να την υποβάλλετε. Μάλιστα, πώς μπορεί ο κύριος λέει, να λέει, ο συνάδελφος να λέει ότι σπαταλάμε το χρόνο μας, ενώ όταν τόνισα και στη συζήτηση για την Αίγυπτο, έχουμε ένα ψήφισμα εδώ και μετά από αυτό, αυτό το ψήφισμά μας και την πίεση από την Κομισιόν και την Ιρλανδική κυβέρνηση, οι Αιγύπτιοι συμφώνησαν να τον απελευθερώσουν. Σας ευχαριστώ. Αλλά αυτή είναι μια πολύ απλοϊκή ε, εικόνα για τη διεθνή πολιτική. Δεν μπορεί να ασκεί κανείς τη διεθνή πολιτική γράφοντας ε, ψηφίσματα. Εντάξει, λειτουργήσε μια φορά, αλλά πιστεύετε πως ο κόσμος στην Ταζανία ε, θα αντιδράσει. Έχουν αυτή την πολιτική και τους ενδιαφέρει η δική μας αντίδραση. Ούτε καν μας υπολογίζουν. Βεβαίως μπορεί πάντοτε κανείς να ασκήσει πίεση. Όμως, ε, ε, όσο λιγότερο μιλά κανείς για το πρόβλημα, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι να δράσουμε δηλαδή με τρόπο που να πιάσει εξαπίνη στον εχθρό. Να είναι στοχευμένες οι δράσεις μας δηλαδή. Ε, πρέπει να, να δυσκολέψουμε αυτόν τον οποίο θέλουμε να πιέσουμε. Εν γέννη πιστεύω πως αυτή η πολιτική δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Κύριε Σούσνιες, δεχόσαστε άλλη μια γαλάζια κάρτα. Από ε, την κυρία Χιμένες, ναι. Θέλω να σας ζητήσω αν έχετε αδερφές ή κόρες, έχετε μητέρα. Δεν σας ενδιαφέρει τι γίνεται εκεί στις γυναίκες. Εμένα με ενδιαφέρει. Το ίδιο και τους περισσότερους που είμαστε εδώ. Και αυτό που λέτε εσείς, ότι δεν αλλάζει τίποτα, δεν είναι αλήθεια. Εγώ σας εγγυώμαι. Έχω πολλούς φίλους σε Βενεζουέλα που είναι εξόριστοι, που δέχονται απειλέ, που είναι φυλακισμένοι και μου λένε σας παρακαλούμε μη σιωπήσετε, μη σιωπήσετε εσείς γιατί θα πρέπει κάθε υπόθεση να την υπερασπίζετε με μεγάφωνο. Εμείς αυτό είμαστε εδώ, το μεγάφωνο αυτών που δεν έχουν φωνή. Τους δίνουμε εμείς τη φωνή μας. Ε, γιατί γι' αυτό μας έχουν εκλέξει οι πολίτες μας, για να μιλούμε εξ ονόματός τους και να υπορασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ για 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολύ προσωπικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Ρωτήσατε κατά πόσο έχω παιδιά. Έχω παιδιά. Αλλά αυτό αφορά την ιδιωτική μου ζωή. Παρακαλώ να μην ρωτάτε πράγματα που αφορούν την ιδιωτική μου ζωή. Και ναι, βέβαια, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Και ναι, και πάντα μπορεί να πει κανεί ότι αν πει κανεί κάτι, κάτι μπορεί να αλλάξει. Τι περισσότερε στιγμέ όμω δεν αλλάζει τίποτα. Κυρίω εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παράγει τόσο μεγάλο αριθμό ψηφισμάτων. Ίσως αν είχαμε ε, παράγει λιγότερα ψηφίσματα, τότε θα είχαμε μεγαλύτερα αποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά είναι τόσα πολλά τα ψηφίσματα, δεν μπορεί να προλάβει ο κόσμος να καταλάβει αυτά που λέμε. Ευχαριστώ, κύριε Πολτσακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακούγοντας τον συνάδελφο Σόσνιετς, πρέπει να πω ότι ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα μου έλειπε ο κύριος Κόλμπιν Μίκε. Ε, είναι αυτό θλιβερή ανακάλυψη για μένα σήμερα το πρωί. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε για την Τανζανία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι που υποφέρουν. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφου που περιέγραψαν την κατάσταση στη Τανζανία. Είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτο μια κυβέρνηση την οποία είχαμε εμπιστευτεί και είχαμε θρέψει ελπίδες για αυτήν. Μπροστά στα μάτια μας αυτή η κυβέρνηση να μεταμορφώνεται σε ένα καθεστώς που καταπιέζει, καταστέλει την αντιπολίτευση, την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ, κάνει κατασχέσεις ιδιοκτησίας των πολιτών. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να αναφέρουμε. Αυτό δεν είναι κάτι άχρηστο κύριε Σόσνιετς. Αυτά χρειάζεται να υποθούν ε, και έχουμε τρόπους ε, να δράσουμε. Και αυτό ε, σας είπε ο κύριος Κέλλη. Τώρα εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί κατά της ε, κυβερνήσεω της ε, Τανζανίας και να πει σαφώς ότι δεν μπορεί να την υποστηρίζουμε πια. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα δώσω το λόγο στον κύριο Σόσνιετς. Λυπούμε. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Επιτρόπο γιατί δεν ήμουν εδώ από την αρχή της συζήτησης. Ε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν έξι ταυτόχρονες ε, άλλες υποχρεώσεις ε, επιτροπές. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή Έλεγχου του Προϋπολογισμού, Έχουμε επίσης και έναν προπαρασκευαστικό διάλογο και ταυτόχρονα και την Ολομέλεια και άλλα τέσσερα, τρία πράγματα δεν μπορούμε να είμαι πανταχού παρών. Πιστεύω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τανζανία, το capacity building, δηλαδή η δημιουργία, η βελτίωση των υποδομών είναι κάτι που είναι σημαντικό, αλλά ας το κάνουμε και εδώ πρώτα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί ε, συνάδελφοι θα ήθελα να να είναι εδώ για να συζητήσουμε και να δούμε τι γίνεται με την αναπτυξιακή πολιτική, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τη συνεργασία και σε ό,τι αφορά τις ε, ψηφοφορίες, επειδή θα ξεκινήσουν όπου να είναι, παρακαλώ Πρόεδρε να ξέρετε ότι πρέπει να κλείσετε στη μία τις ψηφοφορίες, γιατί πρέπει να είμαστε και στις πατρίδες μας για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή και να συζητήσουμε με τους ε, συμπολίτες μας. Θέλουμε να τους εξηγήσουμε ε, και να τους ε, κάνουμε να καταλάβουμε τι κάνουμε εμείς για αυτούς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Πολύ σύντομα. Την Τρίτη το ξαναθέσατε αυτό το θέμα, κύριε Ρούμπιχ, και το μήνυμα το έχω ε, διαβιβάσει. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε πιο γνωριά για να ολοκληρώσουμε και νωρίτερα και ξέρω ότι υπάρχουν ταυτόχρονα άλλες συνεδριάσεις, επιτροπών και, και άλλες. Και έχω ζητήσει και από το Προεδρείο και από τη διάσκεψη των Προέδρων και άλλα ε, όπω όπως είναι η διάσκεψη των Βέλων των Επιτροπών να μην οργανώνουν ταυτόχρονα ψηφοφορίες κυρίω, αλλά και συνεδρία επιτροπών εν γέννη ταυτόχρονα με την ε, Ολομέλεια εδώ στο Στρασβούργο και ελπίζω να ληφθούν τα σχετικά μέτρα. Τώρα εξ ονόμας της Ευρωπαϊκής να ακούσουμε τι έχει να πει ο επίτροπο κ. Μίμητσα. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Για σειρά δεκαετιών η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτής απόλαυσαν στενές και καρποφόρες σχέσεις με την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας και ήταν βασικό εταίρο αναπτυξιακό η Ευρωπαϊκή Ένωση και από του σημαντικού εταίρου για το εμπόριο και τι επενδύσει. Αυτή η συνεργασία ε, ρίζωνε σε κοινέ θεμελιώδεις αξίες, όπω ήταν η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και με κοινή συμμετοχή στην πρόθεση της ειρήνης, αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και περιφερειακή ολοκλήρωση. Όμως, τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε συρρήκνωση του δημοσίου χώρου στην Τανζανία μέσω απειλών, παρενόχλησης, δίωξης και αύξηση των περιορισμών όσον αφορά τη δραστηριότητα των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών, των ΛΟΑΔΜΕ, των κοινωνικών ΛΟΑΔΜΕ, των μέσων ενημέρωσης και πολλών πολιτικών κομμάτων. Ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου επανειλημμένα υπονομεύθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ανησυχίε δημοσία το Σεπτέμβριο και αυτό μέσω δηλώσεως στην 31η Σύνοδο των του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη. Και επαναλάβαμε αυτά τα στοιχεία μέσω δηλώση είπα τη εκπροσώπου τη κ. Φεντερίκα Μογκερίνη, που εκφράστηκε εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ενώσεω και δημοσιεύθηκε αυτό το έγγραφο στι 15 Νοεμβρίου. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, οδήγησε σε αυξανόμενη πίεση από από τις αρχές της Τανζανίας για να υποχρεωθεί ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωση να αποχωρήσει από την Τανζανία. Και τελικά οδηγηθήκαμε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να τον ανακαλέσουμε στα, στο κέντρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαβουλεύσεις. Αυτή είναι μια στάση άνευ που δεν ευθυγραμμίζεται με τον μακροχρόνιο διάλογο που είχε καθιδρυθεί με την Τανζανία. Σε αυτή τη φάση, μαζί με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διεξαγάγει μια συνολική αναθεώρηση των πολιτικών και σχέσεων ε, με την Τανζανία. Ε, αυτή η αναθεώρηση θα συμπεριλαμβάνει επίσης θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και την αναπτυξιακή μας συνεργασία. Όπως υπογραμμίστηκε στην δήλωση της 15ης Νοεμβρίου, είναι σημαντικό να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Τανζανία διατηρώντας τις επαφές με φορείς από όλε τις σφαίρες πολιτικών, οικονομικών, πολιτικών κύκλων, την κοινωνία των πολιτών επίσης. Ο διαθρωμένος πολιτικός διάλογος με την κυβέρνηση της Τανζανίας θα επαναληφθεί από τη στιγμή που η αναθεώρηση της σχέσεως έχει ολοκληρωθεί εν ώψη αποκαταστάσεως των δεσμών μας επί μιας πιο σταθερής ε, και μελλοντοστραφούς σχέσεως. Α δούμε τώρα και το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με την Αφρική. Το, στα τον Νοέμβριο του 2017 συμφωνήσαμε σε, πάνω σε μια ατζέντα, σε ένα πρόγραμμα κοινών συμφερόντων, κοινών αξιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θα εξετάζει τις σχέσεις με κάθε αφρικανικό εταίρο με ένα σφαιρικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά μας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη σε καλές σχέσεις με σταθερές δημοκρατικές ε, κυβερνήσεις όπως θέλουμε να είναι στην Τανζανία που θα συμμετέχει αυτή η κυβέρνηση Τανζανία στην όλη διαδικασία της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε. Έλαβα έξι σχέδια ψηφισμάτων. Εκ μέρους των διαφόρων πολιτικών ομάδων περατώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αργότερα. Η πρώτη ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί σε 40 λεπτά. Καλά τα μαντάτα. Στις 12 και 40 θα τελειώσουμε και μπορούμε αυτό να το εγγυηθούμε διότι ο υπεύθυνο θα είναι ο κύριος Βίλαντ ο οποίος πολύ συχνά έχει ε, επενεθεί για τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεων. Αυτά είναι τα καλά μαντάτα. Θα τα πούμε λοιπόν σε 25 λεπτά. Μείον 30 δευτερόλεπτα, λέει πρόεδρος. Κύριε Ζούμπιχ, έχετε κάτι διαδικαστικό το οποίο θέλετε να αναφέρετε αποφασίστηκε στο Προεδρείο σε ό,τι αφορά τη συντάξεις των βουλευτών να μπει ε, μια ηλικία 65 έτη και υπάρχουν δαπάνες 5% παραπάνω ε, πλέον. Θα ήθελα να πω ε, και να γραφεί στα πρακτικά ότι στην Επιτροπή Προπολογισμών ήμουν εισηγητή ε, για το προπολογισμό τη Ένωση και στράφηκα κατά αυτή τη απόφαση ε, και θα γίνει καταγγελία και στο δικαστήριο, διότι δεν είναι σύμφωνο ο κανονισμό αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ και θέλω να γραφεί στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα το διαβιβάσω αυτό. Θα κάνω τα δέοντα πρέπει να διακόψουμε μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 12. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Herr Kollege Lambert hat uns Wort. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. ο κύριος Λάμπερτς ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας... Ε, ησυχία! Ναι. Κάποιοι κάνουν πολύ θόρυβο. Λοιπόν, λάβαμε όλοι, αγαπητέ Πρόεδρε, ένα δέμα πριν από κάποιες εβδομάδες από μια αμερικανική μάρκα εταιρεία που λέγεται Facebook. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό το δέσμα ε, χαρτιού και πλαστικού αποτελεί ε, σπατάλη ενέργειας ε, διαπιστώνω πως η Αμερικανική εταιρεία μας στέλνει υλικό διαφημιστικό για να μας ε, κάνει να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες της ε, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε στη διάρκεια της, της επίσκεψης του Προέδρου της Μάρκ Τζούκερμπερκ εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και επιμένω ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις η εταιρεία αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμπερτς. Νομίζω ότι είναι ε, δυνατό και η αποστολή πίσω στην εταιρεία του δέματος αυτού, αλλά αυτά που είπατε εσείς νομίζω ήταν πάρα πολύ με την έκθεση και της κυρίας ε, Παρακαλώ. Α, ο κύριος Καβαντά θέλει το λόγο. Je serai πάρα πολύ σύντομο. Στηρίζω αυτό που ο κ. Λάμπερτ. Και να σα πω ότι παρά οποιαδήποτε χρήση σε τριμερή διάλογο, που δεν έχει καμία σχέση να γίνεται lobbying, πριν από τρει εβδομάδε, αφού ψηφίσαμε στην Ολομέλεια το κείμενο για το copyright, τρει εβδομάδε μόλι μετά το YouTube, η Google και κάποιοι άλλοι ήταν εδώ στις ε, εγκαταστάσει του Ευρωπαϊκού και συγκεκριμένα στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματο του Και αυτό δεν τον τιμά ε, ούτε τον ίδιο την ομάδα του για να μα κάνουν να αλλάξουμε άποψη. Κύριε Πρόεδρε, να γραφτούν στα πρακτικά ε, τα αιτήματά μα. Δηλαδή, να απαγορεύεται ε, στις διοργανικές φάσεις και μετά την Ολομέλεια να είναι κοντά ε, λιγότερο ή περισσότερο σε εμά ε, οι λομπίστε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Καβαντά. Όπως είπα, όμως τώρα θα περάσουμε ε, στην, στην απόφαση για την ΟΝΕ. Ο κύριος Γκίγκολ θέλει να μιλήσει για αυτό το θέμα. Έχετε δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αξιολογήσαμε προσεκτικότατα το σχέδιο διαπραγματικής θέσης του Κοινοβουλίου. Ακούσαμε και τη δήλωση του Προέδρου της ΕΚΟΝ. Όμως είμαστε πεπισμένοι ότι το σχέδιο διαπραγματευτικής θέσεως του Κοινοβουλίου δεν είναι αρκετά καλή. Δεν αρκεί να, να ελέγξουμε τους κινδύνους των ευρωπαϊκών τραπεζών και να αποφύγουμε την χρέωση των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων και να το εκμεταλλεύονται οι Τα κόκκινα δάνεια είναι περισσότερα τώρα από ό,τι ποτέ πριν από την οικονομική κρίση. Οι νέοι κανόνες όμως για την κάλυψη των κόκκινων δανείων θα ισχύει για νέα δάνεια και μόνο για αυτή τη μερική λύση η θέση του Ευρωκοινοβουλίου είναι πιο δύναμη από αυτή του Συμβουλίου και από αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελάχιστες απαιτήσει για παροχή πιστώσεων για κόκκινα δάνεια είναι κάτι απαραίτητο. Έτσι οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να διασώζουν προβληματικές ε, τράπεζες στην επόμενη οικονομική κρίση. Αυτοί που θέλουν πιο ανίσχυρους κανόνες για αυτά τα δάνεια διατέχουν τον κίνδυνο η Τραπεζική Ένωση να μην ολοκληρωθεί. Έτσι δε χειρότερο. Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για την αγορά πιστώσεων. Αυτό σημαίνει ότι Blackstone, BlackRock και άλλες αγορές και άλλοι αγοραστές πιστώσεων μπορεί να διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους αυτοί που είναι χρεωμένοι να διώκονται τα σπίτια τους. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν αρκεί αυτή η διαπραγματευτική θέση. Και ζητάμε από τους ε, συναδέλφους να ζητήσουν επιτροπή να ξανασχεδιάσει τη διαπραγματευτική θέση για να έχουμε καλύτερη προστασία των καταναλωτών και να έχουμε στεναρότερου κανόνες για τι τραπεζέ μα. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη για να μιλήσει για την απόφαση αυτή. Έχετε και εσείς δύο λεπτά στη θέση σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που λέει ο συνάδελφος Γκίγκολ δεν είναι σωστό, δεν αληθεύει. Είναι ισορροπημένο συμβιβασμό. Ταυτόσιμο ουσιαστικά με την ομόφωνα ψηφισμένη θέση του Συμβουλίου. Και είναι κάτι ευπρόσδεκτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό εξασφαλίζει πολύ συνετή προσήγγιση για τα κόκκινα δάνεια, αποφεύγοντας τον κίνδυνο άκαμπτων διατάξεων αυτών που ζητάτε εσεί. Τέτοιε άκαμπτε διατάξει θα επηρεάσουν αρνητικά καταναλωτέ και μικρομεσαίε επιχειρήσει. Βρίσκω αντιφατικά τα επιχειρήματά σα. Κάντε προπαγάνδα υπέρ των καταναλωτών. Αυτό που θέλετε να κάνετε είναι ακριβώ αυτό που θα φέρει σε δύσκολη θέση, θα φέρει στα χέρια των Αμερικανικών hedge funds εκείνου που έχουν στεγαστικά δάνεια και αυτού που έχουν μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεύτερον, ο λόγος για τον οποίο οι πράσινοι προβάλλουν αντιρρήσεις είναι βασικά πολιτικός διότι εμεί στάσαμε ισορροπημένο συμβιβασμό με το ΕΛ και δεν σα άρεσε. Και είμαι υπερήφανο γι' αυτό. Διότι έχουμε πολλέ αποκλίνουσε απόψει στο ΕΛΚΑ. Είμαι περήφανο διότι στο Κοινοβούλιο καταφέρνουμε να βρίσκουμε και κοινό τόπο και μαζί να θεσπίζουμε καλή νομοθεσία. Αυτό κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη και όχι πιο αδύναμη. Και γι' αυτό πρέπει να εγκρίνουμε αυτό το συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκολτιέρη. Ακούσαμε μία ε, αναφορά υπέρ, μία κατά. Ποιος είναι υπέρ της απόφασης. Κατά της απόφασης. Εγκρίθηκε λοιπόν. Εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο. Επομένω, ε, μπορούμε να περάσουμε στι οργανικέ διαπραγματεύσει. Πηγαίνουμε στην έκθεση ΖΙΦΚΑ, ονομαστικά ε, ειδική πλειοψηφία. Αγαπητείτε εδώ, ονομαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Έγινε δεκτή. Πηγαίνουμε στην έκθεση Σαλήνη. από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή τροπολογίας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 109 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226 ε, ονομαστικά. 226 ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίφθηκε. 2.23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.27 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Για διαδικαστικό. Θα σας στείλουμε ένα τεχνικό. Αλλά προς το παρόν αναζητήστε ένα άλλο μηχάνημα που να λειτουργεί. 225 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρόταση κομισιόν τώρα, ονομαστικά ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίθηκε η έκθεση Θέλει το λόγο εισηγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω την ε, αναβολή προ την Ήτρη για ε, διοργανικέ διαπραγματεύσει σύμφωνα με το 69. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται και πηγαίνουμε στην έκθεση τη συναδέλφου Μλίναρ. Καταρχάς, τροπολογίες της καθήλων αρμόδια επιστοπής μπλοκ υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνονται. 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 74, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. 150 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 203 ονομαστικά ψηφίζουμε, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Απορρίφθηκε. 204 ονομαστικά ψηφίζουμε, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Απερίφθηκε αυτή. 205 άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 202 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Πρόταση Κομισιόν μαστικά. Άρχεται ψηφοφορία ψεφίσατε όλοι. Πέρας. Έγινε δέκτη έκθεση η εισηγήτρια Μλίναρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τη μεγάλη υποστήριξη, συνάδελφοι. Σύμφωνα με το άρθρο 59, θα ήθελα να προτείνω το θέμα να απευθύνει στην Επιτροπή Ήτρε για διοργανικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό το αίτημα. Κλείστε όμως το μικρόφωνο σας πάλι κυρία Μλίναρ. Περνάμε στην έκθεση της συναδέλφου Γκρίφιν, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή έκθεση Γκρίφιν και πηγαίνουμε στην έκθεση του συναδέλφου μας Τάγκ, αρχικά τροπολόγηση καθήλων αρμόδιας του σαν μπλοκ, ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές δεκτές. Τώρα, τροπολογία 2, συνδέεται με τα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6, με τα πρώτο τμήμα, η ψήφη υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 2, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 6, με τα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε τροπολογία 9, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε 14 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε Τρόπο 27 ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 28 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. εγκρίθηκε. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 έως 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 63 να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τις τροπολογίες από 56 ως 58. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. 63 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 54 και 60 ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν για 41 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 55 και 61 ταυτόσιμες. ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 50 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 53 και 59 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 62 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τρόπο 24. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε πρόταση της Κομισιόν συνολικά με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πηγαίνουμε τώρα στην έκθεση Ροζάτη. Καταρχά, τροπολογίε καθήλων αρμόδια Επιτροπή, μαζί όλες οι ψήφοι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 6 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 9 σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, ποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε το πρώτο τμήμα. Τρίτο τμήμα, λέει ο πρόεδρος, ονομαστικά. Ψηφίσαμε, ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 16 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε. τρόπο 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. 32 ψήφι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 33 ψήφι υπέρ, α, όχι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, ονομαστική κλίση έχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 40 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε και πάμε στην πρόταση της Κομισιόν με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Και δεκτή έκθεση. Και τώρα πηγαίνουμε ε, στο ψήσιμο για το Ιράν, αρχική παράγραφος 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14, πρώτο, αρχικό και πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε θέλετε. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Το ψήφισμα συνολικά με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. Πηγαίνουμε στο ψήφισμα για την Αίγυπτο και ιδίω την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοινό ψήφισμα αρχικά, παράγραφος 11 αρχικού κειμένου πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Όχι, συγγνώμη. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17, αρχικό κείμενο. Ψήφι περ. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την παράγραφο 11, το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 17, αρχικό κείμενο. Ψήφι περ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19, αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές ε, δεν είναι σαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Άρχιτε ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίθηκε Recital ε, H ε, ψήφι περ. κατά αποχές δεκτό L ψήφι περ. κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος τώρα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές και εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στο ψήφισμα για την Τανζανία, στο G, το recital, πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, το σύνολο του ψηφίσματος ψήφι υπέρ, κατά αποχές Πηγαίνουμε στην έκθεση της κυρίας Μακλάρκιν, ε, μία ενιαία ψηφοφορία, ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Die Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πηγαίνουμε στα ψηφίσματα σε ό,τι αφορά ε, την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την Ιαπωνία, δύο τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, όχι. Παρακαλώ να με ακολουθείτε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 2. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ψήφι πέρ. Να ελέγξουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίφθηκε τροπολογία 9 ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 4 ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 4 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. το 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ένα τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. οκτώ τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Πηγαίνουμε στο ψήφισμα σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την προστασία του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Δημοκρατία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 2. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά του ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα προχωρούμε στην έκθεση της συναδέλφου Εύη, δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητήου 2017, για 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία να ελέγξουμε την 5 ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε απορρίπτεται τροπολογία 6 πέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία τροπολογία 6 Ψηφίσατε όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. μα σκόντε τα χέρια σας δεν θα έκανα λάθος. Τροπολογία 7 ονομαστικά έρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 13 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14, μονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 21, αρχικό κείμενο ονομαστικά. Ψηφίζουμε άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ονομαστικά την τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της 22 παραγράφου ονομαστικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγρα... Μάλλον τροπολογία 16. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 26. Αρχικό κείμενο ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 33, αρχικό κείμενο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 19D με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ε, μάλλον, συγγνώμη, πέρα ψηφοφορία απορρίφθηκε. Τροπολογία 20D, ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρόπο 21D, ονομαστική κλίση, έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. για 1D, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη X υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι εγκρίνεται εγκρίνεται εγκρίνεται λάθος έκανα λάθος έκανα τρία τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται αρχικό κείμενο στην ετοξιγέψη AC, άρχεται ψηφοφορία ονομαστική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πηγαίνουμε στην έκθεση Βίξτρεμ. Τροπολογία 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά θα χρειαστεί να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 4. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ε, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 9. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 αρχικό κείμενο. Ελέγχουμε την τροπολογία 1 άρχεται ψηφοφορία. Haben alle Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 αρχικό κείμενο σε 4 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά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 Παράγραφος 19 αρχικό κείμενο σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφο 23 αρχικό κείμενο σε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 8 τροπολογία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται αρχικό κείμενο 26 παράγραφος πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος ελέγχουμε.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 Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψήφι περ. Κατά. Πολλές αποχές. Ιδέως ε, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε τελικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν μου επιτρέπετε να ε, πω ότι εδώ ε, πριν ολοκληρώσω τις ψηφοφορίες μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ε, όλους τους συνεργάτες. Είναι η τελευταία ψηφοφορία από το τέλος χρονιάς αυτή για μένα. Dass die alle rechtzeitig nach Hause zu kommen, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Okay όσοι ε, δεν θέλουν να ακούσουν τις ε, επεξηγήσεις ψήφου να ε, εγκαταλείψουν ησύχως την αίθουσα θα παρακαλέσω και να θυμηθούμε τι συνέβη αυτή την εβδομάδα και τον Όλεγκ Σεντσόφ και σεβασμό σε όλους. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία ονομαστικά άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Έγινε δεκτό το ψήφισμα.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 Er, Συνάδελφος ε, Σούλικ ε, έχει ζητήσει το λόγο. oder Frau Herr Kollege Sulik, ist das noch Κύριε Σούλικα, αξιοκολουθείτε να θέλετε το λόγο. Όχι, μάλλον. Επομένως, να περάσουμε τώρα σε επεξηγήσεις ψήφου. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με τις αιτιολογήσεις ψήφου από τις χθεσινές ψηφοφορίες που επειδή κράτησε πολύ οι ώρες ψηφοφορίας δεν ε, ακούσαμε όλες τις αιτιολογικές ε, ε, όλες τις αιτιολογήσεις ψήφου. Μετά θα ακούσουμε αυτές που έγιναν την Τετάρτη στις 5 και μετά θα ακούσουμε τις ε, αιτιολογήσεις ψήφου για τις σημερινές ψηφοφορίες. Άρα έχουμε πολλές αιτιολογήσεις ψήφου. Ε, είναι λογικό, είχαμε και πολλές ψηφοφορίες, αλλά το αργότερα στις 3 παρατέταρτο πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί η αίθουσα για την έναρξη της επόμενης συνόδου Ολομέλειας στις 3 το μεσημέρι και όσοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν ε, τις προφορικές αιτιολογίες θα τις δώσουν γραπτός. Ξεκινούμε λοιπόν με τις αιτιολογήσεις ε, ψήφου Βιώτη Ριούμπιχ ε, για το νέο προϋπολογισμό του 2019 ο συνάδελφος Βιέγας. Έχει το λόγο πρώτος. Δεν είναι εδώ όμως ε, ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, ήταν δύσκολη η διαδικασία η δημοσιονομική φέτος, ιδιαίτερα και γι' αυτό και ευχαριστώ τον κύριο Βιώτη για τη σκληρή του δουλειά. Επίσης συνέβαλα στο σχέδιο προϋπολογισμού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους οργανισμούς της Ένωσης στο τομέα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Δυστυχώς η εντολή έχει επεκταθεί αλλά περιμένουμε πραγματικά οι οργανισμοί να δώσουν περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους. Ε, φαίνεται πως το Συμβούλιο αυτό πιστεύει πάντως. Εγώ όμως ως Ευρωβουλευτής το θεωρώ αυτό απαράδεκτο. 943 εκατομμύρια ευρώ που πετύχαμε στο Κοινοβούλιο αντιστοιχούν στις κύριες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, έρευνα, νέοι, μικρομεσές, ε, κλιματικές αλλαγές, ε, μεταναστευτικό και γι' αυτό το υπερψήφισα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάμικινς. Ο κύριος Χάνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για τον ε, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο ως συνήθως ε, προεδρεύσατε σε αυτήν την ε, συνεδρία της Ολομέλης και να, ευχηθώ σε όλους συναδέλφους και προσωπικό καλά Χριστούγεννα. Τώρα, να σας πω ότι ο γαλλικός προπολογισμός θα κλιμακωθεί πέρα από τον ε, προϋπολογισμό. Ε, τότε μας λέτε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κανόνες και τα λοιπά. Όταν μια ευρωσκεπτιστική κυβέρνηση στην Ιταλία φάνηκε ότι θα παραβίασε τους κανόνες, καταδικάστηκε ε, καθολικά ε, από τις Βρυξέλλες. Το ίδιο θα ισχύσει όταν θα κάνει το ίδιο και ο Μανουέλ Μακρόν. Ευχαριστούμε κύριε Χάναν. Έκθεση Βιώτη Ρούμπιχ, ολοκληρώθηκαν τα σχόλια και επεξηγήσεις ψήφου. Τώρα πάμε στην σύσταση Σίλβα Περέιρα. Ο κύριος Σαμαρζή. Μετά από τη ΣΥΤΑ έχουμε το ΙΖΕΦΤΑ και προστίθεται αυτή στην μακρά, στο μακρύ κατάλογο συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που είναι ζημιογόνες για την Ένωση, για τους πολίτες και για τον πλανήτη. Κάνετε σπουδαίες ομιλίες για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά αυτό δεν σας ενοχλεί διόλου να ψηφίσετε μία, ψηφ... μία συμφωνία η οποία είναι πιο κλιματοκτόνα όλων των εποχών. Ωραία λόγια για τη βιοπικιλότητα, αλλά δεν σας ενοχλεί καθόλου αυτό να, δίνετε τις, ε, να προσφέρετε τις φάλαινες ε, στη σφαγή. Ε, ωραία λόγια, αλλά αυτή η συμφωνία θα χαμηλώσει προς τα κάτω για να εξισώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μεγάλα λόγια και για τη δημοκρατία, αλλά δέχεστε τα εθνικά κοινοβούλια να, να μην έχουν λόγο. Γι' αυτό το λόγο καταψήφισα αυτή τη συμφωνία που είναι υπέρ των πολυεθνικών και όχι υπέρ των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μαρζέ. Επόμενος ε, ο συνάδελφος Ούρμπαν Κρέσπο. Δεν είναι εδώ ο κύριος Ούρμπαν Κρέσπο, η κυρία Αλμπιόλ Γουσμάν. Σε αυτή τη σύνοδο του Ευρωκοινοβουλίου υπερψηφίστηκε η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Όμω θα ήθελα να πω ότι το 99% των πολιτών τη Ευρώπη δεν έχουν ιδέα. Και δεν έχουν ιδέα διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι το θέλησε. Θέλει να διαπραγματεύεται με τα δικαιώματά μα και τον πλανήτη, χωρί κανεί να το ξέρει και κανένα να την αμφισβητεί. Όμω αυτή η συμφωνία μοιάζει πάρα πολύ με το TTIP που διαπραγματευόταν με τη ΣΥΠΑ ή με αυτήν που υπογράφηκε με τον Καναδά. Όλες αυτές οι συμφωνίες όπου οι πολυεθνικές έχουν περισσότερη εξουσία από τα κράτη μέσα από τα δικαστήρια διαιτησίας ε, ε, όπου οι οι κανόνες μας για το περιβάλλον δεν ισχύουν καθόλου εφόσον η Ιαπωνία θα γεμίσει την αγορά μας από παράνομη ξυλία και από παράνομη ε, αλληλεία. Τα μεγάλα ωφέλη πάνε πάντα στους μεγάλους ομίλους και αυτό γίνεται με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των φιλελευθέρων, των σοσιαλδημοκρατών, καθώς και του ΨΟΕ. εμείς από την Ευρωπαϊκή Αριστερά καταψηφίσαμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκούσμαν. Δεν βλέπω τον κύριο Μορέλη, δεν βλέπω και τον κύριο Βιέγας. Επομένω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπενίτο Θηλουάγα. Αυτή η έγκριση αυτής της συμφωνία θα έχει τεράστιες συνέπειες για τους πολίτες. Είναι μια συμφωνία που δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε να τροποποιηθεί στα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό είναι σκανδαλώδε γιατί η διαδικασία ήταν πραγματικά αδιαφανή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια υποτιθέμενη διαφάνεια διαβουλεύθηκε μόνο με το λόμπι των μεγάλων εταιριών. Έτσι καταφέρνουν να επιβάλλουν, όπως έγινε και με τη ΣΕΤΑ, ε, τον αρνητικό κατάλογο για τις υπηρεσίες δεν, ερωτού, δεν αδιερωτώνται για δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγεία, οι μεταφορές ή η ανάθεση των διαφόρων εργασιών στο, δημοτικό επίπεδο. Αυτό αυτή είναι μια αβάσταχτη μείωση της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων των εργατικών και της δυνατότητας καταπολέμησης της, της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας. Γι' αυτό και δεν το δεχόμαστε. Ευχαριστούμε κύριε Μπέντο Θελουάγα. Ακολουθεί ο συνάδελφος Χάναν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με υπέρ μια συμφωνία ελευθεροπορίου Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ιαπωνία υπέρ του ελευθεροπορίου και όσο πιο είναι πληρέστερη η συμφωνία, τόσο καλύτερο για όλε τι πλευρέ. Σα καλώ όμω να σκεφτείτε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο διαφορετικών αρχιπελάγων, των δύο νησιωτικών μοναρχιών στα δύο άκρα της Ευρασίας και το διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζονται ως εταίροι εμπορικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι κανένας διατείνεται ότι στις στι συνομιλίε Ευρωπαϊκή της Ιαπωνίας ότι ένα μήνα η νήσι Χόνσου, ε, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να παραμείνουν υπό του κανονισμού του Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ούτε κάποιο δεν ότι η εμπορική συμφωνία θα συνδέεται με την ελεύθερη διακίνηση και εκτό αν δεν άκουγα προσεκτικά, δεν είπε κανεί ότι η Ιαπωνία θα πρέπει να παραμείνει σε μια τελωνιακή ένωση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη σύναψη τέτοια εμπορική συμφωνία. Εν αυτή τη ενία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο όχι προσπαθώντα να βρει μια αμοιβαία επωφελή λύση, αλλά με ένα βαθμό ε, αντεκδίκηση. Σε τέτοιο βαθμό που καθιστά μια συνθήκη σχεδόν ανέφικτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χάναν για την ε, έκθεση αυτή τελευταία ο κύριος Μπούτι Κόφερ. Κύριε Πρόεδρε, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ιαπωνία δεν είναι τέλεια. Οι τροπολογίες της δικής μου πολιτικής ομάδας δείχνουν ακριβώς που θα έπρεπε να είχαν υπάρξει βελτιώσεις. Αλλά κατά την άποψή μου ε, το γεγονός ότι τελικά ε, δεν ε, έχουμε καταλήξει σε μια καλή συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και να την απορρίψουμε εντελώ. Υπάρχουν ε, θετικά και αρνητικά σίγουρα. Υπάρχουν εμπορικοί, οικονομικοί λόγοι που πρέπει να αναφερθούν, και νομίζω ότι κυρίως οι στρατηγική λόγοι είναι σημαντική, δηλαδή η προάσπιση του πολυμερού συστήματος σε μια εποχή που έχουμε πιέσει από δύο υπερδυνάμεις ε, και είναι ε, λόγοι για να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση εξού και την υπερψήφισα εγώ προσωπικά και από ε, λόγους αφοσίωσης προς την πολιτική μου ομάδα εκεί που άλλοι ψήφισαν κατά εγώ απήχα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η έκθεση Σίλβα Περέρα και πηγαίνουμε στι εκθέσεις για την μάλλον στην έκθεση ε, για την οικονομική συμφωνισμό και εταιρική σχέση. Πάλι Περέρα. Δεν βλέπω τον κύριο Φλακ, δεν βλέπω τον κύριο Κέλλη, κύριο Άντερσον. Εν γέννη και σε ελεγγύη με την Ιαπωνία και το λόγο τη Ιαπωνία καλωσορίζω αυτή τη συμφωνία. Είναι ένα βήμα προ καλύτερη και πιο δίκαιη εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώση που δίνει προτεραιότητα στα ρυθμιστικά πρότυπα για το περιβάλλον και άλλα βασικά θέματα που έχουν σημασία για του πολίτε. Όμω εξακολουθώ να έχω κάποιε ανησυχίε και γι' αυτό στο τέλο απήχα από την τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα και τη συμφωνία. Καταρχά, δεν υπάρχουν διευθετήσει σωστέ για την παρακολούθηση του αντιχτύπου που υπάρχει για την ασφάλιση των σιδηροδρόμων σε σχέση με τι πρακτικέ εφαρμογέ και υλοποίηση του ανοίγματο των διαδικασιών ε, ε, διαγωνισμών για του σιδηροδρόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Θα έπρεπε να αποκλείεται εκ των προτέρων με συμφωνία προστασία των επενδυτών μέσω ε, διευθετήσεως των διαφορών μέσω διεθνούς δικαστηρίου. Ε, είναι κάτι αντιδημοκρατικό και δεν ενδείκνυται σαν λύση. Παρομοίω, η συμφωνία θα πρέπει πιο συγκεκριμένε διατάξει που θα προβλέπουν την προστασία για το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν νομοθεσία και να ρυθμίζουν και διαφυλάσσοντας κατά τη εμπορευματικοποίηση ε, του ύδατο και άλλων ε, κοινοφελών υπηρεσιών. ευχαριστώ πολύ ολοκληρώσαμε ε, την ε, έκθεση κ. Περέρα. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Πέτρελ, έχουμε μία ε, αιτιολόγηση ψήφου από την κυρία... Τον... Όχι, από τον κύριο Πέτρελε. Δεν είναι εδώ. Όχι. Δεν ήταν Πέτρελε. Λάθος κάνω, λέει ο πρόεδρος. Πέτρελε είναι εισηγητής. Πόσπισιλ είναι ο ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο λέει, για αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο το θέμα, σημαντικότατη έκθεση. Χαίρομαι που ενεκρίθη το κείμενο στην αρχική φιλόδοξη μορφή του. Διότι με την Ιαπωνία δεν πρέπει να έχουμε απλώ εμπορικέ και επιχειρηματικέ σχέσει. Δεν πρέπει να είναι αυτή η χώρα μόνο εμπορικό εταίρο, αλλά είναι μια βασική ασιατική δημοκρατία. Είναι μια ισχυρή οικονομία και στον παρόντα κόσμο που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του 21ου αιώνα όπως είναι η τρομοκρατία και άλλα παγκόσμια προβλήματα, οι ισχυρές οικονομίες θα πρέπει να συνεργάζονται. Όχι μόνο σχετικά με τις εμπορικές ε, σχέσεις, αλλά σε άλλου τομεί. Ελπίζω αυτή η συμφωνία να ενισχύσει έτσι περαιτέρω τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία. Όχι μόνο στον επιχειρηματικό τομέα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πέτερλε λέει ο πρόεδρος. Και πηγαίνουμε τώρα στην έκθεση του συναδέλφου Νίκα για το Horizon Europe. Η πρώτη ομιλήτρια κυρία Νταμάτο που λέει το μάτι και έχει δύο λεπτά κιόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ συχνά ο τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία είναι αυτή η τομή στου οποίου ε, εφαρμόζονται μειοπικέ πολιτικέ. Εμεί θεωρούμε ότι είναι επιταρχική σημασία για το μέλλον των πολιτών. Ε, για να έχουμε κέντρα τεχνογνωσίας και θα πρέπει να έχουμε στέρεα βάση για τις επιχειρήσεις για να μπορούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις πιο μεγάλες ε, προκλήσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι αναγκαίο να έχουμε 120 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα Horizon ε, Europe που θα υποστηρίξει την έρευνα και την κοινοτομία. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πέρα από την αναγκαιότητα να υπάρχει μεγαλύτερη συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα θέλαμε να διατηρηθεί ένα εργαλείο που θα έχει προορισμό την αυξανόμενη έρευνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα ειδικό προπολογισμό που θα συνοδεύει και άλλες ευκαιρίες που θα δίνονται για την ε, ρηξικέλευτη έρευνα. Όσον αφορά τον, τη ρήπανση των πόρων θέλουμε να έχουμε δέσμευση για τον προπολογισμό, για να, για να αντιταχθούμε στην αλλαγή του κλίματο, να έχουμε καλύτερη ενεργειακή απόδοση, να διευκολύνουμε τοπικέ πρωτοβουλίε για αυτοπαραγωγή και κατανάλωση. Το κείμενο θα μπορούσε να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι καρπό μια πολύ δύσκολη συζήτηση και με κάποιου που καμιά στιγμή ήθελαν να ικανοποιήσουν τι ωρέξει των μεγάλων λόμπι παρά να ανταποκριθούν στι αντικειμενικέ ανάγκε τη κοινωνία αλλά έχουμε μια θέση συμβιβαστική, η οποία ανταποκρίνεται και σε απαιτήσει εκείνων που εκπροσωπούν συμφερόντων και λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε των ανθρώπων. Τέλο, και αν θέλουμε βέβαια να επαγρυπνούμε και στο μέλλον, διότι αυτή η αρχή τη καινοτομία, όπω αποκαλείται, δεν θα πρέπει να στραφεί κατά των πολύ μικρών και μικρομεσών επιχειρήσεων και των πολιτών. Και είναι θετική η ψήφο μα. Είναι θετική, διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η αλλαγή περνά και μέσω τη υποστηρίξεω τομέων που είναι τόσο σημαντική, όπω είναι η έρευνα και η καινοτομία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ανταμάτο Η κυρία Σπυράκη δεν τη βλέπω, οπότε ο κύριος Μάμικινς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η επιστημονική έρευνα μας βοήθησε να ικανοποιήσουμε συναδέλφους, να ανταποκριθούμε σε προτεραιότητές τους, να προωθήσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ε, τεχνογνωσία και αριστεία ε, συνοδεύτηκαν, συνόδεψαν αυτά τα προγράμματα ε, για τη γνώση. Γι' αυτό στηρίζω την έκθεση αυτή για το Horizon ε, Europe που παγιώνει την έρευνα στον ευρωπαϊκό χώρο και θα προωθήσει και νέα projects. Ως σοσιαλιστής δημοκράτης υπερασπίζω την αρχή της ανοιχτής επιστήμης και πιστεύω πως η διάδοση της καινοτομίας ε, είναι ε, απαραίτητη. Όμως ε, πρέπει να εγγυηθούμε πως οι επιστήμονες μας θα παραμείνουν στην Ευρώπη γιατί χώρες όπως είπα ο Καναδάς και η Αυστραλία φαίνεται να προσελκύουν τους ερευνητές λόγω των καλύτερων κοινωνικών συνθήκων και των περισσότερων πόρων που δίνουν στην έρευνα. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις κοινωνικές μας συνθήκες εδώ στην Ευρώπη και τους πόρους που αφιερώνουμε στην έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνουμε τώρα στην επόμενη έκθεση, ολοκληρώσαμε την έκθεση του κύριου ε, Νίκα. Ε, είναι η επόμενη έκθεση, δεν βλέπω τον κύριο Γκρτζίπ, άρα πηγαίνουμε στην έκθεση Χολμάιρ Στίβενς ε, για τα πορίσματα και συστάσεις της Επιτροπής για την κυρία Μάκοβε έχει καταρχά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε και να εξηχνιάζουμε με αποτελεσματικό τρόπο την τρομοκρατία. Πρέπει να δώσουμε ερευνητικέ ε, εξουσίες στην Ευρωπόλ, ούτως ώστε να αποφεύγεται η τρομοκρατία, η κυβερνοτρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος κλπ. Ε, η Europol είναι ειδικευμένο φορέα για την καταπολέμηση τρομοκρατία, αλλά μπορεί να στηρίξει τα κράτη-μέλη μόνο κατόπιν αιτήματο. Και κάποια κράτη-μέλη δεν ζητούν αυτό και κάνουν ανάλυση, μπορεί να κάνει ανάλυση δεδομένων, δεν μπορεί να πραγματοποιεί έρευνε. Η τρομοκρατία και η χρηματοδότηση τρομοκρατία είναι διασυνοριακό έγκλημα. Γι' αυτό ένα ενίο φορέα, ένα ευρωπαϊκό φορέα όπω η Europol θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικότερο για την εξυχνίαση που πραγματοποιείται από ότι τα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Και καλύτερο αυτό παρά η ποινική συνεργασία μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών. Οι ερευνητικέ εξουσίε θα πρέπει να συνοδεύονται από μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη της Europol. Θα πρέπει αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε όμως την τρομοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Μακοβέη. Δεν βλέπω τον κύριο και εδώ. Ο κύριος Μάκιμιν, ε, Μάμικιν, συγγνώμη, ξανά. Ευχαριστώ. Τα κράτη αντιμετωπίζουν αυξανόμενη βία ακροδεξιού τύπου. Ε, το η άφηξη μεταναστών, προσφύγων και εθνοτικές ε, ε, μειονότητες ε, δέχονται επιθέσεις και στη χώρα μου τη Λετωνία έχουμε το, τα ίδια φαινόμενα. Θα πρέπει η πρόσφατη επίθεση εδώ στο Στρασβούργο να μας θυμίσει πως ο κίνδυνος υπάρχει πάντοτε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να, να εντοπίσουμε ε, και να, τέτοιου είδους περιστατικά και να αντιδράσουμε γρήγορα όταν αυτό χρειάζεται. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιου είδους προκλήσεις ε, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και γι' αυτό και η απάντησή μας θα πρέπει να είναι διασυνοριακή και γι' αυτό και ε, είναι πρόσδεκτο το αίτημα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου να, να εργαστεί περισσότερο σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αρμόδιους οργανισμούς και επίσης είναι πρόσδεκτα οποιαδήποτε άλλα μέτρα προτείνει η Κομισιόν. Ευχαριστούμε συνάδελφέ Μαμίκινς. Ο κύριος Ξύπη δεν είναι, ο κύριος Νέκοφ δεν λείπει, η κυρία Βόζεμπεργκ επίσης, οπότε έτσι τελειώνουν οι επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Χολμάγερ Στίβεν. Τώρα έχουμε την έκθεση Μακάλιστερ, ετήσια έκθεση για την εκτέλεση της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Η κυρία Μακοβέη, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. μεγαλύτερες απειλές στην ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι η προπαγάνδα του Κρεμλίνου και η ρωσική προπαγάνδα που θέλει να αποδιερθρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που δεν υπακούν στην ε, ρωσική, στις ρωσικές εντολές. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε όμως να γίνει αν δεν υπήρχαν και σύμμαχοι, συνένοχοι χώρες μέλη. Εάν θέλουμε να σταματήσουμε την καταστροφική δράση της Ρωσίας στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης, θα πρέπει να καταργήσουμε τον κανόνα της ομοφωνίας. Ψευδείς ειδήσει διαδίδονται όταν γίνεται λόγος για τις διαμαρτυρίες στη Γαλλία, το Βέλγιο και τις κατοχώρες. χώρες και χρειάζεται ισχυρή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράνομες προσαρτήσεις, κρίση προσφυγικό, ε, είναι αυτά όλα απειλές που φοβίζουν όλο, όλα τα κράτη-μέλη και ο Πούτιν ε, είναι υπέρμαχος του διέρευε και βασίλευε. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν βλέπω ούτε τον κύριο Κρέσπο, ούτε τον κύριο Πιοτρόφσκι, ούτε την κυρία Σουίτσα. Οπότε τελείωσε. να επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Μακάλιστερ. Ούτε για την έκθεση Πάσκου είναι εδώ ο κύριος Πιοτρόφσκι. Οπότε περνάμε στην έκθεση Αουστρεβίτσιους 2017 Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον λόγο έχει ο κύριος Σκρίπεκ. Δεν είναι εδώ. Σκρίπεκ, όχι. Δεν θα μας ε, εξηγήσετε. Καλώς. Πώς πισίλ. Σας ευχαριστώ. Εγώ στήριξα την έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι έχει ένα πολύ καλό επίπεδο. Είναι πολύ καλύτερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Εγώ είμαι δικηγόρος και η αποστολή μου είναι να απαγορεύσω την θανατική ποινή παγκοσμίω. Βλέπουμε ότι οι θανατικές ποινές ε, έχουν πέσει κατά 7-8% αλλά δεν αρκεί αυτό. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει στο θέμα και να μην υποτιμά το θέμα αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε την χρήση της θανατικής ποινής. Εγώ στήριξα την έκθεση και ελπίζω να υπάρξει κάποια βελτίωση του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πόσπισιλ. Οπότε τώρα έχουμε την κυρία Σαμπόρσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δυστυχώς, όπως έχει ξανασυμβεί πολλές φορές σε αυτή τη θητεία, ακόμα και αυτή η ετήσια εκθέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα έδωσε μια στρεβλωμένη εικόνα για το πώς έχει η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύσουμε και έχουμε ένα σωρό προτάσεις για αυτό το κείμενο. Αλλά αυτά δεν εμπίπτουν στις αρμοδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με τις συνθήκες και εμένα με εντυπωσίωση ότι στην έκθεση περιλαμβάνεται ακόμα και κάποιες αρχές που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Κάποιες αρχές που καθιλώνται στον ΟΗΕ. Και επομένως αυτό το έγγραφο το οποίο έχουν επικαλεστεί δεν το χορηγεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. όλα αυτά είναι παραπλανητικά. Όλες αυτές οι ιδέες ε, αποπροσανατολίζουν Γι' αυτό και εγώ δεν μπορούσα να ψηφίσω την έκθεση. Σα ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Ο κύριο Σόσνιερ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι χειραγωγείται η πολιτική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτω ώστε να υπάρχει κάποια ανατροπή των ηθών παγκοσμίω έχει γίνει όργανο προπαγάνδας. Ε, καταπιέζονται οι σεξουαλικές μειονότητες. Και από προσανατολιζόμαστε από πιο ουσιαστικά προβλήματα. Πρόκειται για κάποια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση. Μιλάμε για τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολεως, μιλάμε για ε, τα δικαιώματα της γυναίκας και τελικά όλα αυτά τα χειραγωγεί αριστερά παντού στον κόσμο. Μα τι, κάνουμε εμπόριο μόνο με αυτούς με τους οποίους συμφωνούμε. Τι γίνεται με την παιδεία. Λέμε ότι η παιδεία πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Όχι, η παιδεία σημαίνει γνώσεις. Άμα την παιδεία την κάνουμε προπαγάνδα, τότε πάει αλλού η υπόθεση. Γι' αυτό και εγώ ψήφισα κατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσαν λοιπόν οι υπεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Αουστρεβίτσιους γιατί δεν βλέπω και τον κύριο Μικολάσικ. Περνάμε λοιπόν στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Βίρκουνεν Μαρινέσκου Τέλιτσκα για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Τον λόγο έχει ο κύριος Μπενίτο Ζιλουάγκα. Ο μηχανισμός Connecting Europe είναι μοντέλο είναι όμω το αντίθετο από ό,τι χρειαζόμαστε τώρα που πιέζουν τα πάντα τα κλιματικά. Οπότε θέλουμε να έχουμε ένα μοντέλο βιώσιμο για τι υποδομέ, για τον αγωγό του αερίου και του φυσικού αερίου και ακόμα και για τον βυσκαϊκό κόλπο όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να μην έχουμε πια ορυκτά καύσιμα και θα υπάρξει χρηματοδότηση για αυτό το φυσικό αέριο, αλλά μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως τα αποτελέσματα επί του κλίματος θα είναι πάρα πολύ βλαπτικά. Οπότε προτάσετε η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, αυτή η άρχη. Όμως θα πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση και όχι να προάγουμε τέτοιες αμφίβολες μεθόδους. Αυτός ο μηχανισμός Connecting Europe θα χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Συνοχής για να μην έχουμε ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης προωθείται η ιδέα της στρατιωτικοποίησης για τις μεταφορές και η διπλή χρήση, πολιτική και στρατιωτική. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Τελειώσαμε λοιπόν με την έκθεση Βίρκουνεν Μαρινέσκου Τελέτσκα. Μετά στην έκθεση Γκάλερ δεν υπάρχει κανείς. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου που αφορούν την έκθεση Σαλίνη για το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και τη σχετική υπηρεσία. Μία επεξήγηση ψήφου έχουμε από την κυρία Μάιερ. Ε, ευχαριστώ. Υπερψήφισα την έκθεση και όπως μου υπέδειξε η Βρετανική κυβέρνηση υπέρ των τροπολογιών 25 και 14 για να μπορούν οι Βρετανικές εταιρείες να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά μετά το Brexit. Δεν κάνει πολλά σωστά η κυβέρνησή μας ε, τελευταία, αλλά σε αυτό έχουν δίκιο. Έχει ζωτική σημασία η Airbus, το Stevenage και η Ιταλείς την ε, περιφέρειά μου να συνεχίσουν να εργάζονται. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποδώσει 700 εκατομμύρια λίρες στη Βρετανική βιομηχανία. Βεβαίως ε, θα πρέπει να κανονίσουμε τις μελλοντικέ μα σχέσεις πριν αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το Brexit ε, δεν θα υπάρχουν ευρωβουλευτέ εδώ πέρα Βρετανοί να υποβάλουν τροπολογίε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και εμεί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ανησυχώ ότι είναι τραγική συμφωνία που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Μάιερ, αγαπητοί συνάδελφοι. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Με ειδοποιούν εδώ πέρα ότι ο κύριος Μπενίτο Σιλουάγκα μίλησε για ένα λεπτό ενώ είχε δύο λεπτά γιατί εκπροσωπούσε την κοινοβουλευτική του ομάδα για την έκθεση Βίρκουνεν Μαρινέσκου Τέλιτσκα. Οπότε θα ήθελα τώρα να του δώσω την ευκαιρία να ε, συνεχίσει την παρέμβασή του. Ευχαριστώ. Τι να έχω και τα δύο λεπτά ή να συμπληρώσω. Okay. Κύριος του Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο μηχανισμός Connecting Europe είναι το αντίθετο από ό,τι χρειαζόμαστε. Στους αντίποδες από ό,τι χρειαζόμαστε. Και το κατευθυνόμενο μη βιώσιμο μοντέλο. Οι υποδομές όπως το MidCat, το ELTAP και ο εξηλεκτρισμός του κόλπου της Βισκαΐας. Τι θα γίνει με το φυσικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια που ξοδεύονται, ενώ αυτό που θα προκύψει θα είναι πολύ βλαπτικό. Αυτό βλάπτει την αρχή της αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας, διότι αντί να κόψουμε την κατανάλωση, έχουμε τέτοιες μεθόδους αμφίβολες. Και αυτό θα γίνει με συρρήκνωση των πόρων των Ταμείων Συνοχής. Θα γίνουν χειρότερες οι ένωσες της Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε να μην στατικοποιούμε επίσης τις μεταφορές με τη διπλή χρήση, πολιτική και στρατιωτική. Αυτό από την πίσω πόρτα κατά αυτόν τον τρόπο κάνουμε κακό σε όλες τις τομιακές πολιτικές. Θα πρέπει να έχουμε μια Ευρώπη ειρήνης και οικολογικού μετασχηματισμού. Γι' αυτό και ψηφίσαμε κατά ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Μπενίτο Ζιλουάγκα και με συγχωρείτε και πάλι. Περνάμε τώρα στην έκθεση Ροσάτη. Εταιρική φορολογία εταιριών με σημαντική ψηφιακή παρουσία. Την κυρία Γεσλογιέσκα δεν τη βλέπω όμως. Οπότε τον λόγο έχει ο κύριος Σοσνιέρτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενικά είμαι κατά της αυξήσεως της φορολογίας. Εφόσον δεν είναι δίκαιη η επιβολή φόρων, τότε θα πρέπει να μειώσουμε αυτό το, τους φόρους τους οποίους πληρώνουν οι έχοντες, αλλά να μην αυξήσουμε τους φόρους τους οποίους οι μη έχοντες αναγκάζονται να πληρώσουν. Ίσως θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε και εθελοντικού τύπου φορολογικές ρυθμίσεις. Κάτι το οποίο είναι πάντα θετικό. Εγώ θέλω λοιπόν να πλουτίζει ο κόσμος εφόσον φυσικά το κάνει αυτό εθελοντικά, ενώ το αντίθετο δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό. Και σύν της άλλης έχουμε να κάνουμε με μια προϊούσα γραφειοκρατικοποίηση των συστημάτων. Εάν πράγματι θέλουμε να κάνουμε μια σωστή αναλογία για να καταλάβουμε το παράδειγμα, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργία του ίντερνετ και όχι να ελέγξουμε το ίντερνετ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση για τα συγκρόμενα συμφέροντα και προστασία του κοινοτικού περιπολογισμού στην Τσεχία. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η έκθεση αυτή έγινε δεκτή με μία μόνη τροπολογία. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τις, ε, ε, τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαίων. Και είναι σαφές ότι τα επιχειρήματα αυτά α, της τσεχικής πρωθυπουργίας δεν είναι δυνατόν να περάσουν, ιδιαίτερα μετά από την παρέμβαση ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως το, Amnesty, το, το Διεθνής Διαφάνεια κτλ δεν θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα που να αυξάνουν την διαφάνεια από τη μία αλλά από την άλλη να δημιουργούν προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε από πλευρά του Πρωθυπουργού με σαφείς παραβιάσεις και καταχρήσεις. Είναι σαφές ότι ο, ο Πρωθυπουργός της χώρας μου έχει αγοράσει πάρα πολλές οικονομικές δραστηριότητες, ε, έχει συγκεντρώσει υπερβολικά και δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στην Τσεχία. Σας ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε ο κύριος Πόσπισιλ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της ψηφοφορίας που προηγήθηκε λέγει ότι ο Πρωθυπουργός Μπάμπης έχει πρόβλημα. Αυτό το οποίο κάνει ο Μπάμπης σε τσεχικό επίπεδο ε, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δείξει ακριβώς το τι συμβαίνει στην χώρα μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση αυτή με αντικειμενικό τρόπο, με ουδέτερο τρόπο για να καταλάβουμε εάν αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες του Μπάμπη είναι δικαιολογημένες ή όχι. Το ότι είναι πρωθυπουργό ο ίδιος προφανώς δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Επίσης δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα αποκλειστικά σε τσεχικό επίπεδο. Ε, είναι σαφές ότι οι ελεγκτικές αρχές στην χώρα μου επηρεάζονται από την κυβέρνηση. Ως εκ τούτου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει σωστά τον ρόλο της και θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να λειτουργεί ορθότερα. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Τελειώσαμε και με τις επεξηγήσεις ψήφου για αυτήν την έκθεση. Και Περνάμε τώρα στην κύρια Εύη, δραστηριότητες ε, της ε, διαμεσολαβητού και θα δώσετε την τελευταία επεξήγηση ψήφου του έτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι δραστηριότητες λόμπι αποφασίζονται φυσικά και κλεισμένο των θυρών και η Ευρώπη εξακολουθεί να μην θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κάτι το οποίο αυξάνει το κόστος ε, και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Η έκθεση της ε, συγκεκριμένης υπηρεσίας φέτος αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως τις πιθανές Συγκρούσει συμφερόντων για τον τέος πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόσο, και τον παρόντα πρόεδρο φυσικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ντράγκη. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση της ηθικής και δεοντολογικής ακεραιότητας των συγκεκριμένων προσώπων. Και είναι σαφές επίσης ότι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν θα πρέπει να μην έχουν τέτοιου είδους ε, διασυνδέσεις. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Τελειώσαμε λοιπόν και με την επεξήγηση ψήφου για την δική σας έκθεση και τελειώσαμε με όλες τις επεξηγήσεις ψήφου για σήμερα, για φέτος. Η συνεδρία θα μέχρι τις 3 η ώρα. Γεια σας. Uh, uh, καλησπέρα συνάδελφοι. Συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε την ε, συνεδρίασή μας. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν από τα Χριστούγεννα, οπότε ας είμαστε αποτελεσματικοί και ας κυλήσουν όλα ομαλά. Τα πρακτικά της της συνεδρίασης και το κείμενο που υιοθετήθηκαν είναι διαθέσιμα, υπάρχουν σχόλια, όχι. Οπότε θεωρούμε πως κρίνονται. Τώρα θα προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τις ε, σπάνιες νόσους. Πρώτος ομιλητής είναι η συντάκτης Μάιστερ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγοι μείναμε, ε, είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι περισσότεροι έχουν φύγει, λογικό αυτό και σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα κανεί θέλει να ασχολείται με ωραία πράγματα και όχι με ασθένειε συνό. Θέλουμε μια σταθερή υγεία και στην Ευρώπη με τα ε, βήματα πρώτα τη ε, ιατρική ε, ήδη σχεδόν όλα είναι καλά. Το γεγονό όμω είναι ότι υπάρχουν και κάποιε σπάνιε νόσοι με τι οποίε τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά και αυτά ακριβώ τα πράγματα θέλουμε να βελτιώσουμε. Όταν μιλάμε για σπάνιε νόσοι εννοούμε ότι πλήττουν ένα άτομο να 2.000 2000 ε, και σίγουρα αυτό ε, μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλο ποσοστό, όμως ε, υπάρχουν 6 με 8 χιλιάδες διαφορετικές σπάνιες ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά πλήττονται 30 εκατομμύρια άτομα από αυτά στις νόσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστιος αριθμός. Τι σημαίνουν όλα αυτά για αυτόν τον κόσμο όταν πάρουν μια διάγνωση που κανείς ελπίζει να είναι και η σωστή γιατί υπάρχει έλλειψη βεβαιότητας σε ό,τι αφορά αυτές τις παρνίες ενώ και το πώς διαγνώνονται η ανασφάλεια αυτή δεν ε, είναι μόνο ανασφάλεια που νιώθουν οι γιατροί αλλά και οι ασθενείς και συγγενείς γιατί αν είναι γνωστή η νόσος παίρνει ένα φάρμακο και περνάει το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο ε, και πρέπει να το πω γιατί έχω και ίδια εμπειρία. Ο πατέρας μου πέθανε από μια σπάνια νόσο και ο αδερφός μου νέος σε ηλικία πέθανε από μια σπάνια ασθένεια. Η έρευνα άργησε, δεν μπόρεσε να βοηθηθεί ούτε ένας ούτε ο άλλος από τα ε, επιτεύγματα της έρευνας. Ο πατέρας μου ήταν πολιτικός ε, και έλεγαν κάποιοι εγωιστικά ότι δεν θέλαμε έρευνα να δώσουμε τότε χρήματα. Και πριν από έξι ε, χρόνια και ο γιος μου αρρώστησε. Ήταν το πρώτο κρούσμα μιας ε, νόσου σπανιότατης και ακόμα η έρευνα δεν έχει προχωρήσει. Ε, είναι μία ε, στις περιπτώσεις, ε, μία, μία νόσος. Έχει βοηθήσει κάποια άτομα η έρευνα, αλλά δεν μπορεί να τον βοηθήσει τον ίδιο. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κατάλληλη διάγνωση, δεν υπάρχει γνωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. Πηγαίνει κανείς με δοκιμή trial and error που λέμε. Δοκιμή και αν αυτή είναι επιτυχημένη ή όχι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί μακροπρόθεσμα Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε να υπάρξει περισσότερη έρευνα, να το κάνουμε αυτό με χρηματοδότηση, με ενίσχυση η βελτίωση των δικτύων που ήδη υπάρχουν ε, για τους ε, ε, πάσχοντες από μια σπάνια νόσο. Σίγουρα η ιατρική έχει κάνει πολλά βήματα προόδου σε κάποιους τομείς, αλλά σε άλλα τομεί, είναι ακόμη στα σπάργανα η ιατρική. τροπικές νόσοι, υπάρχει να μπορεί κανείς να πάρει ατροπικό ιό, όπως συνέβη με τον μου και κανένας να μην το έχει ανακαλύψει και να μην ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσουμε ε, πρόσβαση ε, των συμπολιτών μας ε, σε καλή διάγνωση, καλή θεραπευτική αντιμετώπιση δυνατών και καλά φάρμακα επομένως. Και θα σα διαβάσω τώρα ε, τις τρεις ερωτήσεις που είχαμε να καταθέσουμε προ την Κομισιόν. Ποια μέτρα έχει λάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή για να εξασφαλιστεί η ακριβή και έγκαιρη διάγνωση ε, των σπάνιων ε, νόσων, καθώ και πρόσβαση οικονομικά προσιτά φάρμακα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση τη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο τρόπο προωθεί η Επιτροπή την έρευνα στο τομέα των σπανιών και στην ανάπτυξη νέων βελτιωμένων μεθόδων για την έγκαιρη διάγνωση, πώ προτίθεται να σε αυτέ τι προσπάθειε και να επιτύχει βελτιωμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πάσχοντε από σπάνια νοσήματα σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη ερώτηση. Πώ προτίθεται η Επιτροπή να εγγυηθεί την πρόσβαση σε ενημέρωση και σε φάρμακα, καθώ και σε ιατρική θεραπεία στου τη από σπάνια νοσήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή προωθεί τον καλύτερο συντονισμό και τη μάθηση σε όλα τα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόγνωση και την ποιότητα ζωή του ασθενού Τρίτη ερώτηση, ποια είναι τα σχέδια της Επιτροπής για την εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης των οργανώσεων ασθενών που υποστηρίζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους. Για παράδειγμα, μέσω του κοινού Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις σπάνιες νόσους. Ευχαριστώ πολύ. Στον Επίτροπο τον κύριο Ανδρουκάητης θα δώσω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Καταρχάς, ως Επίτροπος, όπως και εσείς κάνατε, θέλω και εγώ να εκφράσω την ελληνική μου προς τα θύματα της φρικτής αυτής επίθεσης στο Στρασβούργο. Γνωρίζετε ότι έχουμε τρεις θανάτους και αυτό είναι πολύ οδυνηρό για μένα που είμαι και γιατρός στο επάγγελμα. Η κυρία Μάισνερ άνοιξε την καρδιά της και θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου προς εσάς για τις εμπειρίες που είχατε. Μετά από 20 χρόνια το έργο επισπανίων ασθενειών έχει δημιουργήσει δίκτυο τεχνογνωσίας και δράσεων. Υπάρχει πλαίσιο πολιτικής με τα κράτη-μέλη και ενθαρρύνουμε καινοτομία Τόμους, τρόπους εργασίας. Αγαπητέ Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, έχω έξι ερωτήσεις. Σε τρία λεπτά είναι αδύνατον να απαντήσω. Διότι ξέρω ε, ότι είναι πολύ λεπτομερείς οι ερωτήσεις. Να απαντήσω μία προς μία, διότι θέλω να παρουσιάσω μία πληρέστατη εικόνα. Αν μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, έχω πάνω από τρία λεπτά. Καλώς. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων. Πρώτα απ' όλα είναι η έγκαιρη διάγνωση των σπανίων ασθενειών. Σημαντικότατο αυτό. Κάναμε συγκεκριμένα βήματα να εξασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς να ε, μπορούν να διαγνωστούν το ταχύτερο δυνατόν. Με την έγκριση τη οδηγία, πρώτα απ' όλα, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων ασθενών σε δυσυνιακό επίπεδο, για την περίθαλψη, τα κράτη-μέλη έχουν καθορίσει εθνικά σημεία επαφή. Έχουμε 28 εθνικά σημεία επαφή. Αυτό είναι εφικτό είναι για να ενημερώνονται και γιατροί και ασθενεί, κυρίω που έχουν σπάνιε ασθένειε και ασθενεί, πώ μπορούν έχουν πρόσβαση στην ενδεδειγμένη τεχνογνωσία και γνώση που προσφέρεται προ του ασθενεί στην πατρίδα του ασθενού. Είναι διευκολύνουμε επαφέ ε, με άλλο κράτο μερο με σημεία επαφή άλλο κράτο μέρο. Δεύτερον, ψηφιακή υπηρεσία για ηλεκτρονική υγεία. Λειτουργεί υποδομή, υπάρχει, έγινε αυτό. Βοηθάει ανταλλαγή απόψεων διασυνοριακά να εξετάζονται να εξετάζει το ιστορικό στενό. Και ξεκίνησε το δίκτυο, το διευρωπαϊκό, στην Ευρώπη και έχουμε πάνω από 900 μονάδες περίθαλψης υγείας από πάνω από 300 νοσοκομεία που έχουν διασυνδεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφορά διευκολύνει την πρόσβαση σε επίκαιρη, έγκαιρη μάλλον διάγνωση και θεραπεία ανθρώπων ε, που έχουν σπάνιες ασθένειες με πολύ, ε, πολύ λίγα κρούσματα. Και έτσι υπάρχει επαφή μεταξύ των διαφόρων δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν πρόσβαση πληροφορίε. Σύστημα κλινική διαχείριση των ασθενών λειτουργεί. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο πέρσι, όπου επαγγελματίε τη περίθαλψη από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς συζητούν πραγματικές υποστασθενών και κάνουν εικονική διαβούλευση και θεραπεία. Αυτό οδήγησε σε επιτυχέστατη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ κλινικών γιατρών, εντοπίζοντα και καλύπτοντα ανάγκε ασθενών και τώρα πάνω από 250 ασθενεί από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα έλαβαν, είχαν, έτυχαν αυτή τη έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Αυτό δείχνει αποτελεσματικότητα. Μετά η άλλη ερώτηση για πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για θεραπεία. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε αρχές του έτους για οικονομικό αντίκτυπο για τα φάρμακα και τα κίνητα για τη φαρμακοβιομηχανία και πιστοποίηση για προστασία, τα μέτρα τονίζουν την έγκαιρη αντιμετώπιση των σπανίων ασθενειών και την έγκαιρη πρόσβαση στα φάρμακα. Και δίνει η μελέτη στοιχεία, συλλέγει την εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία του, κανονικού, του κανονισμού για τα ορφανά φάρμακα. Και ο κανονισμός για τα παιδιακά φάρμακα ή τα ορφανά φάρμακα, ε, η ανάλυση θα τελειώσει πριν το τέλο θητεία μου. Ίσως την άνοιξη του επομένου χρόνου. Επίσης, μέτρα για να προωθήσουμε την έρευνα στον τομέα των σπανίων ασθενειών και τη βελτίωση μεθόδων ε, έγκαιρης το ε, διάγνωση, στο έδωμα πρόγραμμα πλαίσιο και το Horizon έχουν, έχουν προωθήσει πάνω από 200 προγράμματα για σπάνιες ασθένειε σε πολύ φορητικούς τομεί και παρέχουμε πάνω από ένα δις ευρώ που χρησιμοποιούνται για τις σπάνιες ασθένειε. Ανέφερα κάποια παραδείγματα. Τα ευρωνομική και, και η Neuromics, προγράμματα που εστάζονται από της βελτίωσης διαγνωστικών μεθόδων για μεγάλες ομάδες σπάνιων ασθενειών, συμπερισμένων ασθενειών των νεφρών και σοφαρντή και προγράμματα για το ανοσιοποιητικό σύστημα βελτιώνουν τις δυνατότητες που έχουμε τα επόμενα χρόνια. Έχουμε διάφορες ομάδες, συστάδες μέτρων που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον περίπλοκο χαρακτήρα των σπανίων ασθενειών. Τώρα ερώτηση. Μέτρα για βελτίωση αποτελεσμάτων στον αφορά τη θεραπεία σπανίων ασθενών. Να πω ότι υπήρξε γνωμοδότηση του πάνελ εμπειρογνωμόνων για τη βαθμολόγηση όσον αφορά την πρόσβαση στον τομέα τη υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συμπεριλαμβανομένων των Ισπανίων ασθενειών. Και ολοκληρώνεται πιλωτικό πρόγραμμα, όπω αποκαλείται, για αποτελεσματικότερη προσμέτρηση της δυνατότητα πρόσβαση στην περίθαλψη υγείας ξεκίνησε το όλο πρόγραμμα κατόπιν ετήματος του Ευρωκοινοβουλίου και τώρα προχωράμε. Δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. Πρόσβαση στις πληροφορίες ε, καταρχάς να αναφέρω την κοινή δράση για σπάνιες ασθένειες που υποστήριξε την τελευταία τριετία την ανάπτυξη και βιωσιμότητα την, του Orphanet, της βάσης δεδομένων για σπάνιες ασθένειες. Και κωδικοποίησαμε τις σπάνιες ασθένειες στο σύστημα πληροφοριών για τις ασθένειες για να βοηθήσουμε την κατανόηση του περίπλοκου αυτού ζητήματο. Το δηλαδή, βάση δεδομένων είναι το μεγαλύτερο αποθετήριο πληροφοριών για τι πάνε ασθένειε σε παγκόσμιο επίπεδο και ένα μεγάλο κονσόρσιουμ ευρωπαϊκών εταίρων το χειρίζεται. Υπάρχει και διευθύνουσα ομάδα για την πρόθεση τη υγεία αποφυγή ε, των ασθενειών και μη διάδοση ασθενειών και κωδικοποιούνται σπάνιες ασθένειε και έχει προτεραιότητα αυτό και θα εφαρμοστούν εκεί βέλτιστες πρακτικέ. Σύμφωνα το πρόγραμμα Όρφα Coach θα υποστηριχθεί με 750.000 ευρώ με το πρόγραμμα εργασιών του 2018. Στόχος, να στηρίξουν τα κράτη-μέλη για καλύτερη συλλογή πληροφοριών για σπάνιες ασθένειες. Συλλογή πληροφοριών από 28 κράτη-μέλη. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για, για καταχώρηση σπανίων ασθενειών. Μητρό Προωθείται η διαλειτουργικότητα των εμφιστωμένων μητρώων και θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης, να βοηθήσουμε δημιουργία καινούργιων αρχείων. Έχουμε το EuroCAD και το CSBA. Εφαρμόστηκαν αυτά τα προγράμματα. Άλλη ερώτηση που κάνατε για πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και φάρμακα μας Η οδηγία για δεσυνοριακή κάλυψη των ασθενειών βοηθά τους πολίτες για ιατρική περίθαλψη άλλα κράτη-μέλη και σαφώς να ενημερώνονται για τους κανόνες για αποζημίωση, κάλυψη των εξόδων σε διασυνοριακό επίπεδο. Τώρα όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στη δυνατότητα κάλυψη των εξόδων των ασθενών με σπάνια ασθένεια. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τι σπάνιε ασθένειε που χρειάζονται ειδική θεραπεία. Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το βάση δεδομένο OFANET που είναι μοναδικό πόλο για συνάθρηση γνώσεων τη ασθένειε και για συλλογή πληροφοριών για πρόσβαση στη θεραπεία. Ζητώ συγγνώμη, διακόπτει ο Πρόεδρο. Οι διερμηνεί είπαν ότι μιλάτε πολύ γρήγορα, κύριε Επίτροπε. Μιλάτε πολύ γρήγορα, κύριε Επίτροπε. Και οι διερμηνεί παρακαλούν, αν είχα την καλοσύνη να μιλάτε λίγο πιο σιγά. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, έχουμε πίεση χρόνου. Λίγουλάκι πιο αργά, αν μπορείτε. Ε... Uh, Βέβαια, μιλούσα για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ισπανίων Ασθενειών και την καταχώρηση των ασθενειών και την πρόθεση που ήταν. Ε, α, εδώ, το είπα. Για να πετύχουμε και αυτό το κάλυψα, με συγχωρείτε. Ξέρω ότι σας ε, τάραξα και σας μπέρδεψα, λέει ο Πρόεδρος, συγγνώμη. Που είχαμε μείνει στη βάση δεδομένων όρφαν. Πάμε στα φάρμακα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ορφανά φάρμακα επαναπροσδιορίσε ε, χρηματοδότηση σε άλλους αγνοούμενους ε, παραμελημένους τομείς και δεξιότητες. Πρόκληση, ισορροπία μεταξύ κινήτων για έρευνα, να διατεθούν σωστά τα χρήματα και να υπάρχει πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για όλους και κυρίως σε αυτούς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες. Διεξάγεται μελέτη επ' αυτών των θεμάτων και θα χρησιμοποιηθεί μελέτη για αξιολόγηση των του κανονισμού για ορφανά φάρμακα και για παιδιατρικά φάρμακα. Μιλάμε για τεχνολογία, την αξιολόγηση για την τεχνολογία την υγεία. Εάν πετύχει αυτή η προσπάθεια, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για την τρίτη υποερώτηση, για πρόθεση καλύτερου συντονισμού και εκμάθηση στα κράτη-μέλη. Οι σπάνιες ασθένειες είναι τομέα συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και αν γίνει συνεργασία, δίνει προστιθέμενη αξία. Εδώ βλέπουμε πραγματικά την επικουρικότητα εν Όπου δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν θέματα σε τοπικό επίπεδο, αν δεν αντιμετωπιστούν σε τοπικό, πάμε σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό. Και αυτό ταιριάζει με την επικουρικότητα. Συνεργαζόμενοι μπορούμε να μοιραστούμε δεδομένα και τεχνογνωσία, να ξεπεράσουμε τον καταγραμματισμό και τι γεωγραφικά μενεκτούσε περιοχέ και να δοθεί σωστή διάγνωση ασθενή δημιουργήθηκε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς και ενισχύει τη συνεργασία των ερευνητών, των γιατρών και εκείνων που αναπτύσσουν θεραπείες μπορούν να συνεργάζονται αυτοί μεταξύ τους και δημιουργούν ένα δίκτυο διάγνωσης και δίκτυο ομάδων εργασίας για να δουν αυτοί οι άνθρωποι πώς να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Και βασίζουμε και στη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δικτύων Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς σε επικοινωνία με εθνικά συστήματα υγείας και να πάμε και στην πρωτογενή θεραπεία σε βάθος. Να βρούμε μονοπάτια, ή εύκολα μονοπάτια για την επίτευξη έγκαιρης διάγνωσης. Για τις άλλες ερωτήσεις. Το τρίτο τμήμα. Για βιώσιμη χρηματοδότηση των οργανώσεων ασθενών που στηρίζουν επίση τα ευρωπαϊκά δίκτυα για τις σπάνιε αναφοράς. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς οικονομικά και οργανωτικά στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος e-health και δεύτερον μέσω του μέσου για τη της Ευρώπης, Connecting Europe. Δεν υπάρχει άμεση χρηματοδότηση των εκπροσώπων των ασθενών. Κάθε ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς λαμβάνει 200.000 ευρώ ετησίως από το πρόγραμμα eHealth. Και αυτό στηρίζει το δίκτυο και βελτιώνεται η δυνατότητα συντονισμού των δικτύων, οργανώνονται συναντήσεις με εκπροσώπους των ασθενών. Το πρόγραμμα eHealth προωθεί επίσης χορηγίες για ΜΚΟ και οργανώσεις ασθενών. Το ΡΟΡΤ επίσης είναι σημαντικός φορέας και ορίζοντας 2020 και το σχετικό πρόγραμμα για το 2018 θέλει να συστήσει ευρωπαϊκό κοινό, κοινό πρόγραμμα συγχρηματοδότησης πάνης ασθένειας. Εκεί μπορούν να συμμετάσχουν τα ευρωπαϊκά δίχτυα αναφοράς και οι οργανώσεις ασθενών. Είναι ένα πρόγραμμα ε, που διαρκεί πάνω από μία πενταετία. Έτσι εξασφαλίζεται βιωσιμότητα μετά το 2020. Και γι' αυτό προτείναμε στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υποστήριξη να δίδεται μέσω άμεσων χορηγιών. Και τώρα είναι στο χέρι όλων μας αυτό. Και οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαθωτικά ταμεία, δημιουργώντας κέντρα και να χρησιμοποιήσουν και το κοινωνικό ταμείο για να στηρίξουν την εκπαίδευση των ιατρών και τις δεξιότητες γιατρών και του νοσηλευτικού ε, προσωπικού. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι που μου δώσατε δυνατότητα να σας διαμερώσω για το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων για τις ασθένειε. Αυτές οι δράσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα ε, του προγράμματο για την υγεία και την έρευνα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνουμε η αξία στου ασθενεί και στου οικογένειε. Διασυνδέοντα την τεχνογνωσία σε όλη την Ευρώπη, ε, αυτή είναι η δική μου προτεραιότητα και στόχο μου. Σα ευχαριστώ. Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διεξοδικότατη η απάντησή σα, τουλάχιστον όπω τα βλέπω τα πράγματα. Θα πάμε τώρα στου ομιλητέ που εκπροσωπούν τι διάφορε πολιτικέ ομάδε και θα μιλήσει ο καθένα ε, ένα δίλεπτο. Η κυρία Πίτικα είναι εκ μέρους του ΕΛΚ έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή καταρχάς γιατί δραστηριοποιήθηκε ε, πραγματικά ε, για το θέμα των σπανίων νόσων. Εάν είναι κάτι που πρέπει να φτιάξουμε, Να ξέρουμε ότι υπάρχουν 8.000 σπάνιες νόσοι και 10% των Ευρωπαίων υποφέρουν από κάποια σπάνια τέτοια ασθένεια. Ε, είναι σπάνια στη πόλη του ή στη σπάνια στο κράτο μέλο του, που δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουν όλε τι γνώσει, τι θεραπευτικέ δυνατότητε ή τα, την αγωγή. Γι' αυτό και χρειάζεται μια τελείως νέα ευρωπαϊκή συνεργασία που θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα ε, για άλλες ε, νόσους, ε, γιατί θα πρέπει να έχουμε για όλες τις δυνατότητες για όλες τις σπάνιες νόσους. Όπως είπατε, έγκαιρη διάγνωση χρησιμοποιώντας την ε, πρωτοβουλία διασυνοριακής υγείας και το e-health είναι και παραδείγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να διοχετεύσουμε κάποια παραπάνω κονδύλια από το Horizon στο μέλλον ώστε να φτιάξουμε δίκτυα και σημεία αναφοράς για τις σπάνιες νόσους για, ως παράδειγμα για να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ε, Δυνατότητε οι γιατροί να μπορούν να, να κάνουν διάγνωση για αυτές τις σπάνιες νόσους εγκαίρως. Και να υπάρχουν βέβαια και οι οδηγίες για περαιτέρω αγωγή στους ανθρώπους που υποφέρουν από αυτές τις νόσους. Τέλος, είναι ένα θέμα για τη ιατρική ε, και των ορφανών φαρμάκων που είναι εξαιρετικά δαπανηρά, αλλά και πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι τόσο δύσκολο. Γι' αυτό θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα ευρωπαϊκό ταμείο που θα αγοράζει τα ορφάνα φάρμακα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ, αλλά πρέπει να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αν δεν έχουμε μεγάλη ημερήσια διάταξη, θα σας ζητήσω να σέβεστε την, ε, το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ Μαμίκινς, δύο μισή λεπτά τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Περίπου 5.000 με 8.000 διαφορετικές σπάνιες νόσοι επηρεάζουν 6 με 8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, δηλαδή 30 με 37 εκατομμύρια άνθρωποι. Κλινική έρευνα στον τομέα των σπάνιων νόσων είναι πολύ κατακαιρματισμένη. Το πρόβλημα αυτό μπορούμε να το λύσουμε μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωπαϊκός στόχος ε, για τις σπάνιες νόσους είναι να υπάρχει ειδική πρόσβαση στη διάγνωση, την ενημέρωση και την ε, φροντίδα. Να, καταρχάς να εξασφαλίσουμε ότι οι σπάνιες νόσοι θα κωδικοποιηθούν επαρκώς και θα μπορεί όλα τα συστήματα υγείας να, τα, να τις αντιμετωπίζουν. Στήριξη έρευνα στις ευρωπαϊκές ε, χώρες για τις σπάνιες νόσους, ε, βελτίωση της αναγνώρισης και της ορατότητας των σπανίων νόσων και έπειτα ε, δημιουργία δικτύων και κέντρων αριστείας και εμπειρογνωμοσύνης ώστε να μπορούν οι εμπειρογνώμονες των διάφορων χωρών να ανταλλάσσουν απόψεις και να εντοπίζουν διαφορετικές δυνατότητες αγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τη στήριξη στην έρευνα μέσω του Horizon 2020 στα ευρωπαϊκά πλαίσια προγράμματα πλαίσια για την έρευνα και την καινοτομία και για την πλατφόρμα καταγραφής των σπανίων νόσων που αναφέρθηκε από τον Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σπάνιες νόση είναι το μέσο που μπορεί κανείς να δει πρόοδο να δημιουργήσει συνεργασία, έρευνα και ανάπτυξη. Και αυτό ακριβώς επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε σε Επόμενος εκ μέρους της Άλντε, κύριος Γιάκοφτσίτσε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ...10% περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχουν προσβληθεί από κάποια σπάνια νόσο. Πάνω από 5.000 είναι αυτές οι σπάνιες νόσοι. Μία σπάνια νόσος, είναι σπάνια, όταν από αυτήν ε, έχουν προσληθεί λιγότεροι από 2.000 άνθρωποι. Και μιλάμε για προσωπικές τραγωδίες. Ε, μας τις περιέγραψε και η συνάδελφος Μάισνερ. Πρέπει να μιλήσουμε για τις ανθρώπινες αυτές ζωές και τη μοίρα αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να προσέξουμε αυτά τα οποία ακούσαμε και μιλάμε εδώ για τη δημόσια υγεία, την ιατρική, αλλά αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε βάσεις δεδομένων, δημιουργία δικτύων και μεταξύ της Ρήγα, του Ταλίν, της πόλης μου, να μπορεί να γίνει ανταλλαγή δεδομένων και αυτό να γίνεται ως το δυνατόν πιο έγκαιρα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για προτάσεις σημαντικές, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σπάνιες νόσους. Μου φαίνεται όμως, κύριε Επίτροπε, ότι αυτό το οποίο πρέπει να προτείνεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ένα παγκόσμιο συνασπισμό. Μια παγκόσμια συμμαχία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και άλλες οργανώσεις. Είναι όριμος ο καιρός για κάτι τέτοιο. Η Ιαπωνία, η και πλούσιες χώρες θα έπρεπε να ενταχθούν σε αυτή τη συμμαχία και όλες, σας, όλες όσες χώρες το θέλουν για να υπάρχει μια κοινή βάση καταπολέμηση αυτών των σπάνιων νοσών. Γιατί αν ε, έχουν προσβάλει 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, ε, δεν ξέρω παγκόσμια τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να πολύ περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ρόλο μπορούμε να ασκήσουμε και εμεί. Λόπε Μπερμέχο για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από 6.000 είναι οι σπάνιες νόσοι οι οποίοι ε, έχουν προσβάλει πάνω από 30 εκατομμύρια Ευρωπαίου, είναι χρόνιες νόση σε μεγάλο βαθμό και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των πληγέντων. Όπω λέει το Γιούρντι, είναι λίγο συχνέ μεν οι νόσοι αυτέ. Όμω οι πάσχοντε είναι πολλοί. Είναι πολλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενεί. Έλλειψη πρόσβαση σε διάγνωση, σωστή ενημέρωση, κοινωνικέ επιπτώσει, εκπαιδευτικέ, εργασιακέ, αναψυχέ κτλ. Ανισότητα σε ό,τι αφορά τι διαθέσιμε θεραπείε, υψηλό κόστο φαρμάκων. Πολύ μακρύς ο κατάλογος των προβλημάτων, αλλά οι λύσεις περιορίζονται στην ε, υιοθέτηση ε, μάλλον μέτρων που προτείνουν χρηματοδότηση για δημόσιους πόρους, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Πράγματι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε με τη δημόσια υγεία, γιατί μόνο έτσι μπορούν όλοι οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε διαγνώσεις και θεραπείες επίσης όρις, να μην εξαρτώνται από τους οικονομικούς πόρους τους δικούς τους ή των συγγενών τους, γιατί Ακριβώς αυτό είναι που προκαλεί και μια επιπλέον ανισότητα. Να απαραίτητο λοιπόν ε, να δοθούν πόροι και για την έρευνα και επιμένω δημόσιοι πόροι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ιδιωτική έρευνα λόγω του κόστους ακριβώς που δημιουργεί η επίλυση των προβλήματων αυτών και χρειάζονται πόροι για την μη ιατρική παρακολούθηση, τη στήριξη, την κοινωνική, την, την οικογενειακή για την αποκατάσταση κτλ. κτλ. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε αυτές τις δημόσιες πολιτικές που είναι αναγκαίες, ώστε οι ασθενείς να μην υποφέρουν πέραν της ε, πάθης αυτής ε, ε, και, του προβλήματος να, να υποφέρουν και από αυτήν την αδιαφορία και την απαθή. Κυρία Μιράντα τώρα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι σπάνιες νόση μας ανησυχούν. Μία, οι σπάνιε νόσοι όντω είναι σπάνιε, αλλά οι άνθρωποι που υποφέρουν από τι σπάνιε νόσου είναι ε, πολλοί. Γνωρίζω πολλέ οικογένειε που πληρώνουν υψηλό κόστο. Ε, για, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μελήσουν, για να συγκεντρώσουν χρήματα για αυτές τις ε, ε, ακριβές ε, αγωγές. Συχνά αυτές οι οικογένειες αισθάνονται μόνες. Μια ασθένεια μπορεί να πλήττει έναν άνθρωπο, όμως μπορεί να, να επηρεάσει και πολλούς περισσότερους. Η, Κομισιόν αναγνωρίζει πως οι ασθενείς ε, είναι ιδιαίτερα απομονωμένοι και ευάλωτοι. Είναι σημαντικό, όπως είπε ο Επίτροπος, να κωδικοποιηθούν, να, να αρχιοθετηθούν και να γίνουν έρευνες, να ανοίξουν ειδικευμένα κέντρα και ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις πάνες νόσους. Και επίσης για μας είναι απαραίτητα περισσότερα κονδύλια να μπορέσουμε να, χρησιμο... να συνεργαστούμε διασυνοριακά ε, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να αποφεληθούν από αυτές τις αγωγές. Επίσης για τα, σπάνια, για τα ορφανά φάρμακα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει περισσότερα κονδύλια ώστε αυτοί οι άνθρωποι να, ε, να μπορούν να θεραπευθούν ισότιμα με τους υπόλοιπους. Έλισεν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ τα όσα μας είπε η κυρία Μέστερ. Ε, λοιπόν, ε δεν θα διαφωνήσει κανείς εδώ ότι ε, ένα σωρό κόσμος που αγωνίζεται με αυτές τις ε, σπάνιες νόσους αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία να είναι προσιτά. Όμως, Πρόεδρε, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Πρέπει να γίνονται επιλογές και αυτές οι επιλογές γίνονται από τα κρατημέλη. Οι Ολλανδοί θα πρέπει να αποφασίζουν πώς θα είναι η υγεία στην Ολλανδία, αν κάποιο φάρμακο αποζημιώνεται από την ασφάλιση ή όχι. Είναι θέμα του Εθνικού Κοινοβουλίου. η φροντίδα για τους ηλικιωμένους, ε, η... τα κονδύλια για την υγεία είναι εθνικό θέμα και πρέπει να παραμείνει εθνικό θέμα. Υπάρχουν 28 27 κρατημέλη με 27 διαφορετικά συστήματα υγείας. Θα ήταν πολύ κακή ιδέα να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τα συστήματα υγείας και να φτιάξουμε ένα μόνο ευρωπαϊκό υγειονομικό σύστημα, γιατί αυτό θα ήταν ίσως ο στόχος των ευρωπαϊστών εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμως αυτό θα γίνει εις βάρος, αν γίνει εις βάρος των υπολείπων. Η Ευρώπη αποτελείται από διάφορα έθνη και λαούς. Ο καθένα έχει τις παραδόσει του και τα χαρακτηριστικά του. Δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει μόνο ένα μοντέλο που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Η ε, θεραπεία είναι θεραπεία ε, ε, ανακράτωση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ορίζεται από, τον από τα εθνικά κράτη, όχι από τον πύργο του Στρασβούργου. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη δικασία προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου. Δεν βλέπω να είναι κανείς, οπότε να πάρει το λόγο επίτροπος ε, για να κλείσει τη ζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα να απαντήσω στον τελευταίο ομιλητή αν με επιτρέπετε. Αν στην Ολλανδία εσείς έχετε 10 άτομα που είναι ασθενείς σπάνιο νοσήματος, δεν υπάρχουν κλινικοί, δεν υπάρχουν επαγγελματίες υγείας, δεν υπάρχουν δυνατότητες αυτά τα 5 άτομα να λάβουν θεραπευτική αντιμετώπιση. Εγώ 20 χρόνια ασχολήθηκα με τις θεραπείες δεν μπορείς να πας να πεις πού είναι ένα κέντρο αριστείας, γνώσης, διάγνωσης, ε, ε, θεραπείας ε, νόσων. Χρειάζεται συνεργασία. Αυτό πρέπει να μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περί αυτού πρόκειται. Δεύτερη δυνατότητα. Δεύτερη δυνατότητα. Και εδώ απευθύνομαι και σα, ως ο Γιάκοφ Τσίτσε. Είπατε κάτι που είναι μια πολύ καλή ιδέα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο αναφορά είναι σπονδυλική στήλη και μπορεί να μας βοηθήσει τα πανεπιστήμια, τα διάφορα άλλα ιδρύματα, του ερευνητέ και όσους αναπτύσσουν ε, θεραπείε, προηγμένες θεραπείες, θεραπείε ακριβώς όπως τις λέμε, να του συνενώσουμε στο ίδιο δίκτυο. Βέβαια, θα λύνουμε τα κράτη-μέλη να υπογράφουν ε, την ε, συμφωνία για το 1 εκατομμύριο γονιδιώματα. που μπορεί να είναι ένας ε, μηχανισμός που συγκεντρώνει όλες αυτές ε, τις ε, πληροφορίες και μπορεί να αναπτύξει νέες θεραπείες, να είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη για νέες διαγνωστικές δοκιμές και νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σίγουρα η συνεργασία εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ευκταίο. Για τα big data, τα μεγάλα δεδομένα, χρειάζονται και πρωταγωνιστές. Δεν είναι αρκετά υψηλά τα περιφερειακά μητρό. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ θα ήθελα να προωθήσω αυτή τη διαδικτύωση ώστε να έχουμε μεγάλα δίκτυα big colliders και να ενώνουμε που θα δράσουν ως επιταχυντές. Θέλω να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να βρουν τη χρηματοδότηση, γιατί ξέρουμε πόσο θα η έρευνα και πόσο θα τα φάρμακα. Μόνο οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να μας επιτρέψουν την πρόσβαση στις ε, θεραπείες και να μην κάνουμε διάκριση τι σημασία έχει που είναι ο ασθενή, αν στην Κύπρο, στη Λιθουανία ή στην Ολλανδία. Η πρόσβαση στη θεραπεία και στην καινοτομία είναι ένα οικουμενικό δικαίωμα και πρέπει να κάνουμε πιο πολλά για να υπάρχει οικουμενικότητα αυτή. Α είναι και στη Φιλανδία, α είναι και στη Μάλτα ο ασθενή. Πρέπει να το σκεφτούμε όλο αυτό το πρόβλημα. Είναι σαφές βέβαια ότι δεν έχει καμία μόνη της ε, χώρα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μεμονωμένα. Αν ε, δράσουμε ιδιωτικά δεν θα υπάρξουν διαγνώσεις, δεν θα υπάρξουν ε, αποτελεσματικές θεραπείες, θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλά από κοινού μπορούμε να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες, να συγκεντρώσουμε δεδομένα, να δράσουμε πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά και πιο αποφασιστικά και έτσι θα ωφεληθούν και οι ασθενείς στην Ευρώπη. Είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα της δύναμης της συνεργασίας Ισπανής Νόση για την έρευνα, για την κωδικοποίηση τα διάφορα μητρώα και ιδίω για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς. Όμως, πρέπει να φροντίσουμε οι ομάδες ασθενών, οι ΜΚΟ, να μεγιστοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Τα γνωρίζουμε, τα προβλήματα πρόσβασης ε, και έλλειψης δεξιοτήτων για τους ασθενείς με σπάνια νόσο. Έχουμε την ομάδα Βαλέτα, ε, ομάδα συνεργασίας, πρόσβαση στην ε, θεραπεία. των Μπένελουξ, οι χώρες Μπένελουξα και Αυστρία συνεργάζονται επίσης. σε ό,τι δεν αφορά τη νομοθεσία για τα ορφανά φάρμακα. Θα κάνουμε μια ανάλυση που θα μα δώσει τη δυνατότητα να δούμε τι γίνεται με του ασθενεί που έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα. Ολοκληρώνοντα, να πω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει του ασθενεί οι οποίοι υποφέρουν από μια σπάνια νόσο. Είναι αυτή η δέσμευσή μα και την βλέπετε και ε, στο σκέλο υγεία και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ και στο πρόγραμμα Ευρώπη Ορίζον Ευρώπη και σας παρακαλώ να στηρίξετε τις προτάσεις Κομισιόν για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ για την απαντήσεις σας. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο και τελευταίο σημείο της σημερινής σημερινής διάταξης που είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εξάπλωση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων. Πρώτος είναι ο κύριος Σικέρσκι που είναι και ο συντάκτης για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, συνάδελφοι. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανησυχεί για την κατάσταση που έχει προκληθεί από την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στις εκμεταλλεύσεις. Αυτό έχει επηρεάσει τις αγορές, τους κτηνοτρόφους και προκαλεί πολλά και διάφορα προβλήματα. Το θέμα έχει συζητηθεί επανειλημμένα στην Επιτροπή Γεωργίας. Πολλοί ε, βουλευτές από τις χώρες που θίγονται έχουν διοργανώσει ακροάσεις και διασκέψεις επαφές με τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί. Γι' αυτό και ε, στραφήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την προφορική μας ερώτηση για να συζητηθεί το θέμα και στην Ολομέλεια. Πρόκειται για μια σπάνια ε, νόσο των χείρων. Είναι ε, μια λιμώδης νόσος. Είναι ένας κίνδυνος που επιφέρει οικονομικές ζημιές στον τομέα ε, κτηνοτροφίας ε, χείρων. Κάποιες φορές ε, εισάγονται χείρι, χείριο κρέας ή προϊόντα χείριου κρέατος από χώρες που έχουν πληγή από την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων και το μικρόβιο μπορεί να μεταφερθεί και σε μεγάλες αποστάσεις και να ε, πλήξει περιοχές που παλιότερα δεν είχαν πληγεί. Η πρόληψη ε, και η καταπολέμηση της ασθένειας απαιτούν μια γενική ε, συνεργασία όπου συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι κτηνοτρόφοι. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να διαδίδουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τους κτηνοτρόφους έτσι ώστε να μπορούν εκείνοι να παρέμβουν άμεσα ώστε να ε, ε, αναχαιτήσουν τη διάδοση της αρρώστιας. Ε, της νόσου Τα μέτρα ελέγχου έχουν υποδειχθεί από την Κομισιόν, πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης της ε, νόσου, τόσο στις ε, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όσο και στους αγριόχειρους. Με ποιο τρόπο ε, συντονίζει η Επιτροπή όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρχει ε, να, μάλλον να συντονίζονται αυστηρές δραστηριότητε όλων των αρμοδίων ε, αρχών στους τομείς της υγείας των ζώων, της άγρια, χλωρίδας και πανίδας και των οδικών μεταφορών καθώς και στο τελεινικό ε, τομέα. Επίσης, δεύτερη ερώτηση, ποια μέτρα ε, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομή συνδρομής στους πηγέντε και κτηνοτρόφου, σχεδιάζει η Επιτροπή να λάβει, για τον καλύτερο έλεγχο και την εξάλληψη τη νόσου, γιατί μέχρι στιγμή δεν θεωρούνται αρκετά τα μέσα. Τρίτον, πώς αντιμετωπίζει η Επιτροπή της δυσανάλογε απαγορεύσει που επιβάλλουν ορισμένε τρίτε χώρε στι εξαγωγή χείριου κρέατος και χείριων προϊόντων από τα πληγέντα κράτη-μέλη, η κατάσταση της αφρικανικής πανόλης των χείρων πρέπει να θεωρηθεί απειλή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, στους θεσμούς, σε κάθε επίπεδο, περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό. Πώς μπορούμε να ενεργήσουμε, πώς μπορούμε να δράσουμε και να συντονίσουμε τις διάφορες υπηρεσίες ώστε να εγγυηθούμε τη δραστηριότητα, την μεταποίηση, το εμπόριο και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτού του είδους τις απειλές που μπορεί να προκύψουν και να είναι εξαιρετικά αρνητικές για ολόκληρη την Ένωση. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για έκτακτες καταστάσεις, ειδικέ καταστάσεις όπου υπάρχει απειλή για την ασφάλεια διαφόρων τομέων. Πιστεύω πως αυτό απαιτεί μία ε, πανοραμική εικόνα, πολλές δραστηριότητες γίνονται, αλλά είναι σημαντικό να προετοιμαζόμαστε ώστε να μπορούμε να αντιδράμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η πρόληψη, ο έλεγχος και η εκρίζωση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τομέα του χειρίου κρέατος. Είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή χειρίου κρέατος και από τους μεγαλύτερου παραγωγούς στον κόσμο. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από όταν εντοπίστηκε στην Ευρώπη η ασθένεια, έλαβε σημαντικές, σημαντικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείνοντα τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δώσαμε οικονομικού πόρου και ανθρώπινου πόρου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να αναφερθώ στι ερωτήσει σα. Πρώτον, πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητε των αρμοδίων αρχών συντονίζονται στενά να πω ότι πάντα συντώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κίνηση Ευρωπαϊκή Ενώση από την πρώτο σύμπτωμα ε, που εντοπίστηκε τη πανόλη των χείρων. Εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες την τον του χρόνου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν διατομιακή, ε, διοργανική, διασυνοριακή συνεργασία και συντονισμό. Και έτσι θα ελέγχουμε καλύτερα, υπολαμβάνουμε καλύτερα την ασθένεια. Τα κράτη-μέλη και εμπλεκόμενοι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω συνεχώ συνεργάζονται μαζί μας Θέλουμε να αναπτύξουμε και να θεωρήσουμε τη στατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό, για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Καλύπτουμε όλες τις πτυχές της ασθένειας. Από την κακή υγεία των ζώων και τη βιοασφάλεια, από τις οδικές μεταφορές, τελωνιακό έλεγχο, τι γίνεται με τους άγριους χείρους και εκστατείε ευαισθητοποίησης. Τακτικά οργανώζουμε συναντήσεις με τους υπουργούς, τακτικά, κάθε εξάμεινο οι επικεφαλής ε, των κτηνιατρικών τμήματων, οι ειδικοί, κυνηγοί, γεωργοί, περιβαλλοντολόγοι, ε, διοργανώνουν εκδηλώσεις, διασκέψεις, συνέδρια. Και εκεί μπορούμε να παρουσιάσουμε ε, όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε. Η επόμενη συνάντηση, συνεδρίαση γίνεται την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης, όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας και οι Υπουργοί Περιβάλλοντος προσεκλήθησαν από κοινού να συζητήσουν το θέμα για τη διαχείριση στρατηγική για τα αγριογούρουνα, ε, βιοασφάλεια στα δάση και το θέμα της βιοασφαλείας στην κτηνοτροφία και δυνατότητες κατανόησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων σχετικά με τον πληθυσμό των αγριοχείρων. Έχουν ειδοποιηθεί τα Εθνικά Κοινοβούλια των διαφερομένων χωρών. Επισκέφτηκα Διάφορε χώρε Έχω συναντηθεί με επιτροπέ γεωργία, επιτροπέ ευρωπαϊκών υποθέσεων, κοινωνικών θεμάτων και τα συζητήσαμε με τα εθνικά κοινοβούλια. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ελέγξουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειωθεί ο κίνδυνο τη διάδοση ασθένεια μέσω των ανθρώπων. Και στείλαμε οδηγίε συγκεκριμένε στα τελωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κίνδυνο του ανθρώπινου παράγοντα, όπω αποκαλείται, τονίστηκε πρόσφατα σε επιστολή προς τους Υπουργούς Μεταφορών. Την υπέγραψα από κοινού με τη συνάδελφό μου Βιολέτα Μπούλς. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης έχουν γίνει στις πληγήσεις περιοχές. Στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να ενημερώσουμε τους οδηγούς να μην πετάνε ε, κρέατα στους δρόμους. Χρειάζεται έλεγχος ε, ενεργός και παθητικός σε όλη την Ευρώπη σημασία ε, των μέτρων αυτών έχει τονιστεί στα κράτη-μέλη και στα στα δυνατά επίπεδα έχουν γίνει εξτατείε ευαισθητοποίηση. Εμεί θα κάνουμε ελέγχου και αποστολέ να εξασφαλίσουμε εναρμονισμένη εφαρμογή ε, των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των σχετικών μέτρων. Έχουμε ετήσιες διπουργικές συναντήσεις πάνω σε αυτό. Η επόμενη συνάντηση διπουργική η διάσκεψη διπουργική θα γίνει στις Βρυξέλλες. 19 Δεκέμβρη. Σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί συντονισμένη πρόληψη και ύψη στο επίπεδο ετοιμότητας, έλεγχο και κρίζωση τη ασθένειας από τα κράτη-μέλη. Δεύτερη ερώτηση. Τι βήματα σχεδιάζει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καλύτερο έλεγχο και κρίζωση τη ασθένειας. οικονομική βοήθεια που θα δοθεί στους ε, κτηνοτρόφους. Έχουμε τεχνολογία, επιστήμες, οικονομικά μέσα, τεχνικά μέσα. Υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη σωστή τη ασθένεια. Συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγείται προ τα κράτη-μέλη και είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη και κρίζωση ασθένεια. Χρειάζονται πρωτοβουλίε ευαισθητοποίηση που μπορεί να συγχρηματοδοτηθούν στα κράτη-μέλη εκεί που δεν υπάρχει ασθένεια για να αποφευχθεί η διάδοση μέσω ταξιδιωτών κυνηγών και άλλων ομάδων κινδύνου. Περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για την ασθένεια αυτή για το 2013 μέχρι το 2018. Να τονίσω ότι έχουμε πρωτοβουλία που βασίζεται σε σωστή επιστημονική ε, συμβουλή και εμπειρία. Θα εξακολουθούμε να συντονίζουμε διάφορες δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη, έλεγχο και κρίση της ασθένειας. Πολιτικός συντονισμός θα προωθηθεί. Θα οργανώνονται υπουργικέ συναντήσει τακτικά. Έλεγχο και έρευνα τη υφιστάμενη νομοθεσία και τοπικά μέτρα. Χρειάζεται εναρμονισμένη στατική προσέγγιση για τη διαχείριση ασθένεια. Να γίνονται έλεγχοι, αποστολέ. Χρειάζεται τιμότητα, άμεση βοήθεια, επιτόπια, εμπειρογνώμονες να πηγαίνουν στα πληγέντα κράτη-μέλη ειδικοί κτηνίαται να πηγαίνουν στι πληγήσει περιοχέ. Χρειάζεται διεθνή συνεργασία, ενεργή συμμετοχή, προώθηση του παγκόσμιου πλαισίου για την καταπολέμηση των διασυνοριακών ασθενειών στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, να προωθηθεί επίση η έρευνα στον τομέα αυτή τη ασθένεια, να αναπτυχθούν εμβόλια. Περίπου 25 εκατομμύρια έχουν, ευρώ έχουν αφιερωθεί για την ανάπτυξη εμβολίων μέσω έρευνας. Χρειάζεται να αναπτυχθούν συγκεκριμένα προγράμματα σε γειτονικέ χώρε, όπω είναι η Μολδαβία και η Ουκρανία, που συνεργάζονται στι παραμεθόριε περιοχέ. Τρίτη ερώτηση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αντιμετώπιση των δυσανάλογων απογορεύσεων σε τρίτε χώρε τη εξαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζωών των ζώων, χειρίου κρέατος και προϊόντων χειρίου κρέατος. Συνεργαστήκαμε με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους των Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να επικρατεί πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την κατάσταση στον την ασθένεια και τα μέτρα που έχουν ληφθεί βάσει των διεθνών προδιαγραφών. Τελευταία συνάντησή μου έγινε στην Κίνα. Συζητήσαμε αυτά τα θέματα με τους Κινέζους για την εξαγωγή του χειρίου κρέατος. Και περιφερειο περιφερειακά μέτρα ήταν επιτυχή εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όποτε είχαμε ε, ξέσπασμα της ασθένειας. Ε, οπότε είχαμε περιορισμούς εμπορικούς από τις πληγήσεις περιοχές και η υπόλοιπη, περιοχή η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάστηκε. Και δεν είχαμε ε, κάποια ζωονόσο ε, που ξέσπασε μετά. Σε διμερεί επαφέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από του εμπορικού εταίρου να αναγνωρίσουν ε, τα μέτρα περιφερειοποίηση για τι του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα αυθυγραμμίζονται με τι διεθνεί προδιαγραφέ που προωθούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και αποφεύγουμε αδικαιολόγητου εμπορικού φραγμού. Αυτή είναι σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλε οι σχετικέ υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται στενά επ' αυτού και θα ήθελα να αναφέρω ότι την περίπτωση του ΠΟΗ μια υπόθεση προσφυγή κατά της ε, ρωσική απαγόρευση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευμένη περαιτέρω να προωθήσει τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για καταπολεμική η ασθένεια αυτή, να βρούμε μέσα συντονισμού με τα κρατημέλη, του εμπλεκόμενου φορεί. Αυτό θα βοηθήσει τη βελτιστοποίηση τη απάντησης που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την ασθένεια και θα μαζέψουμε όλου του δυνατού πόρου κατά πολέμηση τη ασθένεια και να αποφύγουμε τη διάδοση αυτή τη ασθένεια. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και τώρα για το ΕΛΚ, για δύο λεπτά, ε, ο κύριο Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ όσους ε, έχουν καταστήσει δυνατή την πολύ σημαντική αυτή συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω ε, τον Φιλ ε, Χόγκαν τον Επίτροπο που στήριξε τους Ρουμάνους αγρότες που επλήγησαν από τον ιό. Ρουμάνοι αγρότες δυστυχώς ε, πλήγησαν ε, πολύ σοβαρά από αυτό τον ιό ε, και υπάρχουν οι αποζημιώσεις μεν που δεν είναι και κάτι ικανοποιητικό γιατί το πιο χρήσιμο θα ήταν η πρόληψη. Θα πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη διαφοροποίηση μέτρων για να είναι πιο αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπογράμμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη μόνο παρέχοντα βοήθεια στα κρατη μελη εκ των υστέρων. Πρέπει να αναβαθμίσει τι προσπαθίε τη. Πρέπει να κινητοποιηθεί και να καλεί τα κράτη-μέλη ε, να συμμορφωθούν όταν δεν σέβονται τα ε, μέτρα που και τα πρότυπα. Υπάρχει μια πολύ επιθετική ε, αυτή είναι πολύ επιθετική νόσο, αφρικανική πανόλη των αρχείων και μπορεί να μεταφερθεί και μέσω των μεταναστευτικών, των αποδημητικών πτηνών, μπορεί να διτηρηθεί στο ε, κατεψημένο κρέα για πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι χείροι και οι αγριόχειροι να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και οι κυνηγοί έχουν ένα ρόλο να δραματίσουν. Δυστυχώ δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και πρέπει να πάρει μέτρα η Κομισιόν. Πρέπει να καταλάβει η Κομισιόν ότι αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την πανόλη, δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο μέσο και τρόπο από την καύση των σφαγείων. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται υποδομέ. Κινητέ μονάδε καύση ε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί που έχει χτυπήσει ο ιός. Και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει επαρκή χρηματοδότηση ώστε να υπάρξει και περισσότερη έρευνα για να βρεθεί το εμβόλιο κατά του Ισπανόλης αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρος τώρα για την Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για έξι λεπτά η κυρία Γκυλέρα Καρθία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη που γίνεται αυτή η συζήτηση και με την πρωτοβουλία της ε, Επιτροπής Γεωργίας ε, για την ε, Αφρικανική Πανόλη των Χείρων μια σημαντική συζήτηση όπως και αν, όποτε και αν προέρχεται, όποτε και αν γίνεται συγγνώμη παρότι ίσως δεν είναι ακριβώς πάντα η κατάλληλη χρονική στιγμή. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μέτρα αλλά δεν εφαρμόζονται σωστά εφαρμόζονταν υπαρκώ. Και γιατί το λέω, στην Επιτροπή Γεωργία είχαμε εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση που ουσιαστικά μα δημιούργησαν πιο πολλέ ε, αμφιβολίε από ό,τι μα καθυσίρασαν. το λέω. Και άκουσα πολύ προσεκτικά την παρέμβασή σα. Ε, ξέρω τι κάνετε, κάνετε πάντα δυνατόν. Αλλά δεν μεταφέρεται πάντα σωστά αυτό και σε ό,τι αφορά το εμπόριο και σε ό,τι αφορά τον κλάδο δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλε αμφιβολίε και ανασφάλεια. Παραδείγματο χάρη, ό,τι αφορά τη διάδεση μέσω των αγριόχειρων, πώ θα ελεγχθεί, λένε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει να το πείτε ότι πράγματα γίνονται, αλλά ε, πρέπει να είμαστε πιο βέβαιοι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εγώ είμαι από την Ισπανία, την Ανταλουσία, την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Ε, τη βιώσαμε για 40 χρόνια και την εκριζώσαμε. Αυτό κόστησε πολλά και χρόνο και χρήμα. Τώρα είναι απαραίτητο να το συζητήσουμε και γι' αυτό χρειάζεται και αυτή η συζήτηση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη στρατηγική πολύ περισσότερο από το δικό σα επιδρομοδοτήτων, γιατί έχουμε να κάνουμε και με τι μεταφορέ και με άλλα στοιχεία που επηρεάζουν. Άρα θέλουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Όχι μόνο για την ε, υγεία των ζώων, αλλά πιο γενική στρατηγική. Ποια είναι η άποψή μου. Έχουμε τρεις τιμές. Πρώτον, ε, όταν μπαίνει από τις χώρες της Βαλτικής ή από τη Ρωσία ο ιός ε, και επηρεάζονται και ένα τρίτο της Πολωνίας. η Πολωνία κάπως πολωνια η πολωνια καπως ελεγχει την κατάσταση, τρία τέταρτα της επικράτειας της δεν έχει πληγεί από τον... αλλά δεν φαίνεται να είναι ελεγχόμενα τα πράγματα στις χώρες Βαρτικής. Πρώτης, πρώτος χρόνος αυτός, δεύτερος χρόνος για την Ρουμανία. Τα είπε ο κύριος Μπούντα που ανησυχεί. Η κατάσταση στη Ρουμανία είναι ανησυχητική. Γιατί εκεί είχαμε το εξή. Ξέσπασε μια ε, επιδημία. Και λόγω του παραγωγικού σύστηματος, κατά την ταπεινή μου άποψη, που είναι απαρχιωμένο, κατά πιθανότητα και λόγω του κτηνιατρικού συστήματος που είναι ανεπαρκέστατο. Πάντα προσωπική μου άποψη. Πρέπει να βοηθηθεί η Ρουμανία, διότι τελικά αν δεν βοηθήσουμε τη Ρουμανία, το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όλοι. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι σύστημα παραγωγικό, κτηνιατρικό σύστημα. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα στα συστήματα με ευρωπαϊκά ταμεία, ε, κονδύλια από όλου μα. Και όχι μόνο με το δεύτερο πυλώνα και τη ενίσχυση των δεύτερων πυλών τη ΚΑΠ. Χρειαζόμαστε περισσότερα, η Ρουμανία χρειάζεται περισσότερα κονδύλια για την κατάλληλη μετατροπή και των εξωτρίτων. Κατάσταση στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Έχουμε αιστείε μεμονωμένε με αγριόχειρου. Για να δούμε πώ θα πάει η κατάσταση εκεί. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να μα ανησυχεί περισσότερο πέραν του πώ εξελίσσεται η κατάσταση στη Ρουμανία. Πρέπει γι' αυτό είπα με έκτακτα κονδύλια το πρόβλημα είναι γενικό. Χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική. Δεν μπορούμε να λέμε και να ε, κοινοποιούμε ότι είναι δύσκολη η εκρίζωση. Φυσικά και είναι δύσκολη γιατί είναι ένα ιό. Είναι δύσκολο, το ξέρουμε. Αλλά μπορούμε να το πετύχουμε. Στην Ισπανία το καταφέραμε. Και η Πολωνία αντιμετωπίζει με επιτυχία ε, το πρόβλημα. Επομένω, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αυτή η στρατηγική που σα είπα. Γιατί η παραγωγή και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν ε, κάνει πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου στον τομέα του χείρου κρέατος. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και το να υπάρξει αυτή η εξάπλωση και η, ε, το πρόβλημα από τον, την αφρικανική παλόν των, των των χείρων, αυτό θα δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες για όλη την Ευρώπη. Μας ανησυχεί στην Ισπανία, όχι όμως μόνο γιατί ε, όλη η Ευρώπη πλήττεται. Τι θα γίνει τώρα με τους πληγέντες παραγωγούς από τις χώρες της Βαλτικής, από την Πολωνία, που δεν ξέρω τι θα κάνουν, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Δεν την προκάλεσαν η παραγωγή, η κτηνοτρόφια αυτή την κατάσταση. Το είπατε κι εσείς, μιλήσατε για τους ε, τουρίστες, για τους μεταφορείς, ε, όλους αυτούς τους ταξιδιώτες τέλο πάντων. Όλοι, όλοι έχουν ε, πάλι το λιθάρακι τους και αυτό πρέπει να το πούμε. Και ολοκληρώνω λέγοντας και ρωτώντα εσά, παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, πείτε μου, με ποια κονδύλια δεν μιλάω μόνο για την κοινωνική πολιτική, γιατί κονδύλια δεν υπάρχουν αρκετά ε, για την αγροτική ανάπτυξη, για τη Ρουμανία. Δεν τις φτάνουν. Χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια η Ρουμανία. Λέω λοιπόν με ποια κονδύλια. Αν υπάρχει κτηνιατρικό ταμείο. Αν έχουμε πολιτές μεσομικό πλαίσιο. Μείωση στο πολιετές, μία αύξηση στο κτηνιατρικό Πώ θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εμεί ζητούμε περισσότερα κονδύλια για την υγεία των ζών και δεν θέλουμε ούτε πάγωμα ούτε περικοπέ, όπω γίνεται στο τελευταίο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίση, πέραν των ταμείων και κονδυλίων, στο δεύτερο ερώτημα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερασπιστεί το σύστημα περιφερειοποίησης. Έχουμε ευκαιρία να μην ε, μειώσουμε τις ε, εξαγωγές μας. Παναλαμβάνω, η πιο δύσκολη κατάσταση η αυτή τη στιγμή είναι στη Ρουμανία, πρέπει να τη μετωπίσουμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκοσιεύσκα, ένα λεπτό για την ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Η Πολωνία παρατηρεί από κοντά την εφαρμογή των κανόνων. Δυστυχώ όμω η αφρικανική πανόλη των χείρων στη χώρα μα εξανατολών. Έχουμε προβλήματα εξαγωγών, έχουμε πρόβλημα με την τιμολόγηση και τώρα πριν τα Χριστούγεννα πολλοί κτηνοτρόφοι του τομέα του χειρίου κρέατος βρέθηκαν σε μια παράδεκτη κατάσταση. Ο ιός προχωρεί δυτικά όπου έχουμε τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, το μεγαλύτερο αριθμό εκμεταλλεύσεων, αν προχωρήσει δυτικά θα είναι αφάνταστες οι απώλειες. Θέλουμε να επενδύσουμε στον τομέα της κτηνοτροφίας του χειρίου, να μην περικόψουμε την παραγωγή. Και εσείς θέλετε να μειώσουμε τον αριθμό των μικρών εκμεταλλεύσεων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια τι είδους οικονομική βοήθεια προτείνετε να δώσετε. Κυρίως τώρα όπου οι τιμές έχουν καταρρεύσει και είναι ανεξάρτητα των τιμών από τους παραγωγούς και νομίζω ότι θα πρέπει να αποζημιωθούν. Ο κύριος Ράντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην Κροατία έχουμε προβλήματα με τους αγριόχειρους πέρα από την πανόλη των χείρων όπου υπάρχει ε, ανάμιξη των αγριόχειρων με τους χείρους και κάνουν ζημιές και έχουν πάει και σε περιορισμένες περιοχές και σε νησιά και δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Υπάρχει και ο κίνδυνος της αφρικανικής πανόλης των χείρων που διαδίδεται αυτή η απειλή και έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, κυρίως στα νησιά. Ε, υποστηρίζω όλες τις προτάσεις που ανέφεραν οι συνάδελφοι και που ανέφερε και ο Επίτροπος σχετικά με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους ε, κτηνοτρόφους. Θα ήθελα επίσης να θέσω ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα της ε, μη ισορροπημένης απαγόρευσης των εξαγωγών μέτρα που έχουν θεσπίσει κάποιες τρίτες χώρες. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, χώρες τις οποίες έχει ε, έχουν διαπιστωθεί κρούσματα της αφρικανικής αυτής πανόλης των χείρων και που υπάρχει κινητικότητα των αγριοχείρων. υπάρχει ο κίνδυνο να διοδοθεί ασθένεια και σε γειτονικέ χώρε. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε καλύτερα αυτού που έρχονται σε επαφή με του αγριόχειρου, κυρίω του κυνηγού, και πρέπει να ενημερώσουμε και εκείνους με, τον ένα τον άλλο τρόπο έρχονται σε επαφή με τους αγριόχειρους. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τον σεβασμό των διάφορων κανόνων υγιεινής, κυρίως αυτών που έρχονται σε επαφή με τα αγριογούρουνα. Ε, είναι σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να εκκριζωθεί η ασθένεια στις χώρες που ε, υπάρχει. Ευχαριστώ την Επιτροπή Γεωργίας και τον κύριο Σικέσκι για την ε, πρωτοβουλία. Για 1,5 λεπτό η κυρία Μιράντα έχει το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η αφρικανική πανόλη των χείρων αποτελεί μεγάλη απειλή στην κτηνοτροφία χείρων ε, λόγω των αυστηρών απαγορεύσεων εισαγωγών από τρίτες χώρες για το χείριο κρέας ε, και προϊόντα χείριου κρέατος από χώρες όπου έχει εντοπιστεί ο ιός. Ανησυχούμε πολύ για το πώς η Κομισιόν θα εξασφαλίσει ε, συντονισμό ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές στους τομείς ε, της ανθρώπινης υγείας ε, να δούμε πώς θα ελέγξει επίσης τις μεταφορές. Είπαμε, ε, ε, εσείς θα δώσετε οικονομική βοήθεια στους γεωργούς, στους εκτινοτρόφους, που είναι στη η πρώτη γραμμή του προβλήματος, αλλά πώς μπορεί η Κομισιόν να αναλάβει άμεσα μέτρα ώστε να σταματήσει την εξάπλωση της νόσου. Επίσης ανησυχούμε για το πώς η Κομισιόν χειρίζεται δυσανάλογες απαγορεύσεις ε, που υιοθέτησαν κάποιες τρίτες χώρες για τις εξαγωγές χείριου κρέατος από τα δέκα κρατη που έχουν πληγεί. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ερντός. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη Επίτροπε, η Αφρικανική Πανόλη των Χειρών ε, είναι μια σημαντική πρόκληση για όλη την Ευρώπη. Ήδη σε 10 κράτη-μέλη παντούν κρούσματα. Για την Ουγγαρία καταφέραμε να το περιορίσουμε ε, και στα 20 τα ζώα. Ε, αυτό το καταφέραμε και καλό είναι να υπάρξουν κονδύλια για ε, να δοθούν από τις αρμόδιες αρχές ε, στα κράτη-μέλη για την αποζημίωση των ε, κτηνοτρόφων. Με τον συνάδελφο Ζόγκορ και Ζόλς καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα 15 εκατομμύρια ευρώ για το πρόβλημα, του προβλήματος και παρακαλούμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ή δυνατόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τρίτες χώρες όπως Κίνα, Ταϊβάν ε, ή Χονγκ Κόνγκ να πιστούν ε, να άρουν ε, τις απαγορεύσεις εξαγωγών κρέατος από τις πληγέντες χώρες. Πρέπει να πείσουμε λοιπόν αυτές τις τρίτες χώρες ότι υπάρχει αυτή η θρησαρχή της περιφερειοποίησης, πρέπει να αναγνωρίσουν, άρα η θρησαρχη της περιφεροποιησης πρεπει να αναγνωρισουν αρα η απαγορευση δεν θα πρέπει να αφορά ένα ολόκληρο κρατός μέλλον. Όμως μόνο αυτή τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό τη Αφρικανική Πανδημία των Χείρων και θα παρακαλέσω τι δύο αυτέ προτάσει ε, να τι ε, λάβει υπόψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρο για δύο λεπτά, κ. Φαλκάρθελ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, η Αφρικανική Πανόλη είναι σοβαρή απειλή για το τομέα του χειρού κρέατος και για τα ε, γουρούνια και για τους αγριόχειρους. Ε, σημαντικές οι απώλες για την ε, κτηνοτροφία μας και πλήττονται 10 κράτη-μέλη η προετοιμασία. Σε μια, μάλλον η διάδοση σε μια αγορά χωρίς σύνορα είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ, περισσότερες, σε πολύ περισσότερα κρούσματα και θα πρέπει να συγκρατηθεί εξάπλωση του με τα απαραίτητα μέτρα. Η χώρα μου Ισπανία είναι επικεφαλής της παραγωγής χείριου κρέατος. Επτά δις είναι η αξία του τομέα αυτού. Άρα θα ήταν καταστροφικό να έχουμε πρόβλημα στη χώρα μου. Και γι' αυτό πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να προστατεύσετε τις εξαγωγές υγιών ε, σφαγίων ζώων. Και θα πρέπει να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκριζώσουμε αυτή την νόση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συντονίζεται επίση ε, και να συντονιστεί με τι ε, υπόλοιπε αρχέ, ώστε οι κτηνοτρόφοι να λάβουν τι απαιτούμενε πληροφορίε. Και αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, αυτοί πρέπει να μπορούν να πάρουν τα μέτρα. Φυσικά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα. Τα ακούμε από την Ισπανία. Αν όλα πάνε καλά, για τη Μούρθια, για τη δική μου περιοχή, θα μπορούσε ε, αυτό που έχει προτείνει ο δόκτωρ Φθκαϊνό να είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκρίζωση και ελπίζω να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, uh, Ευχαριστώ συνάδελφε. Φτάσαμε στη διαδικασία προσέγγισης προσοχής του Πρόεδρου. Ο κ. Χέτμαν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, καθόμαστε στην ωραία ζεστή μας αίθουσα, αλλά η κατάσταση χιλιάδων, πολλών χιλιάδων γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπου παράγουν χείριο κρέας είναι πολύ λιγότερο καλή και αισιόδοξη. Η παραγωγή εκεί έχει περικοπεί ή έχει εξαφανιστεί. Η κυρία Γκαρσία έλεγε ότι η Πολωνία τα πήγαινε πολύ καλά. Εν τη αυτή περίπτωση οι κτηνίατροι πρέπει να πω ότι έχουν βγει στους δρόμους, έχουν μπλοκάρει τους δρόμους διότι είναι οργισμένοι λόγω της αφρικανικής πανόλης των χειρών. Χιλιάδες οικογένειες έχουν χάσει τον, ε, τους πόρους τους, την οικονομική τους ε, διαβίωση. Ο κ. Σικέρης Προκερού είχε ετοιμάσει μια διάσκεψη σχετικά με την αφρικανική πανόλη των χείρων και μας έλεγαν οι Γεωργοί ότι χάνουν τη μάχη. Αυτή δεν είναι μια μάχη με τον ιό που χάνουν. Χάνουν τη μάχη κατά της ε, γραφειοκρατίας. Υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης. Υπάρχει ένας αδιάφορος τρόπος με τον οποίο οι αρχές αντιμετωπίζουν το θέμα και όλα αυτά οδηγούν σε μια πολύ ταχεία διάδοση της ασθενείας στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, κάποιοι που έπρεπε να σταματήσουν την παραγωγή, κάποιοι κτηνοτρόφοι σταμάτησαν την παραγωγή και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για αυτού. Υπάρχουν όμω και άλλοι που θέλουν να εξακολουθούν να παράγουν. Πάντω λάβουμε υπόψη. Είναι Χριστούγεννα. Α δείξουμε λοιπόν και κάποια καλύτερη κατανόηση. Κύριε Τέσσερι, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Ανδρουκάητης που είναι εδώ σήμερα. Η Επιτροπή Γεωργία έθεσε αυτή την προφορική ερώτηση γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα προβλήματα. Το είπαν πολύ ξεκάθαρα και το περιέγραψαν το πρόβλημα οι προλαλήσαντε συνάδελφοι. Αλλά με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων ε, δημιουργούνται πολύ σημαντικά προβλήματα και ήδη ε, το 2007 είχαμε ανάγκη, ε, μάλλον από το 2007 μέχρι το 2017 έχουν αυξήσει σε 590.000 ε, ε, τα κρούσματα. Θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Είναι λίγο ο χρόνο, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που ενδιαφέρεται για τη Γεωργία και θέλω να ευχαριστήσω, μάλλον θέλω να ευχηθώ σε όλου καλά Χριστούγεννα και φυσικά τον νέο έτο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Ντέ. Τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριο Γιάκοφτσίτση. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πιστεύω πως θα πρέπει να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, και ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ομάδα για να καταπολεμήσει την βρικανική Πανόλη των Χείρων. Θα πρέπει να υπάρξουν βεβαίως εθνικές ομάδες και περιφερειακές ομάδες αλλά και τοπικές ομάδες διότι τα οριοχηγούρουνα στην Γερμανία δεν θα τα χειριστεί το κεντρικό κράτος, αυτό θα πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα λύσετε εσείς κύριε Επίτροπε το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει αυτό να λυθεί επιτόπου, στα δάση. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια κάθετη δράση που θα φτάσει από τις Βρυξέλλες μέχρι τους Δήμους. Και επίσης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε οι γειτονικέ χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, χώρες ας πούμε των Βαλκανίων, η Ουκρανία, να κάνουν και εκείνες προσπάθειες για να λυθεί το θέμα. Σφαιρικά Επίτροπε, έχετε το λόγο για τις ε, τελικές σας παρατηρήσεις που θα είναι και οι τελευταίες παρατηρήσεις Επιτρόπου για φέτος. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι του Κοινοβουλίου. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα μας είπατε στη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Να ξεκινήσω με τα σχόλια του κυρίου Ντούντα ε, για την κατάσταση στο Ρουμανία. Ξαρχίσαμε να δουλεύουμε με την Ρουμανία από το 2015 όταν δεν υπήρχε ούτε ένα περιστατικό στην, ε, στην Ρουμανία. Αρχίσαμε να χρηματοδοτούμε εργαστήρια, δημιουργήσαμε ε, και εκπαιδεύσαμε υπαλλήλου ε, στη Ρουμανία και τους καλέσαμε σε κάθε συνάντηση ε, διδασκαλίας κατάρτισης. Όταν το 2018 εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα, όχι στο Δουναβί, στις υπόλοιπες περιφέρειες, αμέσως ζητήσαμε από τις τοπικές περιφερειακές αρχές της Ρουμανίας τους φορείς και έστειλα και τη δική μου ομάδα επιτόπου και προσπαθήσαμε να σταματήσουμε αλλά στη Ρουμανία. Παρακαλώ προσέξτε πάρα πολύ γιατί αυτή η αρρώστια, αυτή η νόσος μπορεί να έρχεται από την Ουκρανία στο Δούναβι. Γιατί ο Δούναβης είναι πάρα πολύ δύσκολος από κλιματικής άποψης. Γιατί είναι Natura 2000 και εκεί δεν μπορείς να χειριστείς με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν προβλήματα για την ε, καύση των ε, των σφαγίων λόγω ε, της κλιματικής ε, ε, ιδιαιτερότητας στη Ρουμανία. Όμως έχουμε προβλήματα με τη εκμεταλλεύσεις γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι δεν έχουν καν καταγράψει τα, ε, τα ουρούνια που έχουν στις πίσω αυλές τους. Είναι αυτή η παράδοση, είναι μεγάλη παράδοση και χρειάστηκε να στείλουμε τους καλύτερους μας εμπειρογνώμονες για να μπορέσουμε να κρυζώσουμε το πρόβλημα και να το σταματήσουμε. Και φυσικά και εισάγαμε πολύ αυστηρά μέτρα. Είναι αλήθεια στην περίπτωση της Ρουμανίας πάρα πολύ αυστηρά μέτρα για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και δώσαμε πολλά χρήματα στη Ρουμανία από το 2015. Εσείς αναφέρατε το ζήτημα για τα σφάγια και τις ε, μηχανές. Βοηθήσαμε τη Ρουμανία να εξοπλιστεί και να μπορέσει να εξαλείψει το πρόβλημα και η Ρουμανία έδρασε πάρα πολύ γενναία. Έφερε ακόμα και το στρατό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με πολλά χρήματα. Όμως είναι άλλο πράγμα τα δικά μας μέτρα και άλλο είναι τα η κοινή γεωργική πολιτική και η συνδυασμό με τον Επίτροπο Χόγκανο που επίσης πρέπει να μπορέσει να χειριστεί τα δημοσιονομικά μέσα και είναι μια καθημερινή πολύ δύσκολη δουλειά. Επόμενη συνεδρίαση έχουμε στις 19 Δεκεμβρίου και έχουμε καλέσει υπουργού Περιβάλλοντος, υπουργού Γεωργίας, πάλι όλους μαζί για να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Η απάντησή μου στην κυρία Γκαρσία τώρα. Η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Εκατοντάδες σελίδες έχουμε στη διάθεσή μας. Μιλάμε για αβεβαιότητες. Δεν μπορώ να σας δώσω απόλυτα όλες τις πληροφορίες το τι κάναμε και τι κάνουμε κάθε μήνα, διότι να θεωρούμε τη στρατηγική μας για την Αφρικανική Πανόλη των χειρών κάθε εξάμεινο. Ζητάμε από την ΕΦΣΑ να παρακολουθεί την κατάσταση και να μας δίνει πιστοποιητικά κάθε φορά ε, και τι μπορούμε να κάνουμε, ποια νέα στοιχεία έχουμε, πώς μπορούμε να δράσουμε διαφορετικά πώς μπορούμε να αναμίξουμε τον πληθυσμό, πώς μπορούμε να έχουμε κοινέ μεθοδολογίες για να υπολογίζουμε πάνω κάτω την πυκνότητα των αγριογούρνων και να μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα αφαιρέσουμε τα, τα, τα γουρούνια ώστε να συνεργαστούμε με τα κρατημέλη για να μειώσουμε τις πυκνότητες των πληθυσμών αγριογούρνων, να έρθουμε σε μια ισορροπία. Είπατε για περισσότερα λεφτά. Ε, 95 εκατομμύρια έχουμε δώσει για την ολοκλήρωση των μέτρων, χρηματοδότηση όλων των συγκεκριμένων μέτρων που περιλαμβάνονταν στη στρατηγική για την καταπολέμηση της πανόλης των χείρων. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα είναι η μεταφορά Ουγγαρία, Τσεχία και Βέλγιο ε, που επλήγησαν λόγω των ε, φορτηγών μεγάλων αποστάσεων και αμέσως προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις ζώνες. Στην Τσεχία είχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα, στην Αρλόν στο Βέλγιο επίσης ε, έχουμε ζώνη κρίζωσης και στην Ουγγαρία είχαμε δύο μόνο κρούσματα, όχι και πολύ μακριά, που επίσης απομονώθηκαν. Αλλά κανείς δεν μπορεί να δώσει εγγυήσει πως δεν θα ξαναδιαδοθεί, γιατί η περιοχή του Σέγγι δεν έχει σύνορα. Λίγο διαφορετική η κατάσταση ήταν στην Ισπανία που δεν είχαμε την ίδια δυνατότητα ε, ε, όπως το χώρο Σέγγεν και οι Υπουργοί Μεταφορών ε, δίνουν σημασία στο θέμα γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει μεγάλο ρόλο και είναι πολύ επικίνδυνο σε αυτό το τομέα. Έχω πάει στο Μόσχα, στο Κίσινοφ, στο Μίνσκ, συζητήσαμε αυτά τα θέματα εκεί με τρίτες χώρες. Η πρότασή μας ήταν απλή. Ας οργανώσουμε μια κοινή στρατηγική γιατί είναι πλέον μια πανδημία. Ξέρετε τώρα ότι η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων έχει φτάσει στην Κίνα. Και αν συγκρίνουμε την επέκταση την εξάπλωση της νόσου από το 2014 όταν εμείς αναλάβαμε θητεία όπου είχε εξαπλωθεί μόνο στη Ρωσία και στην Ευρώπη τώρα έχει πάει στην Κίνα και πάνω κάτω το διατηρούμε τα, τα προστατεύουμε τα ανατολικά μας σύνορα την Ρουμανία δηλαδή και τη, μια μικρή περιοχή της Βουλγαρίας αλλά μιλήσατε για επιστημονικά μέτρα. Δώσαμε χρήματα για να ανακαλύψουμε νέα εμβόλια. 29 εκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει για αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω πώς είναι η σημερινή κατάσταση, για την ώρα πάντως δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα για, για εμβολίωση στο μέλλον. Α, ναι, και επίσης μιλάμε όλοι για περισσότερα λεφτά. ξέρετε πολύ καλά, PDP είναι στα χέρια μας, τώρα είναι στα χέρια σας και στα χέρια του Συμβουλίου. Εμείς προτείνουμε μέσα, προτείνουμε την αύξηση των χρημάτων που αφιερώνονται στην πρόληψη και στην ετοιμασία, προετοιμασία αλλά νομίζω πως είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε περισσότερα. Και όπως ξέρετε βεβαίως, να σας πω για το εμπόριο. Στο εμπόριο έχουμε την Επίτροπο Μάλστον, Έχουμε σκληρή σχέση με την Κίνα. Έχουμε επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς ενάντια στη Ρωσία, αλλά από πολιτικής άποψης, ξέρετε, είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε Πάντως μπορούμε να μιλήσουμε για την άρση των εμποδίων και φραγμών. Ε, εμείς στηρίζουμε ε, και υπερασπιζόμαστε αυτό το θέμα και στον ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι πολύ. Βεβαίως η υποχρέωσή μου είναι να σας ε, δώσω στην Επιτροπή Γεωργίας πλήρη ενημέρωση για, αυτό, για το τι έχει γίνει επί των ε, στοιχείων και θα δώσω όλες τις πληροφορίες γιατί δίνουμε τις πληροφορίες αυτές κάθε μήνα και στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και είμαι έτοιμος να σας δώσω τις ίδιες πληροφορίες για κάθε προσπάθεια που κάνουμε ώστε να μην υπάρχει καμία βεβαιότητα για αυτό το θέμα. Είναι δύσκολη καιρή και πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περατούτε συζήτηση. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως θα υποβληθούν προς Κοινοβούλιο προς έγκριση αρχές της επόμενης συνεδρίας, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα προωθήσω αμέσως τα υφετηθέντα ψηφίσματα τη σημερινής συνεδρίασης στους αρμόδιους φορείς και πρόσωπα που αναφέρονται σε ψηφίσματα. Πριν κηρύξω τη διακοπή της συνεδρίας, για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες που συμμετείχαν για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών της Ολομελίας. Αυτό βέβαια σημαίνει τη γραμματεία της Ολομελίας, ε, ε, τους διερμηνείς, ε, τους κλητήρες, όλους αυτούς που συμμετείχαν για την έξοχη δουλειά. Εξαρτώμεθα από εσά. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και διερμηνείς σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Και για αυτούς που απομένουν τους συναδέλφους, τους τελευταίους πολεμιστές τα ίδια, καλευχές και καλή επιστροφή στις χώρες σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε και τώρα ήρθε η ώρα να κηρύξω ε, τη διακοπή της συνεδρίας. Ε, Πέρας αυτής. Γεια σας.